All uh, ladies and gentlemen. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, κυρίσω την έναρξη της Συνόδου Λομέλειας, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Συνόδου Λομέλειας, της 8 η και 9 η Φεβρουαρίου. Θα ήθελα την έγκρισή σας. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Και τώρα μια σύντομη δήλωση ως πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών να ανακεφαλαιώσω κάποια από τα περιστατικά και τα συμβάντα της περσινής χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπη, κυρίες και κύριοι, φίλε και συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς οι Βρυξέλλες, η χώρα που μας φιλοξενεί, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσής μας, υπήρξε στόχος επιθέσεων που προκάλεσαν ε, την θλίψη και τον αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη. Σήμερα, ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις αυτές, εκφράζουμε την ε, αλληλεγγύη μας προς τον λαό των Βρυξελών και τα αθώα θύματα και όσους έχασαν ε, ανθρώπους από την οικογένειά τους, τους αγαπημένους τους. Αυτούς των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα και που πολλές φορές ο πόνος τους διαρκεί ακόμα. Δεν ξεχνάμε, ούτε θα ξεχάσουμε ποτέ, τι συνέβη πριν από ένα, χρόνο. Δεν θα το ξεχάσουμε, διότι υπήρξαν και συνεργάτες από, τη δική μου, την, από το δικό μου το γραφείο που τερματίστηκαν. Τα γεγονότα αυτά δεν θα μας καθορίσουν. Μπορεί να μας επηρέασαν βαθιά, αλλά δεν θα μας εξαναγκάσουν να αντιδράσουμε όπως κάποιοι ήθελαν. Θα διατηρήσουμε ανέπαφες τις αξίες που ως Ευρωπαίοι πρεσβεύουμε. Αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας, που θα είναι πάντοτε η πηξίδα μας. Πριν από ένα χρόνο είπα ότι η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει θα ζήσουμε, θα αγαπήσουμε και θα εργαστούμε. Πιστεύω ότι παρόλα όσα έγιναν αυτό κάναμε. Δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα παραδώσουμε τα όπλα ούτε και στις πιο πιεστικές ε, καταστάσεις. Ε, πριν από ένα χρόνο δεν το κάναμε, δεν το κάνουμε σήμερα ούτε αύριο. Εδώ ο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει. Επιβεβαιώνουμε σήμερα ότι κακώ μα επιτέθηκαν πριν ένα χρόνο και υψώνουμε τον άστημά μα παρά τι εθνικέ διαφορέ, τι πολιτιστικέ μα ανομοιότητες. Αυτά δεν μα χωρίζουν. Θα παραμείνουμε ενωμένοι κατά του μίσου και του τρόμου. Α δείξουμε σε όσους θέλησαν να μα πλήξουν ότι η καρδιά τη Ευρώπη χτυπάει κανονικά. Ας έχουμε ένα λεπτό σιγής. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, δήλωση του Επιτρόπου Ανδρέου Κάιτη, Επιτρόπου Υγείας και Ασφαλείας Τροφίμων. Να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το θέμα όπως το εξέτασε η Επιτροπή μας, η Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίζουμε στη Σύνοδο Λομέλειάς μας για να συζητήσουμε την πολιτική για τα τρόφιμα στα πλαίσια του περιβάλλοντος και της βιώσιμης στήριξης και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. Ως το 2030 οι ανάγκες του κόσμου θα έχουν αυξηθεί κατά 50% κατά 30% σε νερό και κατά 45% σε ενέργεια. Ο τομέας των τροφίμων είναι το 25% της πηγής παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και ευθύνεται για το 60% της απώλειας βιοπικιλότητας παγκοσμίω. 9 από τα 17 μέτρα ε, μεταξύ των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό δείχνει τι ανάγκη για δράση υπάρχει από πλευρά μα και πόσο πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τα συστήματα παραγωγή μα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην Ευρώπη ώστε η παραγωγή τροφίμων να γίνει πιο βιώσιμη. Πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες, τι διατροφικές, καθώς και τον τρόπο που ε, επεξεργαζόμαστε τα απόβλητα με μια υπεύθυνη απάντηση για την επιστηστική ασφάλεια και τι ανάγκε τη αγορά. Θα πρέπει να, να προστατεύουμε τα τοπικά οικοσυστήματα, την γεωργία και του παραγωγού για το μέλλον. Θα πρέπει να μειώσουμε, την, να περιορίσουμε την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και το μοντέλο κατανάλωσης, έτσι ώστε να σεβόμαστε το περιβάλλον και να σεβόμαστε τη βιώσιμη παραγωγή. Πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση από τα σχολεία. Ένα στα τρία εντεκάχρονα της Ευρώπης είναι ήδη παχύσαρκο. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στη βιώσιμη διατροφή και αυτό να ξεκινήσει με την παιδεία, στα σχολεία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να αγοράζουν τρόφιμα ε, που παράγονται τοπικά για να έχουμε ένα, ε, μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή και να στηρίξουμε τι τοπικέ οικονομίε. Θα πρέπει οι προκλήσει αυτέ να χρησιμοποιηθούν ω ευκαιρίε για να αναπτύξουμε νέα επιχειρησιακά μοντέλα με την κοινοτομία. Η παραγωγή μπορεί να διατηρήσει τι περιοχέ τη υπαίθρου σε καλή κατάσταση και με θέσει εργασία 47 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σε 50 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς η πηγή τη διατροφής, είναι και μέρος της ταυτότητάς μας. Όπως έγραψε ένας Γάλλος πολιτικός της αρχής του 19ου αιώνα, πείτε μου τι τρώτε για να σας πω ποιο είστε. Η σημασία των ε, γαστρονομικών προτιμήσεων στις διάφορες ε, περιοχές μας δεν μπορεί να παραμεληθεί. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά βλέπω ότι η γνωμοδότησή μας καλύπτει και αυτό το σκέλος. Η Επιτροπή μας ζητά να υπάρξει μια σφαιρική, βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ασχολείται με την παραγωγή των τροφίμων και την διατροφή με έναν τρόπο πιο ευρύ, ώστε να διασυνδέονται όλες οι διαφορετικέ πολιτικές μεταξύ τους όπως η παραγωγή τροφίμων, η γεωργία, το περιβάλλον, η υγεία, η πολιτική για τους καταναλωτέ, η απασχόληση και η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, να δώσω τον λόγο στον φίλο μα και τακτικό προσκεκλημένο μα, τον κύριο Ανδριού Κάιτη, για να μα ε, παρουσιάσει τι απόψει του. Thank uh, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή των Περιφερειών, εξαιρετικά μέλη τη Επιτροπή των ε, Περιφερειών και αν με επιτρέπετε αγαπητοί φίλοι. Είμαι ιδιαίτερο ευτυχή που έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Σύνοδο σα και θα ήθελα να σα συγχαρώ για το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο προβλέπετε να υιοθετήσετε σήμερα για την ε, αηφόρο πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα. Εμεί είμαστε πρωτοπόροι στην, ε, στην υλοποίηση, στην πράξη αυτών των αλλαγών, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στους πολίτες να επιλέγουν μια υγιεινή διατροφή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση φτηνή σε τιμές κοινωνικά αποδεκτές σε αυτήν την υγιεινή διατροφή. Γιατί οι πολίτες μας πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με την ακριβώς αντίθετη κατάσταση. Σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες γειτονιές υπάρχουν πάρα πολλές αλυσίδες fast food και είναι πολύ πιο εύκολο να, να, να, να επιλέξει κανείς αυτή τη διατροφή παρά υγιεινή διατροφή με φρούτα και λαχαντικά. Η αηφορία, όταν συζητούμε για την αηφορία, η... σχετίζεται όχι μόνο με τους ποδηλατόδρομους ή με τις μεταφορές, αλλά επίσης και με την πολεοδομία, επίσης και με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγιεινή διατροφή. Έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια πιο υγιεινή, μια υγιή συγγνώμη, κοινωνία. Βέβαια οι πολίτες ζουν σε κέντρα παραγωγής, δεν είναι απλώς καταναλωτές. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι στα αστικά κέντρα δεν υπάρχουν αρκετές δυνατότητες ε, επιλογής για τους καταναλωτές τοπικών προϊόντων. Οι πλέον σημαντικές πολιτικές που ακολουθούμε είναι εκείνες οι οποίες ε, συμφωνούνται και αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο. σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην πολιτική, την κοινωνική ή στις δημόσιες ε, προμήθειες. Σε όλους αυτούς τους τομείς, οι επεμβάσεις, παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στην, στην αλυσίδα, μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, να είμαστε περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον. Με πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία, οι καντίνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των τοπικών οικονομιών. Οι πολίτες της Ένωσης, οι περιφερειακές αρχές, έχουν ε, σημαντικό ρόλο να παίξουν για να προωθήσουν μια υγιεινή διατροφή, ιδιαίτερα στις πλέον περιοθεοποιημένες ή ευάλωτες ομάδες, που συχνά είναι εκείνες που πλήττονται δυσανάλογα. Η προστασία του περιβάλλοντος, ένα υγιές ε, υγιείς ε, συνήθειες είναι μια κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών μας για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Δεν ζητούν απλώς πιο υγιεινή διατροφή, αλλά επίσης και τρόφιμα τα οποία να παράγονται με τρόπο ε, βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντω, γιατί σχετίζεται με την αηφορία της παραγωγής τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχώρησε σε ανακοίνωση για την, ε, πολιτική, την αηφόρο πολιτική για τα τρόφιμα στο πλαίσιο της, ε, του θεματολογίου για την αηφορία προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων δημιουργώντας τελικά ένα, μια πλήρη ατζέντα για τα τρόφιμα. Συμβατή και με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030. Με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα ε, βοηθάμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ε, δημογραφικής αλλαγής. Τις επόμενες δεκαετίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι η φυσική πόροι είναι περιορισμένοι και εξαιτία της κλιματική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά ο πληθυσμός θα έχει αυξηθεί. Αναμένουμε να φτάσουμε τα 10 δισεκατομμύρια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικό και, θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα. Η παραγωγή τροφίμων είναι ήδη τεράστια. Όμως πρέπει να γίνεται με τρόπο πλέον πιο αηφόρο πια γιατί έχουμε δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από λοιμό, ενώ ταυτόχρονα ο ΠΟΗ εκτιμά ότι το 1 τρίτο της παραγωγής τροφίμων τελικά δεν αξιοποιείται. Είναι απαράδεκτο αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 80 εκατομμύρια μετρική τόνοι είναι τα τρόφιμα τα οποία κάθε χρόνο καταλήγουν στα σκουπίδια. Ε, με οικονομικό κόστος 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη κατάσταση. Φαντάζομαι 143 δισεκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι όλοι από εσά θα είχατε πώς να αξιοποιήσετε 143 δισεκατομμύρια επιπλέον στις περιφέρειές σας, στις πόλεις σας. Είναι τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή πετάμε. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε αυτή τη σπατάλη των τροφίμων κατά 50% είναι ο στόχος μας μέχρι το 2030. Ε, πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Ε, αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις και αντιμετωπίζοντας αυτή την απαράδεκτη σπατάλη φυσικών πόρων, θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή γιατί το 8% της παραγωγής αερίων ε, του, που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι, αποτέλεσμα αυτής της πατάλης. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τον, την, την πείνα και την κακή διατροφή πιο αποτελεσματικά. Πρέπει να αναδιοργανώσουμε την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης έτσι ώστε να μειωθεί η σπατάλη και σε όλα τα στάδια. Από την παραγωγή στον, στο μεταποιητή, στον εμπορευόμενο, στον τελικό καταναλωτή. Παντού, σε όλα τα στάδια. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, εμπορευόμαστε, ρυθμίζουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμα. Έχουμε μια παροιμία. Ε, φάει μόνο σου το πρωινό, το γεύμα το μεσημεριανό μαζί με ένα φίλο και το βράδυ, το, γεύμα, το, το βραδινό σου να το δώσεις έναν ε, εχθρό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο παραγωγής και το μοντέλο κατανάλωσης. Γι' αυτόν τον λόγο οι πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται στο κέντρο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Το πακέτο μέτρων για την κυκλική οικονομία προσπαθεί να δημιουργήσει κίνητρα για πιο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της, της αηφόρου ανάπτυξης, της αηφορίας στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η καταπολέμηση αυτής της σπατάλης των τροφίμων χρειάζεται την συνεργασία και την εμπλοκή όλων. σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας και αν δραστηριοποιούνται. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα για την σπατάλη στον τομέα των τροφίμων, για να ε, διευκολύνουμε τη συνεργασία είτε δημοσίων αρχών είτε ιδιωτικών επιχειρήσεων και να ε, κινητοποιήσουμε ε, με αυτόν τον τρόπο την λήψη ε, μέτρων. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο που σας είπα, της μείωσης κατά 50% στο 2030, έχουμε διαπιστώσει ότι τα μέλη αυτής της πλατφόρμας ε, με μεγάλο ενθουσιασμό μοιράζονται με τους συναδέλφους τους πρωτοβουλίες, ιδέες και μοντέλα με τα οποία κανείς μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά παντού την σπατάλη ε, στα τρόφιμα. Έχουμε επίσης μια πρόταση, μάλλον έχουμε επίσης την νομοθεσία η οποία ζητά από τα κράτη-μέλη να ε, μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων και να ε, λογοδοτήσουν για την πρόοδο που σημείωσαν. Η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη, θα προσπαθήσει να υποστηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες δίνοντας μια κοινή μεθοδολογία στην οποία θα καταλήξουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη δωρεά τροφίμων, διασφαλίζοντας βέβαια ότι τα τρόφιμα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές να καταλήγουν εκεί. Να μειώσουμε τις πατάλες σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα νοικοκυριά, χωρίς βέβαια να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων. Αγαπητοί, αγαπητά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε από τη δικιά μας πλευρά, την πλευρά της Επιτροπής και με χαρά θα ακούσω τις πρωτοβουλίες που εσείς αναλαμβάνετε σε περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφέρειες, οι πόλεις βρίσκονται στην καρδιά της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό οι που θα εκφράσετε εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικές, θα τις ε, ε, ακούσω με προσοχή. Ε, η πόλεις και οι περιφέρειες βρίσκονται πολύ πιο κοντά στους πολίτες και γι' αυτόν τον λόγο έχουν τεράστια σημασία να, ακούγεται, τεράστια σημασία να ακούγεται η φωνή τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας ρωτώ, εσείς στα δημοτικά σας συμβούλια, στα κοινοτικά σας συμβούλια, έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της πατάλης των τροφίμων. Αυτό είναι το ερώτημά μου προς εσάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας αρχής ε, γενομένης από τις εκπροσώπους των πολιτικών ε, ομάδων. Έχουμε διαφορετικούς χρόνους αγόρευση ανάλογα με το μέγεθος ομάδας. Ο κύριος Άρνο Κόμπατσέρ είναι ο πρώτος εξ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αντριουκάητης για την παρουσία του εδώ, που καταδεικνύει τη σημασία που έχει το θέμα αυτό συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει επίσης ότι έχει αναγνωρίσει η Κομισιόν το γεγονός ότι στον τομέα αυτό πρέπει να κινηθούμε, να αναλάβουμε δράσεις. Σας συγχαίρω λοιπόν, διότι έχετε ήδη λάβει πολύ σημαντικές αποδοτικές πρωτοβουλίες και η δική μας βέβαια Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, έχουμε ε, δημοσιοποιήσει μια σημαντική γνωμοδότηση για τη σπατάλη τροφίμων. Ο να ήταν συγητής και πραγματικά και το πακέτο για την κυκλική οικονομία είναι αξιοσημείωτη πρόταση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ηθική πλευράς πραγματικά είναι απαράδεκτο ε, να ε, υπάρχει πρόβλημα λοιμού ένα τρίτο των ανθρώπων να πεινούν και πάρα πολλά τρόφιμα να πετάγονται στα σκουπίδια στις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Εμείς όμως βλέπουμε και κάτι περαιτέρω. θέλουμε ναι σίγουρα να αποφύγουμε τη σπατάλη τροφίμων. Είχαμε και ένα μια εκδήλωση με τα μέσα ενημέρωσης ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής των ε, Περιφερειών ε, για την παρακολούθηση της κατάστασης και το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών νομίζω δίνει το καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να αποφευθεί η σπατάλη. Σίγουρα πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν και εσείς κύριε Επίτροπε έχετε δίκιο ότι από κοινού οι περιφέρειες οι τοπικοί φορείς ε, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, μπορούν να συνεισφέρουν τα μάλλα σε αυτή την προσπάθεια. Η πρωτοβουλία, η γνωμοδότηση που θα συζητηθεί στη συνέχεια ε, δεν πραγματεύεται μόνο το θέμα της πατάλης ε, τροφίμων, αλλά συνολικότερα μια βιώσιμη πολιτική τροφίμων. Εσείς τονίσατε ότι η παραγωγή, η επεξεργασία τροφίμων ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της γεωργίας. Εξαρτώνται πάρα πολλές θέσεις εργασίας από αυτό, ιδίως στην Ήπεθρο. Αυτό είναι μια πτυχή. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή όμως, ε, η οποία αφορά και την ε, διασπάθηση πόρων, για να μην πω και την επιβάρυνση ε, του περιβάλλοντος. Ε, υπάρχουν θετικά εξωτερικά αποτελέσματα, υπάρχει πράγματι αυτή η προσπάθεια για μια υγιή, για μια νέα κουλτούρα, αλλά υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις για τη χρήση και κατάχρηση και υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Το θέμα είναι πώς θα εσωτερικεύσουμε τα θετικά, εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία. Έχουμε την πολιτική υγείας, πάρα πολύ σωστά το είπατε και βέβαια την πολιτική γεωργία. Θα πρέπει επίση με την γεωργία να φροντίσουμε και με την κατάσταση να προσφέρουμε πιο υγιή τρόφιμα και σίγουρα ε, υπάρχει και το θέμα της εκπαίδευσης και πολιτική εκπαίδευση, γιατί πάρα πολλά έχουν να κάνουν ε, με την οτροπία μας, με την ε, εκπαίδευσή μας. Πρέπει λοιπόν να επιμορφώσουμε τον κόσμο πώς να καταναλώνει και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και σε ό,τι αφορά επίσης το εισόδημα των φτωχών οικογενειών, των αδύναμων οικογενειών και, και αυτοί χρειάζονται ενίσχυση, εισοδηματική ενίσχυση. Θέλω να ευχαριστήσω και για τη μεγάλη υποστήριξη που έχω βρει και συγκεκριμένα ό,τι αφορά συγκεκριμένε προσεγγίσεις. Στο μέλλον, να έχουμε δαφικές προτιμήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ για τη σχολεία, τα βραχονιπιακούς σταθμούς, τα νοσοκομεία, να μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, περιφερειακή, την τοπική ε, ε, κυκλική οικονομία. Θέλουμε επίσης να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου, έχουμε το θέμα των μεταφορών γερικών προϊόντων και άλλα. Θέλουμε προς παραγωγή φιλοπεριβαλλοντική φιλική προς τη φύση. Νομίζω ότι δεν πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε τις προσπάθειες στον τομέα αυτό. Γίνονται πάρα πολλά ήδη βέβαια, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες ό,τι αφορά τις ε, κλίμακε κλίμακες εκμεταλλεύσει ε, στην Ήπεθρο, είναι δύσκολο, αλλά και σε ορεινές περιοχές, για παράδειγμα, που έχουν πολύ διαφορετικές γεωμορφολογικές συνθήκες. Νομίζω θα πρέπει να τονίσουμε το περιφερειακό στοιχείο, την περιφερειακή διάσταση. Αυτό ε, πρέπει να στηριχθεί. Επίσης, και η ορολογία παίζει το ρόλο τη. Ε, το είπατε και εσεί, κύριε Επίτροπε, σε ό,τι αφορά τη σπατάλη τροφίμων. Καταρχά, θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση και να έχουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μα για να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει αυτό. Αλλά και σε ό,τι αφορά την παραγωγή, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι όροι. Τι θα πει βιωσιμότητα και μετά να υπάρχει απαραίτητη πληροφόρηση. Όχι πια πολύπλοκη, δύσκολη επισήμανση, ετικέτες, αλλά σαφή μηνύματα για τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα αυτά έχουν παραχθεί με βιώσιμη, βιώσιμο τρόπο και επομένως κανείς ε, με ίση συνδυσή του μπορεί να τα καταλάβει. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτά όταν θα παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου. Πρόεδρο, συγγνώμη διακόπτω. Let's Ας περάσουμε στον επόμενο μιλητή από την ομάδα των Σοσιαλτικών Δημοκρατών. Ο κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την αρχική του δήλωση. Νομίζω ότι ο τομέας της υγείας, παρόλο που είναι αρμοδιότητα εθνική, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καλό να συζητάμε και χρειάζονται πρωτοβουλίες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και πλήττονται και τα υγειονομικά του συστήματα. Είναι εκτεθειμένα στις οικονομικές αντικσότητες. Πρέπει λοιπόν όλοι να πετύχουν περισσότερα, να καλύψουν περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα. Θα συζητήσουμε αργότερα σήμερα τη σχετική έκθεση για το πού βρισκόμαστε στην παγκόσμια αγορά σε σχέση με αυτά. Άρα είναι σημαντικό να συγκρίνουμε και να ανταλλάξουμε μεταξύ μα ιδέε και απόψει. Όμω την υγεία δεν πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε μόνο υπό την στενή της έννοια. Είναι ένα τομέα ο οποίος καλύπτει και άλλα ε, θέματα και ε, άπτεται και άλλων κλάδων. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια προσέγγιση όπου το υγειονομικό σύστημα να συνδυάζεται και με άλλες παραμέτρους της κοινωνίας. Οι θέσεις απασχόλησης λόγου χάρη, υγειονομική περίθαλψη έχει σημασία για την αποθεραπεία των εργαζομένων που μετά μπορούν να γυρίσουν στη δουλειά τους ε, κανονικά, λόγου χάρη. Χρειάζονται λοιπόν ε, την υγεία οι πολίτε για να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να παραμένουν μεταγωνιστικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω και η υγεία βασίζεται σε κάποιε υποθέσει που ανέφερε και ο Επίτροπο και ο Πρόεδρο τη Επιτροπή. Ε, ο τομέα των ε, τροφίμων, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ πέρα. Πρόκειται να αναθεωρήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική και η επιθυμία μα θα ήταν να είναι μια κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική των τροφίμων. Να επικεντρώνεται στο τι τρώμε, τι πίνουμε, τι καταναλώνουμε και πώς παράγονται όλα αυτά που καταναλώνουμε. Αυτά δεν είναι άνευ νοήματος. Έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Βακτηριακές, την αντίσταση στα αντιβιωτικά, ε, την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Απλώς για να αναφέρω μερικές από τις προκλήσεις που καλό είναι να τις λάβουμε υπόψη. Εάν μπορέσουμε να αλλάξουμε έστω και λίγο τις διατροφικές μας συνήθειες και να Σεβόμαστε περισσότερο τις παραγωγικές απαιτήσει για να υπάρχει καλύτερη υγεία. Θα πετύχουμε πολλά περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, είναι σημαντικό να αναλάβει δράση και ο Επίτροπο για την Υγεία και τα Τρόφιμα να ε, δείξει την απαραίτητη ευαισθησία. Από ό,τι ακούω, από την δήλωση που μόλι μα έκανε, όντω είναι έτοιμο να το κάνει αυτό. Η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στα τρόφιμα διότι 15% των γεωργών κάνουν τις πωλήσεις τους απευθείας προς τον καταναλωτή. Όμως πρέπει να μεγαλώσει το ποσοστό αυτό. Όσο πιο σύντομη είναι η αλυσίδα παραγωγής, τόσο περισσότερο ε, μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα το τι παράγουν οι γεωργοί και τι καταναλώνουμε. Οι διαφορές στις τιμές, οι διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης, είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αν και βεβαίω οι χώρε μα διαφέρουν πάρα πολύ, έστω και μορφολογικά μεταξύ του. Πάντω, την αλυσίδα παραγωγή τροφίμων την έχει λάβει από ό,τι φαίνεται υπόψη τη Επιτροπή στο σχεδιασμό τη πολιτική τη. Ε, η ερώτησή μου είναι, ξέρετε άλλε χώρε που να έχουν κάνει κάτι ανάλογο ώστε να γίνει συντομότερη η αλυσίδα. Ε, το ελεκτικό συνεδρίο πρόσφατα δημοσίευσε έκθεση όπου τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να πετύχει μια αλυσίδα παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη των τροφίμων στο δυνατόν περισσότερο η σπατάλη των τροφίμων πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πιστεύουμε και εμεί ότι 30% λιγότερο στο 2025 είναι ένα θεμετό στόχο. Η Επιτροπή φαίνεται να τον ε, εγκρίνει το στόχο αυτό. Ένα άλλο όμω στόχο είναι να υπάρξει μια ε, βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυαζόμενη με άλλε πρωτοβουλίε. Εν είδη συμπεράσματο να πω προ τον Επίτροπο. Ελάτε στη Δανία, στη Νότια Δανία όπου έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο ό,τι αφορά τη χρήση των τεχνολογικών μέσων για την ευζοία των ζώων, για την υγεία. Να σας προσκαλέσουμε για να δείτε κάποιες νέες ιδέες στον τομέα της κοινοτομίας, της χρήσης της τεχνολογίας για αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ, Σας Ευχαριστούμε. Η κυρία, ο κύριος Μαρτικάινεν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την εξαιρετική άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία του. Θέλω να συγχαρώ επίσης τον εισηγητή της γνωμοδότησης, τον κύριο Κόμπατσερ, που είναι πάρα πολύ καλή ε, και συμπληρώνει το καλό έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή των ε, Περιφερειών σε αυτό το τομέα μέχρι σήμερα. Πολλοί ε, είπαν ορισμένα πράγματα και οι σήμερα με τους οποίους συμφωνώ θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Τα προβλήματα στον επιστημιστικό τομέα και ιδίω ε, η κρίση του κρέατος λόγω του βραζιλιανού κρέατος ε, δεν περιορίζεται ε, στο εξωτερικό, δηλαδή εισαγωγικά κρέατο, μολυσμένου κρέατο από, το, από άλλε χώρε, αλλά και μέσα στην Ένωση εντοπίζεται το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλά τρόφιμα που δεν είναι αυτό ακριβώς που υποτίθεται ότι είναι. Πώς θα τα καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά. Πώς ε, θα αποφύγουμε να έρχεται στην Ένωση παραποιημένο επίσης ε, παραποιημένα τρόφιμα ή λιγμένα ε, Οι καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη Πώς θα το πετύχουμε αυτό, πώς θα καταπολεμήσουμε τη σπατάλη των τροφίμων και τη σπάση φυσικών πόρων. Είναι πολύ προβληματική αυτή η τομή. Όλα δείχνουν ότι χρειαζόμαστε μια πάρα πολύ ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική, γιατί ε, και βέβαια και η περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική υγεία σχετίζονται. Και για να επανέλθω. Στην κοινή γεωργική πολιτική δεν νομίζω ότι θα ήταν βιώσιμο να επανακρατικοποιηθεί. Η χνελασσομάδα τροφίμων επίσης θα πρέπει να είναι σύντομη και αναγνωρίσιμη, χνηλάσιμη η τροφική αλυσίδα. Επίσης, απώλεια ενέργειας, ε, το έχουμε πει και κατά το παρελθόν μας έχει απασχολήσει. Ο είναι αυτός ο οποίος ε, θα προβεί τελικά στις επιλογές αλλά πρέπει να αλλάξουν ε, οι κανόνες της κάπω ώστε να μπορούν να κάνουν ε, σοφές επιλογές καταναλωτές. Η αλυσίδα των τροφίμων μπορεί να μας φέρει περισσότερη αξία, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων τη σπαταλή ενέργεια. Αυτό είναι προ το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο έχει επίσης συγκροτήσει ένα φόρουμ ε, που θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει τη σπατάλη των ε, τροφίμων. Θα είμαι μέλος, ε, ως, μέλος των Περιφέρειων και εμπειρογνώμονες οι πλέον κορυφαίοι στον κόσμο θα συνεργαστούν με αυτό το φόρουμ πλέον για να βρουν λύσεις και ελπίζω να βρεθούν οι λύσεις να δοθούν απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα και βέβαια και η Κομισιόν πάντοτε είναι καλοδεχούμενη στις συναντήσεις μας. Ο Μάρε Κουλτσέσκη, έχετε δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου της Άλντε, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για εμάς που ο Επίτροπος Ανδριουκάητης ε, συμμετέχει στην συζήτησή μας για τα τρόφιμα πριν 30 χρόνια, Γερμανός φιλόσοφος, αναφέρθηκε στους κινδύνους στην, σε μια κοινωνία και η κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθεί μια πυραμίδα στον, στον κόσμο ξεκινώντας από την αποφυγή των κινδύνων για το περιβάλλον που προκαλείται από την παραγωγή των τροφίμων. Η ίδια η έννοια της ασφάλειας τροφίμων είναι απόρρια ε, της, της, της, της λογικής για την παραγωγή ε, τροφίμων με ε, τρόπο βιώσιμο, με τρόπο αηφόρο. και είναι βεβαίω πάντοτε απολύτω απαραίτητο για μια κοινωνία να φροντίζει για την υγεία των μελών τη και για την ασφάλεια των τροφίμων. Η σημασία των περιφερειακών αρχών πρέπει να τονιστεί και στην πράξη. Τα προβλήματα ασφάλειας τροφίμων δημιουργούν ε, προβλήματα και στις περιφερειακές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και έχει πει και ο Επίτροπος, μπορεί να δημιουργήσει ένα μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που να είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά στον κόσμο, όμως κοστίζει πολύ. Και αυτό οδηγεί σε αύξηση των τιμών των τροφίμων. Και το αποτέλεσμα είναι στην αγορά τελικά να εισάγονται τρόφιμα ε, χειρότερης ποιότητας ε, από το εξωτερικό, τα οποία δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά τα οποία οι καταναλωτές προτιμούν γιατί είναι φτηνότερα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, γιατί δεν είμαστε μόνο εισαγωγή. Ε, δεν εισάγουμε μόνο τρόφιμα, αλλά εξάγουμε και τρόφιμα. Και δημιουργεί στρεβλώσει στον ανταγωνισμό. Εάν λοιπόν βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στον τομέα αυτό, θα έπρεπε να προσπαθούμε, θα, θα, καταφέρουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε ε, προσιτές τιμές για όλους, τιμές προσιτές για όλους. Και το ερώτημά μου προς εσάς, κύριε Επίτροπε, είναι το εξή. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που να εγγυάται αυτήν την παροχή, την, την ε, διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας τροφίμων σε το, ε, προσιτές τιμές. Ευχαριστούμε κύριο Γκόρλεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Επίτροπε. Θέλω να αδράξω την ευκαιρία για να καλωσορίσω την Επιτροπή εκ μέρους της Ομάδας των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Να ξέρετε ότι η ομάδα μας εξετάζει το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας κατά εδώ και πολύ καιρό. Διότι από την οπτική γωνία των ε, ε, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι τα τρόφιμα που παράγουμε με τη χρήση των φυσικών πόρων είναι σαν τον αέρα που αναπνέουμε. Το περιβάλλον εντός του οποίου ζούμε είναι ένας φυσικός πόρος ο οποίος πρέπει να διαφυλάσσεται. Εκ μέρους της ομάδας μας λοιπόν να σας πω ότι θα προτιμούσαμε να μην ε, καλύψουμε εδώ και τον τομέα της υγείας. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα θέματα αποτελούν θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Αλλά σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ε, ρυθμιστούν όλα τα θέματα είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα, τρόφιμα με εύληπτες ετικέτες για να μπορούν να καταλάβουν τη σύστασή τους. Τρόφιμα που να είναι ασφαλή για την υγεία τους. Υπάρχουν κάποιες αρνητικές τάσεις στην πολιτική για τα τρόφιμα θα πρέπει να φροντίσουμε η αλυσίδα από το χωράφι στο πυρούνι να μην είναι τόσο μακριά. Δεν θέλουμε οι καταναλωτές να είναι πολύ μακριά από την τοπική παραγωγή των τροφίμων. Επίσης τα χημικά πρόσθετα είναι ένα πρόβλημα. Ως εκ τούτου, καταλαβαίνετε ότι είναι αρνητικές και συνέπειες για την υγεία. Όμως δεν θέλουμε να παρέμβουμε υπερβολικά στις καθημερινές επιλογές των καταναλωτών. Αυτό δεν σημαίνει από την άλλη ότι δεν πρέπει να γίνονται περισσότερα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα τρόφιμα που αγοράζουμε είναι ασφαλή και ότι οι ετικέτες που μπορεί να διαβάσει εύκολα ο καταναλωτής το επιβεβαιώνουν. Πιστεύω ότι όλες οι εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που θα εγκρίνουμε θα πρέπει να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμη τέσσερις σύντομες συνεισφορές. Θα ακούσουμε τους δύο πρώτους για τρία λεπτά και οι υπόλοιποι για λιγότερο και οι υπόλοιποι για ένα για να προλάβουμε. Α, μόλις εγγράφηκε κι άλλος ένας. Λοιπόν, ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Σακρεντέους, την άλλη συγκήτρια. Έχετε τρία λεπτά για την μονοδότησή σας που αφορά τα συστήματα υγείας διότι θέλουμε να προλάβει να τα ακούσει και ο Επίτροπος που είναι επιτεταμένος των θεμάτων υγείας. Κυρία Σακαντέους. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Αργότερα σήμερα θα μας απασχολήσει η έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της υγείας στην Ευρώπη. Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερο κανοποιημένη και ευγνώμων για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τα διάφορα αυτά σχέδια ε, για να εξετάσουμε συνολικά την κατάσταση υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της Κομισιόν. Διαπιστώνουμε στη γνωμοδότηση που εγώ προσωπικά συνέταξα από πλευράς Επιτροπής των Περιφερειών ότι οι χρόνιες παθήσεις κοστίζουν και μάλιστα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους που επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ό,τι αφορά το κόστος τη υγειονομική περίθαλψη, έχοντα υπόψη μα και τη γύρανση του πληθυσμού. Κατά την άποψή μα λοιπόν πρέπει να γίνουν περισσότερα και στον τομέα τη πρόληψη. Και βέβαια εδώ, στον τομέα της πρόληψης, δηλαδή, εντάσσεται και το τομέας των τροφίμων. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ασχοληθεί με το κάπνισμα, όχι όμως με την παχυσαρκία. Γινόμαστε όλο και πιο παχείς και ιδίως τα παιδιά μας. Οι πολιτικοί λοιπόν πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερο στον τομέα της πρόληψης Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να σχολιάσει μέσω του κ. Αντρουκάητη. σήμερα να μας πει τι μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δυνατήσει ο κόσμος. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι στον τομέα των τροφίμων θα πρέπει να θεσπίσουμε μια επισήμαση, μια ετικέτα η οποία θα αναφέρει την ε, σύνθεση, τα συστατικά, δηλαδή κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή αλλά και το οικολογικό ίχνος, το οικολογικό αποτύπωμα. Δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό θα ήθελα να περιοριστώ σε κάποια παραδείγματα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι πολυεθνικοί όμιλοι ε, σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να προσφέρουν όλο και χειρότερη ποιότητα ε, τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πιο συχνά, όλο και πιο συχνά. Τα προϊόντα που παράγονται από ε, πολυεθνικές δεν είναι πια δυστυχώς καλής ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε, και είναι μια αντικειμενική διαπιστώση αυτή, ότι τελικά χρησιμοποιούν το μέγεθός τους οι μεγάλοι όμιλοι για να δυσχεράνουν τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε την εγχώρια γεωργία, να την υποστήριξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ε, ομιλήτρια είναι η κυρία Κάρσον. Okay, uh, that's canceled then, uh, Mr. Ο κύριος Βραμμοβίτσιος, αφού η κυρία Κάρσον τελικά δεν ζήτησε το λόγο, θα μιλήσω λιθουανικά. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη Σύνοδο Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών και για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των τίτλων της Επιτροπής στον τομέα αυτών που μας κάνατε. Ε, από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θεωρούν εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεται σε αυτόν τον τομέα. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να βοηθήσουμε την Επιτροπή να υλοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες. Γιατί τελικά η καταναλώση τροφίμων, οι συνήθειες, οι καθημερινές ε, στη ζωή των ανθρώπων είναι κάτι πολύ σημαντικό για, για όλους μας. Σας εύχομαι πάντως καλή επιτυχία στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε παρουσία του Επιτρόπου που νομίζω για την υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δείχνει πόσο, σημαντική είναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θεματολόγιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ήταν πολύ ε, συναρπαστική η παρουσία σας. Έδειξε μεγάλη προσήλωση στο θέμα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Έχουμε την αγροοικονομία, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους παραγωγής τροφίμων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επιβάρυνση ε, των ε, γεών, αλλά και των ε, υδάτων λόγω των πρακτικών που εφαρμόζονται. Επίσης έχουμε την μαζική κτηνοτροφία, χρήση αντιβιωτικών δεν, δεν, δεν μπορεί να συνδυάζονται αυτά τα δύο. Ήταν ε, επίσης εξαιρετική η έκθεση του συναδέλφου Κόμπατσερ που μιλάει για υγιή τρόφιμα, υγιεινή διατροφή αλλά και για την παραγωγή τροφίμων επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη της υπαίθρου και θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω. Θα δείτε και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ότι συνιστούν σημαντική βελτίωση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Uh, και ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά. Κυρία Εισηγήτρια, μάλλον. Ευχαριστώ που προβλέψατε συζήτηση για το θέμα αυτό. Θέλω να σταθώ και πάλι στη σπατάλη των τροφίμων. Βεβαίω είμαστε κατά τη σπατάλη και αν γίνεται να υπήρχαν και μηδενικά απόβλητα από τη διατροφή. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική πρόληψη ώστε να ενημερωθούν οι πολίτε για να γίνεται σωστά η διαλογή, να γίνονται σωστέ αγορέ, να καταναλώνουν με σωστό τρόπο και να μπορούν να επαναχρησιμοποιούν τα υπόλοιπα. Προκειμένου όμω να σεβαστούμε του στόχου επισητιστική ασφάλεια, ε, υπάρχουν κανόνε που προκαλούν παρόλα αυτά ακόμη σπατάλη τροφίμων. Όλο ιδιαίτερο σκέφτομαι και έχω το νου μου στο νομό τους κανόνες για την εστίαση, την σχολική εστίαση, την ε, εστίαση πολλές φορές επίσης, την ε, δημόσια, που οδηγεί στην ε, σπατάλη το πέταγμα τροφίμων που δεν καταναλώθηκαν. Το βρίσκω λίγο αντιφατικό αυτό. Θα έπρεπε οι κανόνες να προβλέπουν να μην έχουμε τόση σπατάλη τροφίμων. Ευχαριστούμε. Εδώ θα Θέλω να δώσω ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πλευρές της αίθουσα, Ο κύριος Σβουρός. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας αφορά όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί το ξέρουμε όλοι το θέμα. Σε τι ποσοστό υπάρχει έλεγχος στα τρόφιμα τα οποία πηγαίνουν στους πολίτες και θέλουμε να είναι ασφαλή και ελεγμένα ώστε να μην καταλήξουμε στη χημική διατροφή. Σας ευχαριστώ πολύ. right, and Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Κύριε Κάιτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που άκουσα τόσο ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω πάμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση με τις απόψεις μας. Είμαστε στο ίδιο πνεύμα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να α, ε, πω ότι σημειώνω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Απλώς ένα σημαντικό θέμα αναδύθηκε από όσο ακούσαμε. Ο πρόεδρος της ομάδας ECR είπε ότι η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα. Θέλω εδώ να επιστήσω την προσοχή σας στον ορισμό της υγείας. Ο ορισμός της υγείας προκύπτει από τον ΠΟΗ. Είναι κοινωνική, ψυχολογική, σωματική ευημερία χωρί την ύπαρξη νόσων, ασθενειών κλπ. Τα υγειονομικά λοιπόν συστήματα ε, είναι σαφώ εθνική αρμοδιότητα, αναφίβολα. Αλλά όταν μιλάμε για υγεία ενιαία αγορά, για τρόφιμα και παραγωγή, Κάποιοι είπαν ότι η παραγωγή οδεύει από τη μια χώρα στην άλλη. Ε, ότι έχουμε ψηλό ποσοστά σε λιπαρά ε, ζάχαρα και άλατα και αλάτι. Αυτό μπορεί να μείνει μόνο εθνική αρμοδιότητα. Τα προβλήματα δημόσια υγεία μπορεί να παραμείνουν αποκλειστικά εθνικά. Είναι διασυνοριακά, είναι παγκόσμια θέματα πλέον. Μην μπερδεύουμε την ε, υγειονομική φροντίδα με την υγειονομική, ε, τον υγειονομικό φόβο. Εδώ μιλάμε για την κοινή αγροτική και εκτινετρική πολιτική. Ε, πρέπει να, την μάλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την υγεία σε σχέση με τους στόχους βιώσιμους ανάπτυξης, σε σχέση με τόσα πράγματα που είναι διασυνοριακά πλέον. Πρέπει να το καταλάβουμε. Τα θέματα της υγείας αφορούν το πόσο είναι σε καλή υγεία, σε ε, κατάσταση ευζοίας κάποιος έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την ε, καλή σωματική και ψυχολογική υγεία. Δεν μπορεί όλα αυτά να λειτουργήσουν αν ε, δεν συνεργαστούν όλοι οι τομείς μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε από τη στενή προοπτική ε, του αμυγός υγειονομικού τομέα. Κοινή πόρη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια πανευρωπαϊκή διατροφική πολιτική. Πανευρωπαϊκή αναθεώρηση της κοινή αγροτικής και κτηνοτροφική πολιτικής. Πρέπει να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, να σώσουμε τους υδάτινους πόρους μας, τους ε, πόρους ενέργειας. Γιατί υποβάλαμε την πρόταση για την κυκλική οικονομία. Ε, γιατί μιλάμε για τα θέματα υγείας, γιατί είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποια εργαλεία βρίσκονται στα χέρια των αρχών τοπικής αυτοδίκησης, των πόλεων, των περιφερειών, των επαρχιών. Σωστά. Όμως πρέπει να δούμε και την πανευρωπαϊκή θέμα είναι αξία όταν μιλάμε για την υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί αναφέρατε την ε, έκθεση για τις βασικές γραμμές της υγείας. Την επόμενη φορά θα φροντίσουμε να θυσιάσουμε κάτι για την κατάσταση της υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε τα θέματα που αφορούν ε, την υγεία πανευρωπαϊκά. Αναφέρατε την παιδική παχυσαρκία. Χθες στη Μάλτα διοργανώθηκε μια πραγματικά ε, έκτακτη άτυπη μάλλον σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας, όπου το θέμα τη παιδική παχυσαρκία ήταν το πιο καυτό θέμα. Ε, πρέπει εδώ λοιπόν να βρούμε τα σωστά εργαλεία. Πρέπει να βρούμε τρόπου να αναζητήσουμε λύσει, όπω με την ε, ε, έντονη διαφήμιση που να αποφαρίνει τα παιδιά την κατανάλωση των τροφίμων, με το σωστό μάρκετινγκ, με του σωστού δασμού και φόρου για προϊόντα όπω τα υνοπνευματόδη, το αλκοόλ, τα υνοπνευματόδη, τα προϊόντα καπνού και τα ζακχαρόδη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι η κοινωνική εντό εισαγωγικών Ευρώπη που ε, λέμε δεν μπορεί να μην είναι υγιής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρί την υγεία. Και σα μιλάω για τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Δεν μιλάω ούτε για νόσου, ούτε για ασθένειε, ούτε για αυτά τα φοβερά και τι απειλέ που ακούγονται σε σχέση με την υγεία. Δεν είναι η εθνική, δεν είναι η υγεία ένα θέμα αμυγό εθνικό. Ε, δεν μιλάμε μόνο για αρρώστου. Μιλάμε για ανθρώπου που θέλουμε να είναι όσο ε, το δυνατόν υγιέστεροι και όσο το δυνατόν ε, περισσότερο. Θέλουμε να έχουμε πολιτική για τη διατροφή. Μια πολιτική που να προσφέρει τη σωστή διατροφή που να θρέφει του ανθρώπου. Είμαι γιατρό, είμαι γιατρό επαγγελματία και ξέρω τι σα λέω γιατί το έχω δει στη δουλειά μου. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που κάποιοι θέλουν να υπάρξουν σχετικέ πρωτοβουλίε. Είμαστε ε, ε, έτοιμοι να συζητήσουμε θέματα για τη διαχείριση των τροφίμων και τη επιστημική ασφάλεια. Ε, ήδη έχουμε παρουσιάσει ένα πλαίσιο μεθοδολογία στην πρώτη μα συνάντηση. Θα φροντίσουμε στην επόμενη συνάντηση να δούμε πώ μπορούμε να προχωρήσουμε και όλοι μαζί να καθορίσουμε μια μεθοδολογία για να διαχειριστούμε τη σπατάλη των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας ε, παραγωγής τροφίμων από το χωράφι μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Πρέπει να είναι όλα αυτά τμήματα μιας πολιτικής διαχείρισης διαχείριση των τροφίμων. Αναφέρατε πολλοί θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των τροφίμων. Ναι, σήμερα έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε την επαναδιατύπωση της πολιτικής ε, των τροφίμων, της πατάλη των τροφίμων, αλλά δεν έχουμε μια, μια ε, διατροφική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γάλα, τα οποροκεπευτικά και τα λαχανικά στα σχολεία να εφαρμοστεί. Το είδαμε. Χρειάζεται χρήμα. Ζητήσαμε από εσά, τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, να δραστηριοποιηθείτε, να αξιοποιήσετε κονδύλια, πόρου, ό,τι υπάρχει. Γιατί πρόκειται για τα παιδιά, πρόκειται για σχολεία και νοσοκομεία. Πρόκειται για περισσότερο φρέσκο και ε, πρόσφατα παρα, και, φαγητό που έχει τρόφιμα που έχουν παραχθεί πρόσφατα που καταναλώνονται άμεσα. Εδώ αναζητούμε την επαναδιατύπωση κανόνων ε, ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν φρεσκότερα, νοπότερα τρόφιμα από τις τοπικές αγορές. Από τις λαϊκές αν γίνεται. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξετε τους γεωργούς μας. Θέλουμε να στηρίξετε τις τοπικές κοινότητες. Να μείνουν ζωντανές θέλουμε. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για τις προτάσεις, τις ιδέες σας και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο και τη συνεργασία μας θα τη συνεχίσω για να σας βεβαιώσω ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Θα παραμένουμε πιστοί στην τήρηση των υποχρεώσεων μας, των υποχρεώσεών μας και θα θέσουμε και τις πρώτες ε, ημερομηνίες ως στόχους. Να δούμε πότε θα ξανασυζητηθούν οι κανόνες αλλά και για τη σπατάλη των τροφίμων. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις εταιρείε μας να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Ναι, θα δεχτώ την πρόσκλησή σας να έρθω στη Δανία. Διότι έχω πάει στην Κοπενχάγη και είδα εξαιρετικά σχολ... εξαιρετικέ σχολέ και σχολεία όπου μαθαίνετε στα παιδιά ήδη με την αγωγή περί τροφίμων να γνωρίζουν τι τρώνε. Ήταν υποδειγματικό αυτό που είδα. Θα τη δεχτώ την πρόσκλησή σας. Θέλω να δω κι άλλε ε, καινοτόμες ε, λύσει και ιδέε. Και θέλω να δω κι άλλου ε, στο Ελσίνκι, στη Μάλτα, στην Ιταλία. Τα έχω δει κι αλλού. Ταξιδεύω πολύ και βλέπω πώς οι τοπικές κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να ξετρεπώνουν τι καλύτερε πρακτικές και να τι δείχνουν και στου υπόλοιπου. Καλή τύχη λοιπόν, εύχομαι σε όλους μας στην προσπάθεια καταπολέμησης της πατάλης των τροφίμων. Tell Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την ε, δική μου περιοχή που πολλοί δημοσιογράφοι τουλάχιστον έχουν αναφερθεί σε αυτήν ως μια βέλτιστη πρακτική για την ε, μείωση της πατάλης των τροφίμων. Δεν μιλώ για την ποιότητα, αλλά τουλάχιστον για τη μείωση της πατάλης. Σας ευχαριστώ. Ωραία, μπορούμε να ε, περάσουμε στην εξέταση της ε, γνωμοδότησης της ιδίας πρωτοβουλίας. Αρνοκόπατε. Για το ζήτημα των τροφίμων. Νομίζω παρουσιάστηκε ήδη αποτελεσματικά, ε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Όχι, ο λίγο σύντομα το λόγο. Ελάτε. Ουσιαστικά τα είπα και πριν. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, που μας προσέφεραν επιστημονική συνσφορά, τον καθηγητή Σκαμπίνκο και άλλους, ε, οι οποίοι ε, βοήθησαν ιδίως στους εμπλεκομένους ε, φορείς. Ε, έχουμε τις τροπολογίες, τις τροπολογίες που νομίζω ότι βελτιώνουν πάρα πολύ πιο ό,τι αφορά τα περιπιλωτικού προγράμματος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ένα πολιτικό, πιλωτικό συγγνώμη, πρόγραμμα. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια εγκάρσια πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Ένωση για να μπορούμε μετά να δούμε τι θα κάνουμε πρακτικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Νομίζω τα πιο πολλά τα είπα ε, σε ό,τι αφορά αυτή τη γνωμοδότηση. Πράγματι έχουμε συνεχεία ένα άλλο θέμα στη Μεσία Διάταξη που καταπιάνεται με την υγεία γιατί ουσιαστικά και τα τρόφιμα με την υγεία έχουν να κάνουν και με το well-being, την ευημερία, την ευεξία. Τα είπε και ο Επίτροπος αυτά και θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνεισέφεραν στην γνωμοδότηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψήφιση των... Α, όχι, κάποιος θέλει το λόγο πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτό που λέγεται στην γνωμοδότηση ότι θα πρέπει οι οργανώσεις, ε, ε, περιβαλλοντικοί φορείς, κυβέρνηση όλοι αυτοί οι φορείς να συμμετέχουν. Εμείς ασχολούμαστε με την πρόθεση των ε, ε θεμάτων υγείας, τροφίμων, ε, την δημιουργία δεξιοτήτων ε, προς όφελος των πολιτών. Είμαστε και μέλος του προγράμματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις Υγιείς Πόλεις. Θέλω να συγχαρώ για μια ακόμη φορά τον εισηγητή. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψήφιση των τροπολογιών. Έχουμε τρει τροπολογίε. Η πρώτη τροπολογία, ο εισηγητή υπέρ, ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδή εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθυμών 2, ο εισηγητή είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά είναι υπέρ οι περισσότεροι, εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 3, ο εισηγητής είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Κανείς λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται λοιπόν. Ε, γνωμοδότηση συνολικά όπως τροποποιήθηκε, ψήφι υπέρ. Κατά. Κανείς. Εγκρίνεται. Αποχές, συγγνώμη, τις ξέχασα. Εγκρίνεται. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή. Έφτασε ο κύριος Μπαρνιέ. Έχουμε πολύ ε, στενό χρονοδιάγραμμα, οπότε θα περάσουμε απευθείας στη συζήτηση για το Brexit και όχι στη συζήτηση της έκθεσης της κ. Uh, λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ την ε, συνεδρίασή μας. Μια σύντομη εισαγωγή εκ μέρου μου να καλωσορίσω τον ε, κύριο Μπαρνέ. Κύριε Μπαρνέ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας ε, να παρευρεθείτε στην Ολομέλεια. Είχαμε ήδη πολύ καλή συνεργασία και ο στόχος σήμερα είναι με τους περιφερειάρχες, δημάρχους, τοπικούς δημοτικούς συμβούλους να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit. Η πλειοψηφία των Βρετανών επικών έλαβε την απόφαση που έλαβε. Σίγουρα όμως αυτά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα για τις μελλοντικέ γενιές. Θα γνωρίσετε κύριε Μπαρνιό ότι παρά το γεγονός ότι το δικό σας καθήκον είναι ναι, ο τεχνικός συντονισμός ε, των διαπραγματεύσεων, οι συνέπειες δεν θα επηρεάσουν αφηρημένα μόνο κάποιες διατάξεις της συνθήκης ή χιλιάδες ε, σελίδες Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά θα επηρεάσουν σίγουρα τη ζωή κτομμυρίων πολιτών που ζουν και στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στα άλλα 27 άλλα κράτη-μέλη και θα πρέπει να προασπίσετε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Αυτή πρέπει να είναι η βασική μέρη, να πιστεύω, στην όλη αυτή διαδικασία. Πώς το Brexit θα επηρεάσει την πραγματική, την καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών, των πολιτών, των επιχειρήσεων. Σήμερα οι αιρετοί που είναι εδώ παρόντες από όλα τα 28 κράτη και από το ΕΒ θέλουν να ακούσουν και να συνομιλήσουν μαζί σας για το πώς θα επηρεάσει ε, τους ε, ε, πολίτες μας ε, στους Δήμους ε, και στις διασυνοριακές μεθοριακές περιοχές αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα διασυνοριακά. Γνωρίζουμε ότι εκτιμάται το ρόλο των αρχών της τοπικής περιφερειακής αυτοδίκησης. Μπορεί να μην έχουμε εμείς ως Επιτροπή επίσημη αρμοδιότητα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, στη διαδικασία της επικύρωσης κάποιων εμπορικών συμφωνιών, τα περιφερειακά κοινοβούλια θα ψηφίσουν, θα έχουν λόγο. Και βέβαια ε, θα υπάρξει ψήφισμα, το οποίο εμείς θα εγκρίνουμε αύριο με τις δικές μας απόψεις και εκεί μπορείτε να αναγνώσετε ανησυχίες αλλά και πιθανές λύσεις από ε, τις 28 χώρες μέλη και τις τοπικές αρχές. Τα όσα επόμενους μήνες ε, θα παραμείνουμε σε στενή επαφή μαζί σας, ώστε να δούμε κατά πόσο ορισμένες από τις δικές μας προτάσεις θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πριν ε, ολοκληρώσω, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα τον Ιανουάριο στο Λονδίνο στους φίλους μας από την Βρετανική Αντιπροσωπεία τη Επιτροπής των Περιφερειών. Το Brexit σημαίνει Brexit, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα ε, κατεβάσουμε, ε, δεν θα χαμηλώσουμε τις προσδοκίες, ε, το ύψος των φιλοδοξιών μας. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστούμε τα εθνικά περιφερειακά τοπικά συμφέροντα είναι να συνεργαζόμαστε και στη συνέχεια, έχοντα πάντα βέβαια ω γνώμονα τι κοινέ μα αξίε και αρχέ και αυτό κάναμε πάντα στο ε, πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί είμαστε και θα παραμένουμε ενωμένοι, αλλά αυτή την κρίση ε, θα πρέπει να την κάνουμε ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια. Εκ μέρου ε, ε, των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Πόλεων. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τι προτάσεις μας για λύσει ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προ όφελο των πολιτών Σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία στι διαπραγματεύσει, σα Ελπίζουμε η έκβαση να είναι μια καλή συμφωνία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση Και τώρα παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Μπαρνιέ. Ε, merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι περιφερειών, αξιότιμοι κύριοι δήμαρχοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να, σας, να συζητήσω μαζί σας και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής σας έτσι ώστε να έχουμε μια συζήτηση για την διαπραγμάτευση η οποία προβλέπεται δύσκολη, η οποία είναι πρωτοφανής και για να είμαι ειλικρινής είναι πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω δημοσίως για το θέμα αυτό. Θα μου επιτρέψετε για αυτόν τον λόγο πρώτα μάλλον να εκφράσω την αλληλεγγύη μου γιατί μαθαίνουμε ότι μπροστά στην Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο σημειώνονται επεισόδια και θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και την αλληλεγγύη μου προσωπικά στον, απέναντι στο Βρετανικό λαό και στις Βρετανικές αρχές. εδώ και 44 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν μια, ένα κοινή, κοινό στόχο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε την νέα αγορά, να εξαλείψουμε τα σύνορα, να υιοθετήσουμε κοινούς κανόνες, επι, ε, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών προσώπων και υπηρεσιών. Δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, η οποία προστίθεται στην εθνική ταυτότητα. Κάναμε τεράστια βήματα για την δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, για την ειρήνη. Στοιχεία κρίσιμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από κοινού φροντίσαμε για την επανένωση της Ευρώπης μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και καταφέραμε να υιοθετήσουμε φιλόδεξες πρωτοβουλίες, να ανοίξουμε τα σύνορά μας και να χρηματοδοτήσουμε επιμακρών την πολιτική συνοχής, η οποία βεβαίως και ε, εύλογο είναι, είχε μεγάλη σημασία για την Επιτροπή των ε, Περιφερειών, για να καταπολεμήσουμε τις ιστορικές ανισότητες που έπληταν την... και πλήττουν την Ήπειρό μας. Αυτές οι προσπάθειες θα συνεχίσουν, αλλά δυστυχώς χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού έτσι αποφάσισε η πλειοψηφία, πλειονότητα των ε, Βρετανών πολιτών. Αυτή η απόφαση των Βρετανών πολιτών μας δημιουργεί μας, ε, αυτή την εξαιρετική κατάσταση. Γνωρίζετε ότι η επίσημη επίκληση του άρθρου 50 πρόκειται να γίνει από την Βρετανική κυβέρνηση στις 29 Μαρτίου. Και από εκείνη τη στιγμή και επισήμως θα ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, η οποία θα διαρκέσει δύο χρόνια, 24 μήνες ακριβώς. Μετά την ε, επίκληση του άρθρου 50, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς επίσης και ο πρόεδρος Τάσκα του Συμβουλίου και Γιούνκερ της Επιτροπής, θα εργαστούν ε, επί κάποιες εβδομάδες για να καταλήξουν σε κατευθυντήριες γραμμές, ε, τις οποίες έχω ανάγκη, τις οποίες χρειάζομαι, για να διεξαγάγω την διαπραγμάτευση με βάση την εντολή που μου δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μας φιλοξενεί σήμερα. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, το Brexit θα έχει τεράστιες σημαντικότατες συνέπειες στο ε, ανθρώπινο επίπεδο, στο επίπεδο το οικονομικό, το κοινωνικό, το νομικό, το πολιτικό. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι εάν τελικά δεν καταλήξουμε στη συμφωνία, οι συνέπειε θα είναι ακόμα πιο σημαντικές, δραματικές. Έχουμε 4 εκατομμύρια Βρετανούς πολίτες στην Ευρώπη και όλοι οι πολίτες ε, του κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην Βρετανία θα έχουν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επανεισαγωγή ελέγχων στα σύνορα, ελέγχων ε, στη, μεταφορά εμπορευμάτων ή ακόμα και ελέγχων ε, που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην, ε, στις αεναέριες μεταφορές προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα επίσης τη διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας και τα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίω θα ήταν το πρώτο που θα πληγεί από ε, μια τέτοια αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Αυτές οι ανταλλαγές λειτουργούν σήμερα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου το, τις οποίες έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς, με 60 κράτη στις τρίτες χώρες. Και η Ευρώπη βέβαια θα πληγεί. Παρά το γεγονό ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη αγορενία αγορά και των συμφωνιών ελευθερό εμπορίου. Αυτό το σενάριο λοιπόν του να, να μην καταλήξουμε σε συμφωνία, το no deal, δεν είναι αυτό που επιθυμούμε εμείς. Εμείς επιθυμούμε συμφωνία. Εμεί επιθυμούμε να επιτύχουν οι διαπραγματεύσει, Όχι εναντίον των Βρετανών, αλλά σε συνεργασία με του Βρετανού. Γι' αυτό εξ ονόματο των 27 κρατών μελών και όλων των συνεργατών μου δηλώνω ότι η πρόθεσή μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία για την εύρυθμη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία μιας νέας εταιρική σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και, μιας και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό, πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του, του εγχειρήματο αυτού. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρώτη προϋπόθεση είναι τα 27 κρατημέλη να παραμείνουν ενωμένα. Και αυτό πάει χέρι με χέρι με τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 1η Οκτωβρίου και έχω ήδη συναντηθεί με τις κυβερνήσεις και των 27 κρατών μελών. Τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησε ένα δεύτερο γύρο επισκέψεων και επαφών στις πρωτεύουσε των κρατών μελών για να συνομιλήσω και με εκπροσώπους των κυβερνήσεων αλλά και με εκπροσώπους των ε, εθνικών κοινοβουλίων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επαγγελματικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε όλη αυτή την ε, περίοδο. Θα συνεχίσω να έχω πολύ στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον πρόεδρό του, τον ε, κ. Τάσκ, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ταγιάννη, καθώς επίσης και με όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, κύριε Μαρκουλά, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που έχω τη δυνατότητα να συζητώ μαζί σας με την Επιτροπή των Περιφερειών. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν με τα προηγούμενα καθήκοντά μου όταν ήμουν επίτροπος υπεύθυνος για την περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη. Γιατί εσείς εκφράζετε εδώ τις απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης με όλες την, την ποικιλομορφία που αυτή η αυτοδιοίκηση έχει. Όταν μιλάμε για ενότητα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ομοιομορφία. Αλλά χρειάζεται ενότητα για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις. Είναι Προ το συμφέρον μας αυτό, αλλά είναι επίσης και προ το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό θέλω να το ε, πω ξεκάθαρα στους ε, φίλους μας από το Ηνωμένο Βασίλειο και ιδίω αυτούς που βρίσκονται στην αίθουσα σήμερα. Γιατί χρειαζόμαστε και οι δύο πλευρές την Ευρώπη να είναι ενωμένη εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι η ενότητα αυτή θα σφυριλατηθεί ακόμα περισσότερο εάν την οικοδομήσουμε επί τη βάση της διαφάνειας και της μιας ανοιχτής συζήτησης. Πιστεύω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν εν κρυπτό. Δεν μπορούν να γίνουν πίσω από κλειστέ πόρτες. Θα πρέπει η διαπραγμάτευση αυτή να γίνει με διαφάνεια, να είναι ξεκάθαρο σε όλους και να εξηγούμε σε όλους ανα πάσα στιγμή τι συζητάμε και τι πράγμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εξηγήσουμε αντικειμενικά τι σημαίνει να εγκαταλείπει μια χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη χώρα που, τη, που φεύγει, αλλά επίσης και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οφείλουμε να πούμε την αλήθεια και θα πούμε την αλήθεια στους πολίτες μας, θα τους πούμε στα αλήθεια τι σημαίνει Brexit. Δεύτερη προϋπόθεση για να καταλήξουμε σε συμφωνία είναι να πάψει να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε όταν ανακοινώθηκε η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να φύγει και η οποία αφορά 4,5 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους φοιτητές που βρίσκονται στα Βρετανικά πανεπιστήμια ή επίσης Βρετανούς που βρίσκονται στα, στα, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, Πολωνούς φοιτητέ, τους Ισπανούς συνταξιούχους που μπορεί να βρίσκονται στην ε, Βρετανία ή τους Βρετανούς που έρχονται να απολαύσουν τη σύνταξή τους στην, στην Ισπανία τους Ευρωπαίους πολίτες που δουλεύουν ως γιατροί ή ως μηχανικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε είναι από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε. Εκείνοι που επέλεξαν και μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακριβώς όπως εκατομμύρια, χιλιάδες μάλλον άλλοι πολίτες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στο Βερολίνο, στην Ιταλία και αλλού. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανησυχούν και είναι εύλογο και θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να ε, διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι αυτό προτεραιότητά μας από την αρχή των διαπραγματεύσεων και θα συνεχιστεί ως το τέλος. Το σύνθημά μας θα είναι πρώτα οι πολίτες. Και υπ' αυτή την έννοια καλωσορίζω την απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων να ε, εγγράψει δύο ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών για το θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι περίπλοκο γιατί αφορά το δικαίωμα παραμονής, την πρόσβαση στην ε, αγορά εργασίας, την πρόσβαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στο σύστημα υγείας, στην εκπαίδευση. Θα εργαστούμε μεθοδικά για καθένα από αυτά τα θέματα και δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία λεπτομέρεια χωρίς να τη συζητήσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ε, προετοιμαζόμαστε σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη από αυτών των θεμάτων. Θα χρειαστεί χρόνος. Σίγουρα αρκετούς μήνες θα χρειαστούμε. Αλλά πρέπει να εργαστούμε σοβαρά στο θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους φίλους μας από τη Βρετανία. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, σύντομα όσον αφορά τις βαθικές αρχές, δηλαδή την αμοιβαιότητα, την συνέχεια και την μη διάκριση. Έτσι ώστε αυτοί οι πολίτες να πάψουν να αμφιβάλλουν για το μέλλον τους, να φοβούνται για το μέλλον τους. Κυρίε και κύριοι, το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε είναι η εφηβαιότητα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ και καθώ επίση για όλα τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Γιατί συζητούμε. Συζητούμε για τους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπου περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ ε, αποδίδονται για να βοηθήσουμε εκείνους τους πολίτες της Ένωσης, άνδρες και γυναίκες που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο πολύ καλά το γνωρίζετε όλοι σας. Εδώ μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, βοήθεια η οποία απευθύνεται σε περιφέρειες και πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ε, οικονομικές δυσκολίες, ε, δυσκολίες να αναπτυχθούν ή στις εξόχως απόνιτρες περιοχές τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ιούνκερ του λεγόμενου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που το, μέσω του οποίου χρηματοδοτούμε δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αιωλικές ε, ε καταστάσεις, ε, ε, βελτίωση του συστήματος υγείας, συμπεριλαμβανομένων και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προγράμματα έρευνας που χρηματοδοτούνται από τον ορίζοντα 2020 80 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται για επιστημονική έρευνα, για έρευνα και ανάπτυξη μέσω του ορίζοντα. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά τα προγράμματα, για όλα αυτά τα προγράμματα συμφωνήσαμε όλοι μαζί όταν ήμασταν 28 κράτη-μέλη μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα χρηματοδοτούμε από κοινού και τα 28 κράτη-μέλη και εποφελούμαστε και 28 χώρες από αυτά. Κάθε κράτος μέλος, κάθε χώρα οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι όλων των υπολείπων. Και για να είμαι τελείως ξεκάθαρος, όταν μια χώρα αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει ένα πρόστιμο που τη επιβάλλουμε επειδή φεύγει, αλλά πρέπει να τακτοποιήσουμε του λογαριασμού μα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν θα ζητήσουμε από τη Βρετανία να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για κάτι για το οποίο δεν συμφώνησε και δεν έβαλε την υπογραφή της όταν ήταν κράτος μέλος. Αλλά και εμείς 27 που παραμένουμε θα τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, των πολιτών του και των περιφερειών του. Αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνο τρόπος κατά την άποψή μου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να πω και επιτρέψτε μου να επικαλεστώ μάλλον τα λόγια του Winston Churchill. Η τιμή που πρέπει να πληρώσει κανείς για να μεγαλουργεί είναι η υπευθυνότητα. Αυτό ισχύει και για τη Βρετανία, αυτό ισχύει και για μας. Η απόφαση του, του, του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ασφάλεια και όσον αφορά τα νέα σύνορα της Ευρώπης και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην Ιρλανδία. Γνωρίζω την πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και για να διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις εγκύτριες της συμφωνίας αυτής. Γι' αυτό και προσωπικά θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει ε, το Brexit σε αυτόν τον τομέα. Το ζήτημα της ε, τελωνιακής ένωσης. Αυτό μπορεί να συζητηθεί, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύσουμε την ειρήνη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και μια τρίτη προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με τρόπο οργανωμένο. Και προσεκτικό. Θέλω η συζήτηση για τη νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει επί τη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και αυτό, πρέπει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα θα συμφωνήσουμε επί των βασικών αρχών, επί του πώς θα γίνει οργανωμένα η αποχώρηση, έτσι ώστε να έχουμε μία ε, συζήτηση με εμπιστοσύνη για την μελλοντική μας σχέση. Όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για την οργανωμένη αποχώρηση, για την τακτική αποχώρηση, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη μελλοντική σχέση. Όσο καθυστερεί η συζήτηση για την αποχώρηση, τόσο δυστυχώ θα ε, μετατίθεται για το μέλλον η όποια συζήτηση για τη μελλοντική σχέση και τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της αποτυχίας. Κυρίε και κύριοι, η κατάσταση και η συζήτηση αυτή και αυτή τη διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη, αλλά εγώ ε, έχω μια εμπειρία από τις διάφορους θόκους τους οποίους βρέθηκα, ότι τα εμπόδια είναι πιο εύκολο να τα υπερπηδήσει κανείς όταν βλέπει μπροστά, όταν τα βλέπει στη σωστή τους διάσταση τα προβλήματα και προσπαθεί να σκεφτεί τι θα γίνει στο μέλλον, πού θα πάμε μετά. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και ποια είναι αυτή η νέα προοπτική, είναι ακριβώς η νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασίλειου. Από την πρώτη φορά που ψήφισα ως, ε, το 72 ως νέος Γάλλος για να επιτραπεί η ε, προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή κοινότητα, γιατί θα θυμάστε οι παλαιότεροι ότι εμείς κάναμε δημοψήφισμα για αυτό το 72. Θυμάμαι ότι αυτό που μας, συνδέει και, μας συνέβη και μας συνδέει με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κοινέ αξίες και κοινά συμφέροντα. Επομένως μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι νωρίς για να πούμε ποιε θα είναι οι βασικές γενικές αρχές αυτής της νέας συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, ελευθέρων ανταλλαγών η οποία όμως δεν θα μοιάζει με καμία από τις υφιστάμενες. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση. Επομένως, σε δύο χρόνια από σήμερα θα είναι τρίτη χώρα. Σε δύο χρόνια θα είναι τρίτη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε αυτή την επιλογή, το οποίο αυτόματα το οδηγεί να βρίσκεται σε δυσμενέτεστερη θέση από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον αλλά κάρτ να συμμετέχει στην ενιαία αγορά. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο στην ευρωπαϊκή ιστορία για να βασιστούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη συμφωνία εμπορική συνεργασία. Γιατί μέχρι στιγμή όλε οι συμφωνίε τη εμπορική συνεργασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει με πάνω από 60 κράτη τρίτες χώρες, ο Καναδάς πρόσφατα, η Νότια Κορέα, όλες αυτές οι συμφωνίες βασίζονταν σε μια σύγκληση των ρυθμιστικών πλαισίων. Στο Brexit έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί σήμερα τα, τα πρότυπα, τα ευρωπαϊκά, αποτελούν πρότυπο και το Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι το σημείο εκκίνησης της, διαπρα... της διαπραγμάτευσης. δεν μιλούμε πλέον για μια σύγκληση στο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά περισσότερο για το κίνδυνο ε, που δημιουργεί η πιθανότητα της απόκλησης της σταδιακής, δηλαδή του να ξεφύγουν σιγά σιγά αυτά τα δύο ρυθμιστικά πλαίσια. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό και θα, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι ώστε η, αυτή η πιθανή απόκληση, απομάκρυνση του Ηνωμένου Βασιλείου από το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο να μην οδηγήσει σε dumping Πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι, ε, να, να κρατηθούν, να, είναι ενήμεροι για όλα αυτά και να συμμετάσχουν. Πρέπει να σκεφτούμε πόσες αντιθέσεις και πόσες α, παρεξηγήσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια Συμφωνία Ελευθέρου Εμπειρίου, την οποία ας μην ξεχνάμε ότι θα πρόκειται για μια μεικτή του χαρακτήρα συμφωνία ε, εμπορικής συνεργασίας και άρα θα πρέπει να ε, επικυρωθεί από όλα τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κανόνες δίκαιους, θα, οι οποίοι δεν θα δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, δεν θα επιτρέπουν τον ντάμπικ. Αυτό νομίζω θα είναι κέρια σημασίας. Συμφωνώ με την ε, ε, Υφυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, την κυρία Μέη, ότι χρειαζόμαστε μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου φιλόδοξη, ambitious. Ναι, μπορούμε. Αλλά η φιλοδοξία αυτή, εγώ την ερμηνεύω ως μια φιλοδοξία η οποία εφαρμόζεται και στα πρότυπα, τα φορολογικά, τα εργατικά, προστασίας του καταναλωτή και τα περιβαλλοντικά. Θέματα τα οποία δικαίως απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε μια κοινότητα συμφερόντων σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί ξεπερνά το στενό εμπορικό πλαίσιο. Αυτό που έλεγα προηγουμένως αφορά και την έρευνα και την κοινοτομία, τα πανεπιστήμια μας, τα εργαστήρια μας. Ακόμη και αν το ρυθμιστικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της τωρινής μας συνεργασίας προφανώς θα αλλάξει στο μέλλον. Η φιλοδοξία παραμένει και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πετύχουμε περισσότερα ε, μένοντας ενωμένοι στο πνεύμα των δεσμεύσεων που ήδη αναλάβαμε από κοινού στην διάσκεψη των Παρισιών. Την φιλοδοξία επίσης τη διατηρούμε και στα θέματα διεθνούς συνεργασίας, στην ανάπτυξη κυρίως την ανάπτυξη που προσπαθούμε να φέρουμε στην γειτονική ήπειρό μας, αυτή την Αφρική, αλλά και στην εξωτερική πολιτική, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην ανταλλαγή των πληροφοριών, στην ε, καταπολέμηση των ε, υβριδικών απειλών ή των απειλών στον κυβερνοχώρο. Το λέω σήμερα, ε, έχοντας κατά νου τα θύματα των όσων συνέβησαν στο Λονδίνο, αλλά και με τη σκέψη μου στραμμένη στα θύματα των ε, επιθέσεων στι Βρυξέλλε εδώ πέρσι στι 22 Μαρτίου, αλλά και σε όλα τα θύματα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Την ίδια φιλοδοξία την έχουμε σε θέματα άμυνα. Στο επίπεδο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο πάντοτε είχε πολύ ενεργό ρόλο με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και το ίδιο θα συνεχίσει να ισχύει, αλλά και σε πολλέ επιχειρήσει τη Ευρώπη με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια και άμυνα οι προσπάθειες που θα ε, αναλυθούν από τους 27 για την δική τους άμυνα και βάσει των προτάσεων που έγιναν πρόσφατα από την Φεντερίκα Μογκερίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει δυνατότητες συνεργασίας, διμερούς συνεργασίας, την κατάλληλη στιγμή σε συνεργασία με το, με το Βασίλειο. Διότι τώρα, ε, κυρίες και κύριοι, ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παζαρέψουμε. Η ασφάλεια δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά και στην ίδια, στη ίδιο ζύγι μαζί με, την, με το εμπόριο ή τα εμπορικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσουμε για το πλαίσιο, το περίγραμμα αυτή τη νέα εταιρική σχέση. Θα προβλέψουμε την απαραίτητη μεταβατική περίοδο. Χρειάζεται χρόνο για να διαμορφωθεί η εταιρική σχέση, για να δούμε αν θα είναι συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή κάποια άλλη μορφή συνεργασία. Αυτή η μεταβατική περίοδο θα είναι απαραίτητη και θα πρέπει να δούμε, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, είναι πολύ νωρί, θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί και όλε αυτέ οι προσαρμογέ θα ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και όσε νομοθετικέ πράξει προκύπτουν από αυτό. Βεβαίω θα φροντίσουμε να περιοριστούμε στα απολύτω αναγκαία και σε όλε τι περιπτώσει δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει αλακάρτ ε, κοινή αγορά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να ολοκληρώσω αυτήν την παρουσίαση, Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι θα ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουν αυτές οι δυσχερείς διαπραγματεύσεις. Είμαστε σταθεροί αλλά και φιλικοί. Δεν είμαστε όμως ούτε αφελείς. Θα σας τα πω ξεκάθαρα σήμερα, κύριε Πρόεδρε ώστε όλοι να καταλάβουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις της επιτυχίας των διαπραγματεύσεων. Να εργαστούμε ε, μαζί και οι 27 μόνιμα σε πνεύμα διαφάνειας και σε επίπεδο δημόσιο ε, γρήγορα να αρθούν όλες οι σκιές που ρίχνουν οι προθέσεις των Βρετανών να φύγουν από την Ένωση, οι πολίτες να καθησυχαστούν και να μπορέσουμε να αποφεληθούμε πλήρως από τον προπολογισμό και τα όσα ε, προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, όλα να μπουν σε τάξη και γρήγορα σε μια προοπτική για το μέλλον. Με γερά θεμέλια για να συζητήσουμε και τη μελλοντική μα σχέση με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Και μια και μιλώ για το μέλλον των 27, το κοινό μα μέλλον είναι περιττό να επιμείνω στο ότι οι προκλήσει και οι δυσκολίε τη νέα ε, ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται απλώ και μόνο στο Brexit η προτεραιότητα είναι και παραμένει να ενισχύσουμε και όταν χρειαστεί να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή μα Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τι κοινέ προκλήσει που έχουμε απέναντί μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προέδρου τη, του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή δημοσιεύοντα πρόσφατα τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον τη Ευρώπη. Την εβδομάδα αυτή, μεθαύριο, οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν στη Ρώμη για να εορτάσουν τα 60 χρόνια από την υπογραφή τη συνθήκη τη Ρώμη τη συνθήκη ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, παρά την κρίση, παρά το Brexit, παρά τι δυσκολίε, αυτή η γιορτή, η επέτειο τη Ρώμη, δεν θέλουμε να είναι ε, παρελθοντολαχνική και στραμμένη προ το παρελθόν. Όχι. Είναι η στιγμή εμείς ε, οι 27 να κάνουμε μια νέα αρχή για την Ένωση και για να υπάρξει δράση. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το πλαίσιο που έχουμε τώρα μπροστά μας. 14 παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρός με το όριο ομιλίας. Πιο σύντομη παρακαλώ από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Ας σας ακούσουμε όμως και μετά ίσως απαντήσει ο Επίτροπος. Πρώτη παρέμβαση, τριλεπτή από το ΕΛΚ, ο κύριος Μέρφυ. Εκ μέρους του του ΕΛΚ. Θα ήθελα κύριε Μπαρνία να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα αποτελέσει τμήμα ενό ε, συνεχιζόμενου διάλογου. Ω Ευρωπαίο, ε, σήμερα λυπούμε ιδιαίτερα για την απόφαση του Ηνωμένου Βασίλειου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, μετά από μακρά περίοδο οικοτολογίας πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο όπου πλέον πρέπει να βρεθούν λύσεις στις προκλήσεις που θέτει το Brexit τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ μεγάλο μέρος του πιθανού αντικτύπου του Brexit θα είναι άμεσα αισθητό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία, από μια περιοχή που έχουμε σημαντικό γεωργοδιατροφικό τομέα. Ο κόσμος φοβάται για τα περιουσιακά του στοιχεία. Φοβάται για το μέλλον του. Ο Ιρλανδικός τομέας λοιπόν αυτός είναι εκτεθειμένος ε, ε, στη συμφωνία του Brexit εφόσον περιορίζει το εμπόριο και μόνο στον τομέα αυτό το γεωργοδιατροφικό το ποσοστό εξαγωγών από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πενταπλάσιος του μέσου όρου της Ένωσης. Κύριε Μπαρνιέ, πραγματικά χαιρετίζω αυτό που είπατε σε σχέση με το ότι δεν θα πρέπει κανένα κράτος μέλος ε, να είναι σε χειρότερη θέση. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να στηρίξετε τη χαλάρωση των κανόν περί κρατικών ενισχύσεων για περιοχές, για τομείς που δεν περιορίζονται μόνο βέβαια στον Ιρλανδικό γεωργοδιατροφικό τομέα αλλά που θα πληγούν ε, και ξέρω ότι και εσείς και η ομάδα σας αντιλαμβάνεστε απόλυτα τα ζητήματα που αφορούν ε, τα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία και είστε προσιλωμένο στην προσπάθεια εξέβρεση λύσης. Είναι τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, η Βόρεια Ιρλανδία περιλαμβάνει 1,7 εκατομμύρια ε, κατοίκου. Το μπορούσαν να ζητήσουν την Ιρλανδική ή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια μια κακή συμφωνία θα μπορούσε να μας γυρίσει πίσω και να ανατρέψει την πρόοδο των τελευταίων 20 ετών, τιμωρώντας τους πολίτες και των δύο πλευρών αυτής της διαπραγμάτευσης. Κύριε Μπαρνιέ, Ποια είναι η άποψή σας, ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, ε, ανατροπή της καλής κατάστασης που υπάρχει τώρα. Πώς δεν θα διαταραχθούν οι σχέσεις Βορρανότου, θα συνεργαστεί η Ένωση με την Ιρλανδία, ώστε να μην υπάρχει σκληρά, να μην υπάρχουν σκληρά σύνορα εκ νέου στην, στο νησί και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι 27 που θα μείνουμε θα συνεργαστούμε ούτω ώστε να διατηρήσουμε ένα θετικό όραμα ε, για του συμπολίτε μα ότι αυτό το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εστιάσουμε στι προτεραιότητέ μα. Ασφάλεια, απασχόληση, ε, ανάπτυξη, καταπολέμηση των προκλήσεων του μεταναστευτικού προσφυγικού. Θέλω να σα πω επίσης ότι ένας απεσιόδοξος τις ευκαιρίες τις βλέπει γεμάτες δυσκολίες. Εμείς στο ΕΛΚ όμως είμαστε αισιόδοξοι και εμείς βλέπουμε σε κάθε δυσκολία ευκαιρίες. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ ο Μάρκος από την ε, Γερμανία τώρα έχει το λόγο τρία λεπτά κι εσείς. Δεν ξέρω θα μου φτάσουν τα τρία τέλο πάντων, σίγουρα στα θύματα του Λονδίνου είναι η πρώτη μου σκέψη και ιδίω σήμερα που έχουμε την επέτειο του ενό χρόνου από τι επιθέσεις ε, στις Βρυξέλλες. Πραγματικά ε, με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση έμαθα αυτό το νέο. Κύριε Μπαρνιέ, πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, των οποίων γείστε θα είναι από τι πιο σκληρές, σκληρότερε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα υπάρχουν πολλές ανησυχίες, διότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο τα συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να προασπίσουμε. Είναι θέμα επίσης αξιών ε, και ανθρώπους αξιοπρέπειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι ε, έχουν ε, καταφέρει να έρθουν κοντά και παρά τις διαφορετικές καταστάσεις και τη γεωγραφική τους θέση και χρησιμοποιήσαμε την αρχή της ελεύθερης διακίνησης, ελεύθερης κυκλοφορίας κυκλοφορίας. Μπορεί ε, κάποιο να ζει, ένας βρετανός στη Βρετανία ή να ζει σε μια άλλη Ευρωπαϊκή, ε, χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πώς ε, θα εξελιχθεί η κατάσταση για αυτού του ανθρώπου, Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Citizens first, πρώτα οι πολίτε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή και πρέπει να το δούμε. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν επηρεάσει και τις περιφέρειες ε, και ε, πρώτα απ' όλα βέβαια την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία που συνορεύουν ε, και τον Ορπάντ Καλέ, αλλά και στις επόλοιπες χώρες που υπάρχει μεγάλη πρόσβαση. Έχουμε τη Βόρεια Ιρλανδία Βεσφαλία για παράδειγμα που δεν θα είχαμε υπάρξει καν ως ομόσπονδο αν δεν υπήρχε η Βρετανία. Έχοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση και σε ό,τι αφορά και το ΣΕΤΑ και τις διαπραγματεύσεις. Είδαμε πόσο πολύπλοκες ήταν οι διαπραγματεύσει και πόσο θα είναι και με το Brexit. Νομίζω το προδικάζουν. Ε, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο και ε, οι άλλες εμπορικές συμφωνίες σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσουν και οι αξίες μας όμως. Επίσης, τι θα γίνει ε, με την προοπτική του Brexit από την τοπική και περιφερειακή σκοπιά. Μετά από ένα ε, πιθανό ε, Brexit, δεν θα έχουμε μια πιο εντατική σχέση και σχέση σε πολλά επίπεδα με οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα όσο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ για το άρθρο 50 που δεν απαγορεύει ότι μπορεί να αποσύρει ένα κράτος μέλος ε, την αίτησή του για αποχώρηση. Έχουμε αυτή τη διαδικασία, ε, δεν ξέρω υπάρχει αυτή η δυνατότητα πράγματι ή όχι. Μπέρντ Σόμερ από το Βέλγιο και την Άλντε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, το Brexit είναι μια ήττα ε, ε, ηθική και οικονομική και ανθρώπινη, εκτός από οικονομική και εμπορική. Είναι σαφές ότι ε, θα κάνετε ό,τι μπορείτε και μας εξηγήσατε ποιες είναι οι αρχές, οι σαφείς αρχές τις οποίες θα ακολουθήσετε. Αλλά η συμφωνία για το Brexit δεν θα μπορεί να δίνει καλύτερες προϋποθέσεις από ότι η ίδια η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω χάρη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε καμία περίπτωση. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν, τρεις παρατρήσεις. Οι πολίτες, οι πολίτες του ΕΒ που θέλουν να είναι Ευρωπαίοι, θέλουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ε, δημιουργικές λύσεις μπορούμε να βρούμε. Αυτοί που αισθάνονται ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μπορούμε να βρούμε τρόπο για να συμμετέχουν Δεύτερον, ο αντίκτυπος των ε, τοπικών και περιφερειακών αποκλήσεων. Κάποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο από άλλες. Η Βόρεια Ιρλανδία, η Ιρλανδία ίδια. Ε, θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες αλλά και θέματα ασφάλειας. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και για τον προπολογισμό. Τι μπορεί να γίνει ώστε οι προπολογισμοί να μην πληγούν πώς θα καλύψουμε το κενό που θα προκύψει, την τρύπα στον προπολογισμό. Πώς θα μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι οι ανάγκες μας θα καλύπτονται του ή Και για το δικό μας το θεσμικό όργανο, την Επιτροπή των Περιφερειών, είναι υποχρέωσή μας να έρθουμε σε επαφή με τις δημοτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Αγγλία, τη Σκοτία, το Λονδίνο, για να δούμε με έναν διάλογο που θα οργανώσουμε πώς μπορούμε από κοινού να συζητήσουμε το μέλλον μας. Είμαστε σε ένα αχαρτογράφητο πεδίο που κανείς ως τώρα δεν έχει εξερευνήσει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Η, από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία. τον κύριε Μπαρνί, ε, της ομάδας μου σηκώνομαι για να μιλήσω ως ε, περήφανος Σκοτσέζος και φιλοευρωπαίος ε, και ελπίζω και εμείς να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο μέλλον της ευρωπαϊκής συζήτησης ως πλήρες μέλος, ως σκοτία δηλαδή, ως πλήρες μέλος της Ένωσης. Πρέπει να συνεργαστούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και μας βοήθησε. Έδωσε τη δυνατότητα ε, στον κόσμο να μπορεί να ζήσει, να εργαστεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευεργετικό και για τους Σκοτσέζους σε, όλες, ε, σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε λοιπόν μέχρι τώρα ω μέλο του Μεροσύλλου. Ελπίζουμε να συμμετέχουμε στι μελλοντικέ συζητήσει ω ανεξάρτητο πλήρε μέλο ε, τη ε, Ένωση. 62% ε, είναι υπέρ του Remain στη Σκωτία και ιδίω οι τοπικέ περιφερειακέ αρχέ τη Σκωτίας και το Συμβούλιο των Τοπικών Περιφερειακών Αρχών ε, που στηρίζει ε, και εγώ προσωπικά ε, θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους και στη συνέχεια είμαστε μπροστά από ένα δύσκολο μέλλον. Θα απειληθούν με ένα Brexit χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έχουμε πρόβλημα με τις εξαγωγές τροφίμων, ποτών. 5,5 δις ήταν η άνοδος ε, ε, του τζίρου σε σχέση με το προηγούμενο έτσι. Όλα αυτά θα επηρεαστούν. Το Brexit θα επηρεάσει ιδίως εξέλιξη στο τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε, θα απεμπολίσουν οι πολίτες κάποια δικαιώματά τους, ε, θα χάσουν κάποιες δυνατότητες, γεωργία, περιβάλλον, αλληλεία, ε, κλίμα, COP21, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και λίγα σας λέω. Η Σκοτία ε, είναι ευρωπαϊκή, είναι στην Ευρώπη, θέλουμε να διακόπτεται Χαιρετίζουμε το ψήφισμα και ελπίζουμε στη συνέχεια του διαλόγου. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, λέει ο πρόεδρο, είναι η Τζούντιτ Wallis από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, να σα καλωσορίσω, κύριε Μπαρνιέ, στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μεγάλο αντίκτυπο ε, και κοιτάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το τι στάσει θα τηρήσουν και οι δημοτικέ αρχέ. Θέλουμε σε αυτέ τι διαπραγματεύσει να λάβετε υπόψη σα ε, τι περιφερειακέ και τοπικέ κυβερνήσει στην όλη διαδικασία για να βεβαιωθούμε ότι θα βρεθεί σωστή ισορροπία που θα είναι αποφελή για όλου. Η αποχώρηση ενό μέλου από την Ένωση δεν είναι ένα ε, θέμα που δεν θα έχει καθόλου επιπτώσει. Κοινωνικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα είναι αλληλένδετα σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο και για του ε, τελικού χρήστε και δικαιούχου τη συμφωνία που θα επιτευχθεί. Ω ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είχαμε διάλογο με διάφορου εκπροσώπου των ε, κυβερνήσεων, ε, των τοπικών φορέων από τη στιγμή του δημοψηφίσματο και μετά. Ασχέτω των απόψεων που είχαν για την αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρξει διαρκή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και των άλλων 27 κατομελών. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν κοινά συμφερόντα και προκλήσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία στι συζητήσει μα για το μέλλον τη Ευρώπη να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι το μέλλον τη Ευρώπη συνολικά θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά του τη δυνατότητά τη να λειτουργήσει συνολικά, ε, ακόμα και με τι χώρε που είναι μέρο τη Επίρου, χωρί να είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ανάγκη να νομοθετούμε μαζί για να ευημερίσουμε μαζί. Υπάρχουν συγκεκριμένε περιοχέ όπου θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ε, διαχείριση των αποβλήτων, την θεκτικότητα, την διαχείριση τη ενέργεια, την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Εδώ, ένα χρόνο μετά από τι επιθέσει ε, στην Βρυξέλλε, βλέπουμε ότι συμβαίνει το ίδιο αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Εδώ λοιπόν ε, η αυτοδιακυβέρνηση είναι δικαίωμα όσων θέλουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουμε σε συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όσα προβλέπει το άρθρο 8. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ε, Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για να υπάρξει ευημερία για όλους τους πολίτες και ελπίζουμε οι διαπραγματεύσει να προχωρήσουν ομαλά. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου ε, τη Εθνική ε, Βρετανική Αντιπροσωπεία, ο κύριο Χάτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εκ μέρου των τοπικών κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσωπώντα την Ουαλία, τη Σκωτία και την Βόρεια Ιρλανδία. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για την επίσκεψή σας στο Λονδίνο τον Ιανουάριο και την συζήτηση με την αντιπροσωπεία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Υπουργό που ασχολείται με τα θέματα Brexit. Πρέπει να υπάρξει εντατικό διάλογο μεταξύ μα. Οι, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να ε, συνεργάζονται με του ομολόγου του στην Ευρώπη των 27. Θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να ε, μπορέσουμε να έχουμε μια σχέση συνεργασία και μετά, ώστε οι ιδέε μα και οι απόψει μα να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα από τη μια και από την άλλη μεριά. Θέλουμε να μην ξεχνάμε ότι οι εμπορικέ μα σχέσει θα πρέπει να ε, συνεχιστούν. Οι γεωργικοί κτηνοτροφοί μα θα πρέπει να συνεχίσουν τι εξαγωγέ του. Οι νέοι μα φοιτητέ μα θα, θέλουν να συνεχί... θα συνεχίσουν να θέλουν να σπουδάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην οικονομική περίθαλψη και ω όλα τα δικαιώματα που μας κάνουν στους πολίτες με τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να βασιστούμε σε τρεις κοινέ αρχές. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και αν γίνει με τον Brexit, θα πρέπει μέρος ε, της ε, ε, ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων να μεταφερθεί στο επίπεδο των τοπικών κυβερνήσεων. Επίση, οι δημόσιε υπηρεσίε θα πρέπει να σχεδιαστούν περισσότερο στο τοπικό επίπεδο και μετά θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική αυτονομία για τι τοπικέ αρχέ του ΕΒ. Θα πρέπει, Πρόεδρε, ε, να ε, ευχηθούμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει κατά τρόπο ώστε οι τοπικέ και περιφερειακέ κυβερνήσει να ελπίζουν και να συνεχίσουν να υποφελούνται από μια στενή συνεργασία. Θα πρέπει από προγράμματα όπω το Erasmus, η Ευρώπη 2020 και το καταξύ να μπορούσαμε να συνεχίσουμε να υποφελούμαστε. Γι' αυτό λοιπόν σα ευχαριστώ να ε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Κάτι που είναι. Ευχαριστούμε. Ε, έληξε ο χρόνο σα και τώρα μερικές μονόλεπτε παρεμβάσει. Ο κύριο Κορδιέρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Μπαρνιέ, το όνομά μου είναι Βάσο Κορδεϊρό, ε, εκπροσωπώ τις Ασόρες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρχει διαφορετικό αντίκτυπο στι διάφορε περιοχέ τη Ευρώπη από το Brexit. Και σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Μια ερώτηση που είναι σε τι βαθμό μπορούμε να ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα α, λάβει υπόψη τη ακριβώ τι διαφορετικέ συνέπειε που θα υπάρχουν και στι περιοχέ του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι επιπτώσει από άλλε περιοχέ τη Ευρώπη προ το Ηνωμένο Βασίλειο πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη ε, και μάλιστα όσο το δυνατόν πιο άμεσα στις εργασίες σας. Έπειτα, για τις ε, συνέπειες του Brexit, τον προπολογισμό της Ένωσης. Είναι άλλος ένας λόγος που μας κάνει να ανησυχούμε. Υπάρχει και το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία που προκύπτει για να πλήξουν μια από τις θεμελιώδεις αρχές, την πολιτική της συνοχής. Ποια είναι η απόψή σας για το θέμα. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό είναι πραγματικά λίγο. Προσπαθείτε να έχετε μία ερώτηση για να προλαβαίνουμε. Η κυρία Χουντάτ. I'm sorry, I'm sorry, Mr. President. I wasn't... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν είχα προετοιμαστεί δεν είχα καν καταλάβει όμω τον κατάλογο των ομιλητών, συγγνώμη. Ε, κυρία Φρίχελ. Σα ευχαριστώ κύριε Παγνιέ για την παρουσία σα εδώ. Μια και έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου, θα σα ρωτήσω αμέσω. Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται ο ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ειρηνευτική διαδικασία στην Βόρεια Ιρλανδία και για την διασυνοριακή συνεργασία εντό Ιρλανδία. Ε, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της, ε, του ερηνευτικού σχεδίου και την δημιουργία σχέσεων σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε αυτό το κεκτημένο και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Μπαχνία που το αναφέρατε και μόνο σας και αναφέρατε την Βόρεια Ερλανδία και τη σημασία που έχει και γενικότερα για την Ερλανδία. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Μπορούμε να σκεφτούμε, να, να, να θυμηθούμε τι συνέβαινε πριν λίγα χρόνια στη Βόρεια Ιρλανδία και σήμερα αυτά που έχουμε πετύχει τα θεωρούμε δεδομένα. Είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία ε, όποιε διαπραγματεύσει για το Brexit να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην θέσουν ένα αμφιβόλο την ευαίσθητη ε, ισορροπία που έχει δημιουργηθεί με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριος Στένσον, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαγνιέ εκπροσωπώ μια μικρή περιοχή η οποία βρίσκεται στο σύνορο με τη Βόρεια Ιρλανδία και χαίρομαι για το γεγονό ότι αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Εγώ έχω τρία κυρία μηνύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φερθεί με σωστό τρόπο εναντί των κρατών μελών τη και ιδιαίτερα την Ιρλανδία. Και θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρο. Η Ιρλανδία θα παραμείνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήρε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για το Βόρειο τη Βόρεια Ιρλανδία. Εσεί ω Επίτροπο είχατε εργαστεί για την ειρηνευτική διαδικασία και το εκτιμούμε αυτό. Οι πολίτε οι Ιρλανδοί και από τι δύο πλευρέ του συνόρου ανησυχούν. για το, για, το, για το μέλλον αυτής της, της, της συμφωνίας. Επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, τι θα γίνει στο μέλλον για να μην γυρίσουμε στις μαύρες ε, σελίδες του παρελθόντος θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ειρήνη για ολόκληρο τον, την ίσο της Ιρλανδίας. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, αλλά εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία θα έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες θα πρέπει να αναγνωριστεί ε, πολιτικά, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιοχές αυτές με πνεύμα αλληλεγγύη να κάνουν ένα βήμα προ τα μπρο. Ναι, ε, λέει ο κύριος Πρόεδρο, ε, κρατώ τη λέξη αλληλεγγύη, είναι σημαντική. Έχω καταγράψει οκτώ ομιλητές. Bill, Schaeffer, Spiridon, Spiridos, Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then Jean-François Barnier. Can we close on that? That's... Μπορώ να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν έχουμε άλλο χρόνο θα, ξεφύγουμε από το πρόγραμμα. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Ένα λεπτό ο καθένα, παρακαλώ. Κύριο Λάμπρετ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και ε, την Επιτροπή και τον, Επιτροπ... τον πρώην Επιτρόπο Μπαρνί και να πω ότι εμείς βλέπουμε τα πράγματα ίσως και με τα εθνικά γυαλιά ε, αλλά και με τα περιφερειακά και σίγουρα υπάρχουν πολλές διαφορές και σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχουμε επιπτώσει, ιδίω στη Δυτική Ευρώπη. Για την Ολλανδία, από την οποία προέρχομαι, και τι ε, φλαμαντόφωνε περιοχέ θα είναι αισθητέ οι συνέπειε. Ε, και η Ιρλανδία σίγουρα θα πληγεί, αλλά και οι κάτω Πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πληγούν εξίσου οι κάτω Δεν το θέλαμε τον Brexit, αλλά θα μα επηρεάσει. Η Ολλανδική αντιπροσωπεία Πρέπει να σας πω ότι το κόστος το υπολογίζει 17 δις Είναι σημαντική εμπορική εταιρεία η Ολλανδία και το Βασίλειο. Τεράστιες επιπτώσεις στο Ρότερνταμ και στο Σκρίνταμ και πολύ σημαντικές και οικονομικές οι συνέπειες. Ε, καλό τον κύριο Μπαρνέ να το περιλάβει στις διαπραγματεύσεις στο σημείο αυτό και σε έξι μήνες να μας πει τι πρόοδος έχει επιτελεστεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ε, από Ευχαριστώ, Μισελ. Ε, μην το πάρεις προσωπικά. Αλλά την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, με εξυπηρέτησες με διάφορα θέματα που με απασχολούσαν εδώ στις Βρυξέλλες αυτό δείχνει το επίπεδο φιλοδοξιών με το οποίο εργάζεσαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Τώρα, για αυτό που θα συμφωνήσουμε και αύριο ως κείμενο, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία που να δείχνει ότι είναι καλύτερο να μην συμμετέχει κανεί στην Ένωση από όταν είναι μέλο. Αυτό το δεχόμαστε όλοι εδώ στην Ολομέλεια. Όμω πρέπει να γίνεται κατανοητό και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Βρετανική κυβέρνηση και από του πολίτε του Ηνωμένου ε, Βεβαίω, όπω προχωρούμε προ την επιστολή περί του άρθρου 50. Είμαι πολύ αισιοδοξο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Μόλι χθε στου Times λεγόταν, υπήρχαν και άλλε παραποιημένες ειδήσει. Λέγανε οι υπουργοί του Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο και το κόστος ε, του διαζυγίου θα περιοριστεί στα 3 δις. Και δεν θα έχει καμία νομική υποχρέωση το Ηνωμένο Βασίλειο να πληρώνει οικονομικές συνεσφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Brexit. Κύριε Μπαρνιέ, νομίζω ότι με όσα μας είπατε σήμερα θα τα ξαναπείτε και όταν ε, προβλέψετε τι διάφορε καταληκτικέ προθεσμίε. Για να υπάρχει διαφάνεια στην όλη συζήτηση και οι Βρετανοί πολίτε να καταλάβουν τι θα λωστούν όταν γίνεται το Brexit. Uh, next, uh, Michel Schaeffer, Alde. Ο κύριος Σέφερ από την Άλτε, από τις ε, κατοχώρες. Κύριε, Σέφλη. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαγνιέ για την ειλικρίνεια με την οποία εκφράσατε τις απόψεις σας, το εκτιμώ στα Ολλανδικά. Είμαι κοινοτάρχης ε, μιας περιοχής της ε, Ολλανδία και είμαι υπεύθυνο για τα προγράμματα Interreg. Είπατε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο, κάποια τιμωρία, αλλά ότι οι λογαριασμοί πρέπει να κλείσουν. Και αυτό είναι σίγουρο. Έχω το εξή ερώτημα όμως. Δεν, εγκυμον... δεν... Ε, δεν εγκυμονεί ο κίνδυνος να μειωθούν τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα για τα ταμεία συνοχής το οποίο σημαίνει ότι τελικά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και οι διάφοροι οικονομικοί επιχειρηματίε και τα λοιπά φορεί θα λουστούν το κόστο. Ο κύριο Σπυρίδων από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά την ε, αξιόλογη ανάλυση του κυρίου Μπαρνιέ και των συναδέλφων, θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και δεν μπορούμε να απολογίσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες θα είναι αρκετές και ιδίως για τις περιφέρειες που ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Δεν θα επαναλάβω όμως τα όσα υπόθεσαν για να δώσω έμφαση σε αυτό που για μένα αποτελεί προτεραιότητα. Ότι το Brexit δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αιτίε εκείνες που έκαναν τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να ψηφίσουν για την έξοδό τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας έντονος λαϊκισμός και ριζοσπαστισμός, ο οποίος σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα με το μεταναστευτικό πρόβλημα έχει δημιουργήσει έναν ιδιότυπο εθνικισμό που είναι τελείω διαφορετικό από τον πατριωτισμό. Τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν να έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει να πάμε γρήγορα και σταθερά ένα βήμα μπροστά. Να νιώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά του, Να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα για περισσότερο συνοχή και να αποκτήσουμε τέλου κοινέ πολιτικέ ενεργοποιώντας επιτέλους την πολιτική ενοποίησή μας με κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική για την άμυνα και βέβαια όσο είναι δυνατόν κοινή οικονομική πολιτική. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αγοραστός παρακαλώ. From Thessaloniki, Greece. Από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να την αγνοήσει κανείς τα πράγματα πρέπει να κυλήσουν με μεγάλη ταχύτητα. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις και κυλάει ο χρόνος, τόσο ο ευρωσκεπτικισμός θα ανδρώνεται. Το μήνυμα το δίνει ο Περικλής στον επιτάφιο. Ο κόσμος κλαίει και οδύρεται για αυτό που είχε και έχασε, όχι για αυτό που δεν απέκτησε ποτέ. Συνεπώς οι επιλογές πρέπει να έχουν και άμεσες συνέπειες Διαφορετικά η Ευρώπη κινδυνεύει, διότι η συστηματική υποκρισία τόσων ετών που, έχουν δημιουργήσει οι ευρωσκεπτικιστές είναι χειρότερο από το λαϊκισμό. Γι' αυτό πιστεύω, για να μην μπει η ιδέα της Ευρώπης το πιο φιλόδοξο έργο πολιτικής τέχνης, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να βρει τη θέση του στο Μουσείο της Ιστορίας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να οργανωθούμε σωστά προς όφελον των λαών μας και της πραγματικής ιδέας της Ευρώπης. Γιατί έχει ανάγκη η Ευρώπη, την ενωμένη πραγματικά Ευρώπη, η οποία να είναι αλληλέγγυα, με σεβασμό σε κάθε Ευρωπαία και σε κάθε Ευρωπαίο και ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. And then... Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εκφράσω την άποψη της Ανδαλουσίας που είναι ε, στα άκρα νότια ε, της Ευρώπης ε, και είναι και μια πολύ εργατική περιοχή. Είμαστε ειλικρινεί, στήμοι, υπεύθυνοι και χρησιμοποιούμε όλους μας τους πόρους για να βελτιώσουμε την ποιότητα της των πολιτών μας. Πέραν αυτών, θέλω να ζητήσω τον κύριο Μπαρνιέ να λάβει υπόψη το γεγονό ότι υπάρχει και ένα άλλο χερσαίο σύνορο, δηλαδή το έδαφος του Γιβραλτάρ με την Ισπανική επικράτη της Ανδαλουσίας και το σύνορο αυτό διέρχονται σχεδόν 10.000 ε, ε, εργαζόμενοι από την Ανδαλουσία καθημερινά και υπάρχει μεγάλη ε, σχέση μεταξύ Γιβραλτάρ και της περιοχής της Ανδαλουσίας που είναι όμορη με, με, την, με το Γιβραλτάρ. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το ότι οι επιπτώσεις του Brexit θα είναι πάρα πολύ σημαντικές σε μια περιοχή που τιμωρείται ήδη σκληρά από την κρίση και από την ανεργία. Ευχαριστώ, Άλαν Χάτσισον. Κύριε Μπαρνιέ, λέγομαι Άλαν Χάτσισον. Είμαι όμως βέλγος από τις Βρυξέλλες ε, και πραγματικά επειδή ε, είμαι ένας ε, πιστός Ευρωπαίος αυτά τα οποία συμβαίνουν με συγκινούν ιδιαίτερα Ελπίζω αυτά που είπατε να γίνουν πράξη μέχρι το τέλος της όλης διαδικασίας, γιατί είναι πολλές προκλήσεις σε μία λεπτομέρεια. Μπορεί να σας φαίνεται και ανέκδοτο. Είμαι υπεύθυνο ε, για τις σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες. Μην ξεχάσετε τους χιλιάδες ε, υπαλλήλου ε, Βρετανούς υπαλλήλου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τις οικογένειές τους, που έχουν πανικοβληθεί, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί. Και μάλιστα πολλές εκατοντάδες ζήτησαν το βελγική υπηκότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βέλγους υπηκός όλους αυτούς βέβαια τους υπαλλήλους. Απλά ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα που για αυτούς τους ανθρώπους είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Thank you. And now our last speaker. Ευχαριστώ και το τελευταίος μας ομιλητής, ένας από τους δημάρχους μας και μετά ο κύριος Μπαρνιέ θα αντιδράσει σε όλα αυτά. Ο δικός μας Μπαρνιέ, λοιπόν. Ε, κύριε Μπαρνιέ, κύριε συνονόματα, ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικές οι εκλογές που περιμένουμε μετά από λίγες εβδομάδες στην Γαλλία. Το πρωί ήμουν στο Παρίσι, στην ε, ακροασία διαφορετικών υποψηφίων για την πρωτοβουλία των δημάρχων της Γαλλίας και πραγματικά ε, ε, αισθάνθηκα φρίκη που δεν γίνεται καθόλου λόγος για την Ευρώπη. Καθόλου όμως. Και πραγματικά με θλίβει αυτό. Διότι η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που ιδρύσανε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη γίνεται κάτι το τρομακτικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε απόλυτη πυγμή, προ... Επιτροπέ, με την, ε, στη σχέση με την Βρετανική κυβέρνηση, ώστε να φανεί ότι αυτοί οι μαθητευόμενοι μάγοι δεν θα τα πάνε καλά στο δρόμο που επιλέξανε. Ευχαριστούμε. Ξέρω ότι ακούσατε πολλά ερωτήσεις, σχόλια. Προσπαθήστε, αν μπορείτε, έστω και τηλεγραφικά, να τα καλύψετε. Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να χαιρετήσω τον κύριο Στόκ που είναι κρυμμένος τον κύριο Φερχόφστακ που είναι κρυμμένος διότι στην αρχή της ομιλίας μου μίλησα για την αποφασιστικότητα με την οποία θα συνεργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο, κυρίως με τον Πρόεδρο, τον κύριο Τεγιάννη και διάφορους συναδέλφους που θα αναλάβουν τις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Εδώ μιλάμε για το Brexit και την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Σε αυτό το επίπεδο θα ψάξουμε να υπάρξει συμφωνία. Ε, να υπάρξει μια συμφωνία που θα κυρωθεί σε επίπεδο κοινοτικό και ευρωπαϊκό. Από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Βρετανικό, συγγνώμη, Κοινοβούλιο, την Βρετανική Βουλή. Όπως είπα προηγουμένως, οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία που θα πλαισιώσει και θα διαμορφώσει τη μελλοντική μας σχέση, τη νέα εταιρική σχέση με τον Αμένο Βασίλειο, αυτή θα είναι ή θα ήταν μια μεικτή συμφωνία και θα χρειαστεί την κύρωση των 27 Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο Μάικλ μέφι ανέφερε προφανώς ένα θέμα που είναι καυτό για τον ίδιο, ε, όπως και ο συνάδελφος από την Ιρλανδία. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Θα, είμαι, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις συνέπειες της Βετανικής απόφασης να αποχωρήσει από την Ένωση. Να αποχωρήσει και από την Τελωνιακή Ένωση. Και οι συνέπειες θα έχουν αντίκτυπο και στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα και την ενιαία αγορά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, κύριε Μέρφη, κύριε Σάμψον, για να μην ξαναέχουμε σκληρά, για να το πω έτσι, σύνορα. Ξέρω τι ευαισθησίε έχετε και ξέρω και πόσο έθραυστε είναι όλε οι προσπάθειε που έχουν γίνει ω τώρα για την ειρήνη στην Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία. Ξέρετε ότι όταν ήμουν επίτροπος ε, από το 1999 στο 2004 για την περιφερειακή πολιτική, είχα κάνει μια από τις πρώτες μου επισκέψεις ακριβώς εκεί, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και κάτι που δεν ξέχασα ποτέ ήταν η συνάντησή μου την ίδια μέρα, σε δύο διαφορετικά όμως σημεία, με δύο ε, νικητές του βραβείου Νόμπελ, τον κύριο Τράμπελ και τον κύριο Χιούμ οι οποίοι τότε, ε, ο οποίο τότε μάλιστα ήταν και μέλος του Κοινοβουλίου. Και μου είπαν και δύο το ίδιο. Μετά από τα τραγικά γεγονότα που έχουν βιώσει, ότι έχουμε έρθει εδώ γύρω από το ίδιο τραπέζι. Όχι χάρη στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή το Μπέλφαστ και την παρέμβασή τους, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε ως εδώ με το πρόγραμμα Peace, Ειρήνη, ε, και αυτόν τον διάλογο τον υποθάλψαμε, τον στηρίξαμε και είμαι βέβαιος για τον ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, στη Βόρεια Ιρλανδία. Ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Βεβαίω, ε, υπολογίζω στον Ηνωμένο Βασίλειο, το είπα και προηγουμένω, ζυγίζοντα τα λόγια μου, ότι είναι εγγυητή ε, της συμφωνίας ε, της, ε, με παρασκευής, της Μεγάλης Παρασκευής του Ηνωμένων Βασίλειων. Και είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε και εκεί τις κατάλληλες λύσεις. Το λέω βεβαιώνοντας την προσωπική μου ευαισθησία, καθώς και αυτή των συνεργατών μου, για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας εκεί. Για τον κύριο Χάντ έθεψε πολλά σημεία. Είπατε θα είναι σκληρέ διαπραγματεύσει. Εγώ είπα δυσχερεί. Έκτακτε. Ελπίζω θα παραμείνουν έκτακτου χαρακτήρα. Ε, Είπατε να μην επικεντρωθούμε μόνο στο εμπόριο και την οικονομία. Εγώ μίλησα και για πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Θα μου το αναγνωρίσετε αυτό. Είπα citizens first, οι πολίτε πρώτοι. Είπα κι άλλα. Είπα για την κοινότητα αξιών. Τα κοινά συμφέροντα που έχουμε ε, στο Ευενικέ ε, μαζί με τον Ηνωμένο Βασίλειο, ασχέτω Brexit. Μίλησα για τα περιβαλλοντικά, τα δημοσιονομικά και τα φορολογικά την ε, άρνηση που θα έχουμε να υποβαθμιστούν ε, όλα αυτά τα δικαιώματα στι διαπραγματεύσει. Βεβαίω υπάρχει και οικονομική συνιστόσα, υπάρχουν πολλέ νομοθετικέ και νομικέ παράμετροι, αλλά μην ξεχνάμε την αβεβαιότητα ε, που έχει περιβάλλει τους άνδρες και τις γυναίκες της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την απόφαση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, μιλήσατε για τη δυνατότητα ανάστρεψη αυτής της ε, δικασία. Ε, κοιτάξτε, κύριε Χάντσα, να σας πω ότι η απόφαση αποχώρησης από την Ένωση και η κοινοποίηση αυτή τη απόφαση είναι μονομερής. Και μονομερός ε, θα εκφραστεί και στην επιστολή που αναμένουμε στις 29 Μαρτίου από την Τερέζα Μέη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η κοινοποίηση αυτή ε, γίνει, ε, λάβει χώρα, δεν είναι πλέον μονομερή, είναι πολυμερή και απαιτεί την ομοφωνία των 27 για να εγκριθεί. 27 συνενός. Κύριε Σόμε, αναφερθήκατε στα δικαιώματα των πολιτών. Το δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη. Το είπα και προηγουμένω. Οι πρωτοβουλίε των πολιτών οι πρωτοβουλίε των πολιτών που έχουν καταγραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζητούν δημιουργικέ λύσει να βρεθούν. Και αυτό προσπαθούμε και εμεί να είμαστε δημιουργικοί και φάνταστοι σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Θα βασιστούμε και στο δίκαιο βεβαίω. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε ε, στην ε, πολύ στενή αυτή εξέβρεση μικρών κρίκων και λεπτομεριών νομοθετικών σχέσεων. Τα ε, εμπλέξαμε όλα αυτά μαζί, από κοινού θα τα απεμπλέξουμε. Εδώ πέρα ε, δεν μιλώ μόνο ε, για μας, αλλά και για τους ευρωπαίους πολιτικούς. εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε να μην γίνεται τίποτα ε, δεν μιλάμε για κανένα μικρό συμβάν. Μιλάμε για μια κατάσταση σοβαρή, έκτακτη. Βεβαίω θα υπάρξουν συνέπειες και τι ανέφερα και προηγουμένω. Ε, κύριε Σόμερ, αναφέρατε τον προπολογισμό. Όπω και ο κύριο Κορδέρο προηγουμένω. στην ε, δημοσιονομική προοπτική που μας αφορά ε, έχοντας ασχοληθεί με διαφορετικές πολιτικές και ιδίως αυτή τη συνοχής. Έχουμε μια προοπτική επταετίας. Το Ενωμένο Βασίλειο έχει συμμετοχή 14% στο σύνολο αυτών των προπολογισμών. 14%. Το είπα προηγουμένω ε, με απόλυτη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει ένα λογαριασμό ακόμα που ξέρουμε το τελικό του, τον τελικό του αριθμό. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για να δούμε πώ θα διαμορφωθεί το τελικό άθροισμα. Και το γεγονό ότι θα δείξουμε υπευθυνότητα, ότι θα αναλάβουμε τι δεσμεύσει και τι ευθύνε μα, είναι ε, ξεκάθαρο. Και φέτο θα εξασφαλίσουμε την εξακολούθηση των χρηματοδοτήσεων και τη ε, στήριξη όλων των προγραμμάτων σε όλε τι ευρωπαϊκέ περιοχέ και περιφέρειε. Αναφερθήκατε στη σκοτία, κύριε Χάναν. Να θυμίσω με απόλυτη σαφήνεια ότι, κύριε Λουκάνεν, θα του ακούσω όλου. Όλου. Η πόρτα μου θα μείνει ανοιχτή. Άρα θα διαπραγματευτώ μόνον με την κυβέρνηση του ΕΒ. Αυτά είναι τα κείμενα, αυτά προβλέπουν ως κανόνες. Θα τους ακούσω όλους, αλλά δεν θα παρέμβω στις εσωτερικέ σχέσει. σχέσεις. Δεν είναι ο ρόλος μου στο διαπραγματεύσεις. Δεν θα επηρεάσω τις εσωτερικές και θεσμικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Γόλης, Αναφερθήκατε στις δημόσιες διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Ναι, θεωρώ ότι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, το είπα και εγώ προηγουμένως, θα πρέπει να έχουν συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις. Θα υπάρξει συνεργασία. Ελπίζω ότι ε, μόνιμα θα υπάρξουν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΒ Βασιλείου που θα τη θελήσουν αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό και εντόπισα και ανέφερα ξεκάθαρα εδώ ε, τις τι προποθέσει για να πετύχουν όλα αυτά. Και ευχαριστώ που τις ακούσατε με προσοχή. Δεν το είπα για να δημιουργήσω προβλήματα και να πω ότι θα βρούμε εμπόδια. Όχι, για να καταλήξουμε σε συμφωνία τα είπα. Και εφόσον συμβεί αυτό, θα υπάρξει πεδίο συνεργασίας για το μέλλον. Κυρίως σε συνεργασία με τις ε, τοπικές αρχές. Από την άλλη μεριά της μάχης. Κύριε Χάτς, καταλαβαίνω την δική σας οπτική γωνία αλλά το επαναλαμβάνω και σε εσά. Θα υπάρξουν αλλαγέ. Τι να σα πω, το αντίθετο, ότι όλα θα είναι όπω πριν. Θα έλεγα ψέματα. Και μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Θα υπάρξουν αλλαγέ. Το business as usual δεν μπορεί να υπάρξει πια. Κύριε Χάτζ, να είστε βέβαιος ότι σε αυτές τις αντικειμενικά, χωρίς προκαταλήψεις, θα χρειαστεί να κάτσουμε και να δούμε και να μελετήσουμε όλα τα βήματα πρόοδου που έχουμε κάνει από κοινού ως τώρα. Και χωρί να ξεχνάμε, και το λέω στο συνονόματό μου, τον Ζανφρανσουά Φρανσουά Μπαρνιέ, τον οποίο χαιρετώ. Ε, το πνεύμα των συζητήσεων σε πολλές από τις χώρες μας, τη δική μου για παράδειγμα συγκεκριμένα, επίτηδες παραλείπει τα βήματα πρόοδου της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για τις περιαγωγές, είτε πρόκειται για τις διευκολύνσεις της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να τα υπενθυμίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Διότι βγαίνοντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ενιαία αγορά, από την Τελωνιακή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο αυτοβούλος επιλέγει να εγκαταλείψει κάποια από αυτά τα στάδια πρόοδου. Πρέπει λοιπόν να γίνει και μια προσπάθεια ε, εκπαιδευτική, παιδαγωγικού χαρακτήρα καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων χωρίς βεβαίως να το κάνουμε και επώδυνο. Κύριε Κορντέρο, είμαι και ανέκαθεν παρακολουθήσω με προσοχή την τύχη της Ένωσης των εξόχων Απόκεντρων Περιοχών Πιστεύω ότι είναι ε, τυχερή η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τέτοιε περιοχέ. Περιοχέ που τη επιτρέπουν να έχει ένα πάτημα ε, για τα πόδια τη και να πάει πολύ μακρύτερα σε ωκεανού που δεν έχουν καμία σχέση με τα σύνορά μα. Εκεί βρίσκεται η αξία και η επιρροή σα και ξέρω ότι σημασία έχουν αυτέ οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Όμω, μια απάντηση στην ερώτησή σα. Εν μέρη, εξαρτάται από την, από την επιτυχία αυτών των διαμονατεύσεων από το αν θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τις τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό είναι και το πρόγραμμα που έχουμε στις διαμονατεύσεις μας με το, με την Ευρωπαϊκή, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως, είναι άλλη ιστορία, όπως είπα και στην κυρία Χίλ. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές μετά. Είναι άλλη ιστορία και δεν είναι δικός μου ο ρόλος. Ακόμη και αν με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν είναι κάτι που μπορώ να το πω ε, εγώ τώρα. Είναι πάντοτε πολύ δύσκολο να διαμορφώσει κανεί 7 ετή δημοσιονομικέ προοπτικέ. Προφανώ από το 2020 θα υπάρχει μια επιπλέον δυσκολία. Θα είμαστε πλέον 27. Θα έχουμε 10 δι, κατά μέσο όρο, 10 δι λιγότερα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Σε ό,τι μου αφορά, προσωπικά παραμένω από απόλυτα ε, πιστός στην πολιτική της συνοχής, όπως ήταν και πρόεδρος Ντελόρ, γιατί ακριβώς αυτή επιτρέπει να καλυφθούν οι τοπικές αποκλήσεις και ανισότητες. Και τώρα τηλεγραφικά στους υπόλοιπους ε, μιλητές. Όταν ο κ. Λάμες ανέφερε την χώρα του, Βεβαίω κάποιε χώρε θα πληγούν περισσότερο από άλλε. Υπάρχουν ε, εμπορικέ σχέσει διαφορετική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και 27 χωρών. Το Βέλγιο, η Ιρλανδία οι κάτω χώρε θα πληγούν περισσότερο. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου στι προσπάθειε και τι διαπραγματεύσει μα. Επίση, να θυμίσω ότι συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Συμβουλίου των 27 χωρών με τον Κέφερ Χόφστατ και άλλου εκπροσώπου του Κοινοβουλίου για να δούμε τι συνέπειε του Brexit στα τελωνία. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα συμβεί με την Τελωνιακή Ένωση. Όταν μια χώρα βγαίνει, τα εμπορεύματα, τα ζώα, τα νοπά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται όταν βγαίνουν και όταν μπαίνουν στην Ένωση, όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν από την μία χώρα. Άρα, για πολλές από τις χώρες μας, για τις περισσότερες από τις χώρες μας, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθούν αυτοί οι έλεγχοι. Η κυρία Μπορ ανέφερε τις νέες σχέσεις που θα διαμορφωθούν. Να επαναλάβω κυρίε και κύριοι, ότι ο καλύτερο τρόπο να έχει κανεί σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι μέλο τη. Ο καλύτερο τρόπο να έχει κανεί σχέση μαζί τη είναι ακριβώ να είναι μέλο τη. Και σε δεύτερη φάση, η δεύτερη καλύτερη σχέση θα είναι να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ΕΟΧ όπως η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν ή η Ισλανδία. Έχουμε υποχρεώσεις και έναντι αυτών των χωρών. Νομίζω ότι απήντησα ως προς τον προπολογισμό, προς τον κύριο Σπυρίδωνα και στον κύριο Αγοραστό. Αναφέρατε τον έκτακτο χαρακτήρα αυτών των διαπραγματεύσεων. Ακούς, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, και ο, και ο ένας και ο άλλος αλλά να κάνουμε μια σαφή διάκριση εδώ σε αυτή την ιστορία. Οι συνέπειε του Brexit και εν μέρει αυτό θα πρέπει να καλύψω για διαπραγματευτή σε συνεργασία με τον κύριο Φερχόφστατ και το Συμβούλιο τα διδάγματα του Brexit. Τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από τον Brexit. Τα αναφέρατε κι εσείς. Και νομίζω ότι τα εκφράζουν οι Βρετανοί πολίτες. Κάποιες φορές το λαϊκό αίσθημα πρέπει να γίνεται σεβαστό, να ακούγεται. Τα λέει και η Λευκή βιβλό του Ζάμπιν Κλοντ Κλομπ-Γιούνκερ. Δικαιολογεί την ανάγκη μετά τη Ρώμη σε 48 ώρε να προβλέψουμε μια νέα ατζέντα για την Ευρώπη που να ενδιαφέρει του πολίτε, να του προσελκύει, να δείξουμε την προσταθεμένη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα σύνορα, τι κοινέ επενδύσει, την έρευνα, την άμυνα, την ασφάλεια, την ψηφιακή ένωση. Αυτοί είναι οι λόγοι ε, που με κάνουν ε, να είμαι ακόμα υπέρμαχος μιας ευρωπαϊκής ατζέντα. Για το Γιβραλτάρ. Θα είμαι σαφής. Το Γιβραλτάρ θα βγει από την Ένωση μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Χάτινσον, είπατε ότι σας συγκινούν βαθιά όσα συμβαίνουν. Ε, και εμείς συγκλονιζόμαστε και ανησυχούμε για τους υπαλλήλους, κύριε Χάτσινσον, θα θυμίσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ. ευθύς εξ αρχή, όταν ε, είχαμε το αποτέλεσμα του ψηφίσματος για τον Brexit. Πρέπει να προστατευτούν οι ε, ε, υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όποια και αν είναι η εθνικότητά του, γιατί είναι Ευρωπαίοι υπάλληλοι. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα εδώ να επιβεβαιώνω ξεχωριστά όσα είπε ο πρόεδρο Γιούνκερ. Αυτό αφορά τι σχέσει των θεσμικών οργάνων Κάποιος μου κόψε το μικρόφωνο, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, την προθυμία σας και τη συνεργασία στην οποία ευελπιστώ. Thank right, uh, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να καλωσορίσω τους ευρωβουλευτές ε, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη συζήτησή μας. Ε, δύο λόγια μόνο. Είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική εν ώψη και της 60η απαιτία από την υπογραφή τη συνθήκη τη Ρώμη. Ε, και πραγματικά είμαι υπερήφανο για τα βασικά επιτεύγματα, ειρήνη, ευημερία, κοινωνική συνοχή Υπήρξαν πολλές κρίσεις ε, τα πρόσφατα έτη. Αυτό λοιπόν ε, που παρατηρούμε είναι μείωση της εμπιστοσύνη και των πολιτών στην Ένωση. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αυτό. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους και έχει αλλάξει η αντίληψη που είχαν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω θέλω να πω ότι στην δίκη του Μάστριχτ αυτό που ήθελε ήταν να κλείσει το χάσμα μεταξύ Βρυξελών και Ευρωπαίων πολιτών. δημιούργησε την ε, αρχή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης με το ίδιο πνεύμα ε, συγκροτήθηκε για να γίνει ακουστή η φωνή ε, των τοπικών και περιφερειακών αναγκών. Βέβαια το κατά πόσον έχουμε μέσα και εξουσίες για την πρόθεση, την εκπλήρωση των αρχικών προθέσεων των ιδρυτών πατέρων δεν θέλω να επεκταθώ. Αυτό που έχει σημασία πάντως για τους πολίτες ε, είναι όχι η ε, διελκυστίνδα ό,τι αφορά τι εξουσίε ή αλλαγέ των συνθήκων. Ε, θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε τη λευκή βίβλο για το μέλλον τη Ευρώπη, ε, που ελπίζουμε να βοηθήσει την χάραξη του μέλλοντο τη Ευρώπη. Αυτή είναι μια μείζον συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει και θα την κάνουμε και εμεί εδώ. Θέλω να τονίσω ιδίω ένα στοιχείο που είναι η αμφισβήτηση της συνοχής και της προσθέμενης αξίας. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο μονοπάτι. 270 περιφέρειες έχουμε. 60.000 ε, δήμους ε, και μάλλον κοινότητες ε, έχουμε εδώ και εμεί θέλουμε να παραμείνει σε ισχύ αυτή η θεμελιώδης αξία. Οι δήμοι και οι κοινότητες είναι η ατμομηχανή για το ευρωπαϊκό μέλλον. Και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Τώρα, να επανέλθω στη δική μας συνεισφορά στην όλη συζήτηση και ειδικά θέλω να αναφερθώ σε μία πρωτοβουλία που αναλάβαμε από κάτω προς τα πάνω και λέγεται προβληματισμός για την Ευρώπη, Reflecting on Europe. Οι πολίτες μπορούν να μας παρουσιάσουν τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ένωσης. Αυτό το σημερινό γεγονός λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτό το λόγο. Πρέπει να πω ότι συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ντόναλτ Τούσκ. Σας έχουμε διανύμει ε, αυτό το πλαίσιο, αυτό το φυλάδιο. Για τη σχετική πολιτική, ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σε δύο ημέρες από τώρα και εγώ θα συμμετάσχω στον επίσημο ερτασμό της 60ης ε, ε, επαιτίου της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης και είμαι πεπισμένος ότι το κείμενο αυτό όπως και 10 χρόνια πριν με τη διακήρυξη του Βερολίνου, έτσι και μεθαύριο θα αντικατοπτρίζει ότι είμαστε μια κοινότητα αξιών που βασίζεται στη διαφορετικότητα, ε, την ποικιλομορφία και βασίζεται ε, στο δυναμικό των πολιτών, στη βάση. Εκ μέρου ε, της Επιτροπής των Περιφερειών είμαστε έτοιμοι να σας προτείνουμε και εμεί τι δικέ μα Γι' αυτό και η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στον Ευρωβουλευτή κύριο Γκί Φερχόστατ ε, που είναι και εισηγητή για τι δυνητικέ εξελίξει και τροποποίησεις τρέχουσα θεσμική διάρθρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το εγχείρημα αυτό που ξεκίνησε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται σε τρει εκθέσει. Πρώτα απ' όλα, την έκθεση του κύριου Μπροκ ε, και της κυρίας Μπρέσο και του Γιώ Λάινεν ε, την έκθεση για ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις δυνάμει τη συνθήκη τη Λισαβόνας και υπάρχει και δική μου έκθεση για το τι απαιτείται εκτός των συνθήκων, των υφιστάμενων συνθήκων. Υπάρχει και μια τρίτη έκθεση. Έκθεση μπερέ Μπέγκε, η οποία αφορά τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της Ευρώπης για τη δημοσιονομική ικανότητα μεταξύ άλλων της Ευρωζώνης. Επομένως, δεν έχουμε μία έκθεση εκπονήσει. Έχουμε τρει πολύ συνεκτικέ μεταξύ του εκθέσει και νομίζω ότι πρέπει να τι αναγνώσετε από κοινού τι τρει αυτέ εκθέσει για να σχηματίσετε με γενική εικόνα για τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για ποιου λόγου θα κάνουμε, κάνουμε αυτέ τι προτάσει, που είναι ευνόητοι νομίζω. Ζούμε σε δύσκολου καιρού στην Ευρώπη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολλαπλή κρίση που έχει να κάνει με του πρόσφυγε, του μετανάστε, τις ε, συνέπειες της χρηματοοικονομική κρίσης που δεν την έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει πλήρως. Μεταξύ άλλων, αυτές είναι οι προκλήσεις. Τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Αυτό προσπαθούμε να απαντήσουμε και πώ θα τι αντιμετωπίσουμε βέβαια καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι εντό και εκτός ε, αυτό που νιώθουν ε, είναι το ίδιο λίγο πολύ, ότι δηλαδή η Ευρώπη δρά αργά και κάνει πολύ λίγα. Και αυτό και ε, ήταν πραγματικότητα και στη διάρκεια της κρίσης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αντέδρασαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Πώς αντέδρασαν άμεσα ξεκίνησαν το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 400 δις δολάρια. Μετά ακολούθησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα τεράστιων διαστάσεων, πάνω από 900 δις δολάρια, σε διάρκεια 10 ετών, σε ορίζοντα 10 ετών. Και είχαν και το λεγόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ομοσπονδικής Τράπεζας, 1,23 δολάρια. Και όλα αυτά, αυτά τα τρία ε, βλήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης ε, τα εκτόξευσαν ε, μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Και τότε ήταν οι Ρεπουμπλικανοί που ξεκίνησαν και μετά Ομπάμα με τη δημοκρατική κυβέρνηση. Για συγκρίνετε τώρα τι έκανε η Ευρώπη που αντιμετώπισε την ίδια χρηματοπιστωτική κρίση αλλά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και είμαστε ακόμα μέσα στην κρίση. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις τράπεζες δεν έχουμε ολοκληρώσει καν την Τραπεζική Ένωση που τόσο χρειαζόμαστε. Εξακολουθούμε να συζητούμε το επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο και το οποίο είναι πάρα πολύ μικρότερο σε διαστάσει από το Και κάναμε με την ποσοτική χαλάρωση, αλλά πολύ αργότερα και ήταν αμυντική απόπειρα. Η προσπάθειά μα ήταν να αποφύγουμε τον αποπληθωρισμό και όχι να ενθαρρύνουμε τι οικονομίε. Επομένω, αυτό το οποίο μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ερώτημα που θέτουμε είναι πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να αντέδρασαν ανάμεσα και εμείς να έχουμε τόσο μεγάλη δυσκολία. Και νομίζουμε ότι αυτό οφείλεται στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι κατάλληλο προς το σκοπό αυτό και δεν είναι και στο ύψος των περιστάσεων για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμιστεί το στομότερο δυνατό. Και αυτό που κάνουμε στι τρει εκθέσει μα είναι να εξετάσουμε τι πρέπει να γίνει εντό των συνθήκων, εκτό των συνθήκων και ειδικά στην Ευρωζώνη. Τι νέου είδου διακυβέρνηση χρειαζόμαστε συγκεκριμένα. Δεν αρκεί το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη και κάποιοι κανόνε. Χρειάζεται ταμεία, δημοσιονομική ικανότητα Υπουργός Οικονομικών της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Και η σύγκληση, ο κώδικα σύγκληση. Τι θεσμικέ επίση αλλαγέ πρέπει να γίνουν στη δικασία λήψη αποφάσεων εδώ στην Ευρώπη. Ίσως χρειάζεται μια μικρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποτελεί μια πραγματική Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και δεν θα εκπροσωπεί πλέον 28, γιατί 28 είναι οι χώρες, έτσι. Αύριο θα είναι 27. Και μεθαύριο μπορεί να ξανά είναι 28. Όπως γνωρίζουμε όλοι. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα με δύο φορείς ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσωπεί τους πολίτες και το άλλο Συμβούλιο ε, Κρατών που εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπω συμβαίνει σε μια ευρύθμιση λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Αυτό που χρειάζεται επίση είναι ένας προπολογισμό που θα βασίζεται περισσότερο σε αυτό που εμεί λέμε ήδη οι πόροι και εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά από την ομάδα Μοντι, όπω την αποκαλούμε. Και τα τρία θεσμικά όργανα, άρα και το Συμβούλιο μαζί, δημοσιοποιήσαμε μια έκθεση η οποία αναφέρει το είδος της νέας χρηματοδότησης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είμαστε σε θέση στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και πάνω από όλα αυτά, αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι εκθέσεις είναι να διερευνήσουμε νέου τομεί. Να δούμε πού πρέπει να είμαστε παρόντε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη, αμυντική ένωση. Ή, ένα άλλο παράδειγμα, μεταναστευτική πολιτική βασισμένη σε πραγματική ε, δυνατότητα και ικανότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή Συνοριοφυλακή ή δυνατότητα στο μέλλον να δημιουργήσουμε ε, ικανότητα έρευνας ε, ή υπηρεσίας πληροφοριών. Γιατί το βλέπουμε σήμερα και το είδαμε και κατά το παρελθόν ότι ο συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών είναι ελλειπή, είναι ανεπαρκή υπάρχουν συνέχεια κενά, υπάρχουν πάντα παραθυράκια. Για να το πω αλλιώ οι τρομοκράτε δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά η αστυνομία και η συνοριοφυλακή εξακολουθεί να γνωρίζει σύνορα. Δεν είμαστε σε πλεονεκτική θέση απέναντι στους τρομοκράτε. Όλα αυτά πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητο και έπειτα την έκθεσή μα να ολοκληρώνουμε με μία σύσταση και προ τα τρία θεσμικά όργανα. Άρα και, ε, μάλλον προ όλα τα θεσμικά όργανα, άρα και σε εσά ότι θέλουμε να γίνει ένα θεσμικό προβληματισμό παραλλήλου με τον Brexit. Για τον Brexit σίγουρα ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαπραγματεύσει και η συζήτηση. Γιατί η αποχώρηση μια χώρα από την Ένωση δεν μπορεί να είναι εύκολη. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να κάνουμε και μια πιο επιθετική, ε, να ασκήσουμε μια επιθετική δράση και να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα θεμέλια της έκθεσης Μόντι. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ένα διοργανικό προβληματισμό, θεσμικό προβληματισμό αρχίζοντας με τα τρία βασικά θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν, αλλά φυσικά και εσείς ε, και η Περιοφέρειες, η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να συμμετέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Let's give them uh, now the next... Uh, να δώσω τώρα το λόγο στον Έλμαρ Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν με επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά. Έχουμε τις δύο εκθέσεις που έχουμε προετοιμάσει εμείς ε, με την κυρία, εγώ και η κυρία Μπρέσο έχουμε και την έκθεση του κ. Φερχόφστατ, η οποία έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ πιο πολύ ασχολείται με ε, τις αρχές και σίγουρα ο ίδιος μπορεί να σας πει πολύ περισσότερα ε, για αυτό το θέμα. Και η δική μας ε, έκθεση ασχολείται με τις ανάγκες τροποποίησης των συνθήκων. Κάτι που δεν θα γίνει όμως ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Είναι μια πιο, μακρά, ε, πιο ε, μακροσκελής διαδικασία. Θα έχουμε θεσμική συνέλευση, θα έχουμε την ε, διαδικασία κύρωσης από τα κοινοβούλια και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για τη σημερινή ένωση και να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε με τα τρέχοντα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή με την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για να μην έχουμε καμία ε, αρνητική επίπτωση. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει, μας δίνει απίστευτα πολλές δυνατότητες, αν υπάρχει βέβαια βούληση για να εξαντλήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχει επίσης το θέμα της διαφάνειας ε, και των αρμοδιοτήτων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων ως ελεγκτικών αρχών και ο ρόλος βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Και δεν θα πρέπει επίσης να υπάρξει σύγχυση αρμοδιοτήτων. Έχουμε και ένα πρόβλημα όμως, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ των συμπολιτών μας Έχουμε ουσιαστικά δύο βουλές, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχουμε το Συμβούλιο και έχουμε και το Κοινοβούλιο. Έχουμε ένα ε, διτό σύστημα, κοινοβουλευτικό σύστημα. Αλλά σίγουρα ε, η Επιτροπή των ε, Περιφερειών κάποιες φορές δεν εμφανίζεται πάρα πολύ στο προσκήνιο, ιδίως αν υπάρχει κάτι που δεν είναι δημοφιλές το Συμβούλιο είναι το, σώμα που θα πρέπει να λαμβάνει τις νομοθετικές αποφάσεις. Θα πρέπει εσείς να ε, μεταφέρετε τις ε, αιτιολογήσεις ε, και να εξηγείτε γιατί λήφθησαν οι αποφάσεις αυτές. Έχουμε ένα πρόβλημα με την αξιοπιστία. Οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη γιατί δεν ξέρουν ποιος, γιατί πράγμα είναι υπεύθυνος. Υπάρχει το θέμα της διαφάνειας που πρέπει να το λύσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει αποδοχή των πολιτικών διαδικασιών, το να ξέρουμε ποιος πότε πού κάνει τι. Και όχι όταν βρέχει να τα ρίχνουμε στις Βρυξέλλες και όταν έχει ήλιο να λέμε «Α, αυτό είναι χαριστερό με το Βερολίνο» κτλ. Αυτό δεν ε, μπορεί να επιτραπεί. Επίσης, ε, τα είπε και ο συνάδελφος, έχουμε το θέμα της μετανάστευσης. Με τη σημερινή συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την συνοριοφυλακή και αυτό κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μισό χρόνο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη πριν από 15 χρόνια το είχε προτείνει. Αλλά περίφθη από τους υπουργούς εσωτερικών των εθνικών κυβερνήσεων. Για το κατά πόσον αυτό είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα ή όχι, Τώρα λένε αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι. Μακάρι να είχαμε αυτή τη φυλακή από το 2015. Ο Επίτροπος Φρατίνη επίσης. Ιταλός και τέος υπουργό εξωτερικών. Είχε πει ότι θα έπρεπε ε, τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων που είναι και υποψήφια για την Ένωση να είναι ασφαλείς χώρες προέλευσης. Και πρέπει να πω ότι το 2015 από τα ρεύματα των μεταναστών το 40% ήταν από αυτές τις χώρες των βυτικών Βαλκανίων, Αλβανία κτλ. Πώς θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη αποδοχή από τους πολίτες και πώς θα μειώσουμε την ε, ε, δημαγωγία και το λαϊκισμό. έχουμε κάποια όργανα και κάποιες αμοδιότητες και δυνατότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και υπάρχει και το θέμα τη τρομοκρατία. Έχουμε την όλα που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη τρομοκρατία. Όμω, τα περισσότερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν ε, θέλουν να, να κάνουν αυτό που πρέπει. Πώς θα καταπολεμηθεί η διεθνής ε, τρομοκρατία. Πώς θα ευθυγραμμιστούν, δεν θα πρέπει να αυτογραμμιστούν οι προσπάθειες όλων των κρατών Δεν θα πρέπει να μεταλλευτούμε τις αρμοδιότητες που έχουμε. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλούς άλλους τομείς. Για την Οικονομική Νοτιοτική Ένωση θα μπορούσα να μιλήσω, που έχουμε θέματα, ποιες είναι οι συνέπειες επίσης της παγκοσμιοποίησης στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, αυτή η ανισορροπία πώς μπορεί να περιοριστεί η δημοσιονομική ικανότητα, είπε ο Γκίφερ ε, Αυτό μπορεί επίσης δυνάμει της σημερινής συνθήκης να επιτευχθεί. Δεν ξέρω αν πω ε, αυτό και θα γίνω δημοφιλής ότι είμαι, επειδή είμαι Γερμανός, ότι όταν υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα ε, σε μια χώρα ουσιαστικά πρέπει να ε, υποφελούνται από αυτό και οι υπόλοιποι, γιατί αλλιώς είναι χαμένος αυτός που το έχει αυτό Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να γίνει χειρότερη κατάσταση των ισχυρών, απλά πρέπει να ισχυροποιηθούν οι άλλοι που δεν είναι τόσο ισχυροί. Και αυτό μπορεί να το κάνει κανείς ε, μεταξύ άλλων, όχι με λόγια, αλλά με τήρηση των κανόνων. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως και τη φιλοσοφία μας. Επίσης πρέπει να καταστήσουμε φες ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τις εξουσίες μας τι εμπορικές. Όταν λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει να κάνει διμερείς διαπραγματεύσεις με τα ευρωπαϊκά κράτη για να εξασφαλίσει περισσότερο κέρδος και οφέλο για τις ΗΠΑ, αντίστροφα θα πρέπει εμεί να απαντήσουμε όχι, θα είμαστε όλοι ενωμένοι και θα διαπραγματευόμαστε μαζί. Γιατί ό,τι ισχύει για όλου θα ισχύει για τον έναν. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να καθιστούμε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μελών της. Είναι ένα όλον μεγαλύτερο από το άθροισμα των μελών της. Το ίδιο και για την πολιτική, την αμυντική, όπου διατυπώνονται σιγά σιγά προτάσεις. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την αμυντική πολιτική. 200 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέτουν από τους προϋπολογισμούς τους τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνά τους, διπλάσιο από τη Ρωσία. Περισσότερους στρατιώτες έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και καθένας κάνει μόνος του ό,τι έχει να κάνει. 38 διαφορετικούς τύπους μεταγωγικών οχημάτων, τεθωρακισμένων, έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάνω από 80% πρόσθετο κόστος. Εάν δώσουμε 2% από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την κοινή άμυνα, τότε θα έχουμε μια ορχήστρα η οποία θα λειτουργεί και θα φέρνει αποτελέσματα πολύ καλύτερα. Και βεβαίως αντίστοιχα για την έρευνα, για την ανάπτυξη, για τις προμήθειες, εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κερδίσουμε, να κερδίσουμε σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δηλαδή μπορούν να φέρουν τεράστια ε, αποτελέσματα και ως προς την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό όταν κάθε μέλος, η Πολωνοί, η Ρουμάνοι, χώρες της Βαλτικής αντιληφθούν ότι έχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας όσο και τα υπόλοιπα κράτη, τότε θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτή η έννοια της συνεργασίας, των συνεργατικών αποτελεσμάτων, θα είναι το κέρδος μας, να δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και όχι ο καθένας στη γωνιά του. Ίσως υπερβάλλουμε τα λόγια μου, αλλά νομίζω ότι δίνω την εικόνα και θα πρέπει επίσης να πούμε και αυτό αφορά και τα εθνικά αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι μπορούμε έτσι να δώσουμε και σαφή απάντηση έναντι των επιχειρημάτων των λαϊκιστών, οι οποίοι δεν είναι πάντα στα άκρα δεξιά, αλλά και πολύ στα αριστερά της πολιτικής. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν πιστικά επιχειρήματα και απαντήσεις, καθιστώντας σαφές ότι δεν θέλουμε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό το καθιστά πολύ το σαφέ στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε κεντρική διακυβέρνηση, δεν θέλουμε κράτος στην τωρινή εξέλιξη που έχουμε και θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ρυθμίζονται καλύτερα αυτά τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν καλύτερα και να φέρουν προσθεμένη αξία. Η χώρα μου που είναι ομοσπονδιακό κράτος το έχει ζήσει αυτό στο παρελθόν και αυτό προτείνουμε περιφέρειες και εθνικό κράτος στην Συνομοσπονδιακή Γερμανία στο παρελθόν και τώρα αυτό σημαίνει περιφέρεια, εθνι, περιφέρειες, εθνικά κράτη και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπαίνει όμως στη θέση του εθνικού κράτους η Ευρώπη. Και ιδιαίτερα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η περιφέρεια να έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Προερχόμενος από ομοσπονδιακό κράτος μπορώ να το πω αυτό πολύ εύκολα. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε τόσο σημαντικά καθήκοντα, η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την παράδοση, αλλά με την επιδίωξη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και έτσι πιστεύω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να είναι πολύ πιο μπορεί να συμμετέχει περισσότερο και να έχει πολύ περισσότερη επιρροή και στη δράση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να καθιστά σαφές το πώς μπορεί να οργανώνεται η δουλειά αυτή καλύτερα στη συμμετοχή της και στη νομοθετική μας δουλειά. Ευχαριστώ. Thank you very, uh, on this... Εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντική η τελευταία σας παρέμβαση. Να ακούσουμε τώρα το γιο Λάινεν. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ στην Επιτροπή των Περιφερειών. και χαίρομαι που βλέπω κάποιους συναδέλφους μου που ήμασταν μαζί ήδη από τη δεκαετία του 90 να είναι ακόμα εδώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι δύο συνάδελφοι για τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τη στοχοθέτηση του Κοινοβουλίου για τον διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως εγώ να μπορώ να σας δείξω μια διαφορετική διάσταση σε σχέση με τη σημερινή μας συζήτηση. Ε, πέραν της ε, θητείας μου στο Κοινοβούλιο, είμαι και μέλος της ε, Κοινωνίας των Πολιτών και είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεθνούς Κινήματος. Ασχολούμαι όλη μου τη ζωή με αυτό. Ήμουνα υπουργό Περιβάλλοντος, ήμουνα στο κίνημα. Μ' αρέσει εμένα η Κοινωνία των Πολιτών. Γιατί νομίζω ότι οι πολιτικοί χρειάζονται και την όθηση από τους πολίτες. Για οποιοδήποτε θέμα είναι αυτό που τους κινητοποιεί έτσι ώστε να μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με τους πολίτες όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα στα θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ε, ο εορτασμός της ε, συνθήκης της ε, Ρώμης είναι μια πολύ σημαντική ε, ευκαιρία για να εορτάσουμε ακριβώ αυτό, το ευρωπαϊκό ε, κίνημα με το, την ομάδα Σπινέλη στο Κοινοβούλιο, με τους Ευρωπαίου Φεντεραλιστέ. Μιλούμε για το March for Europe στις 24 Μαρτίου, όπου θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στη Ρώμη. Πολλές φορές ε, έχω διαδηλώσει για την Ευρώπη στη ζωή μου, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν η τελευταία φορά ήταν στην ε, Νίκαια η τελευταία φορά για την ε, συνθήκη της Νίκαιας και για 20 χρόνια δεν έκανα τίποτα. Τώρα είμαστε στο 2017 και νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα να βγούμε και πάλι στους δρόμους και να παλέψουμε για την Ευρώπη. Γιατί αρκετά πλέον. Αν δείτε τι γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή ιδέα πραγματικά παραβιάζεται από ψέματα, από άσχημη ρητορική, από υπερβολές. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και καταλήγουν οι πολίτες σε λάθος συμπεράσματα και πρέπει να και καταλήγουν τελικά οι πολίτες να στρέφονται στον λαϊκισμό, στον εθνικισμό, να καταρρύψουμε την Ευρώπη, να υψώσουμε τύχη, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ώρα πλέον να πολεμήσουμε για την Ευρώπη. Χρειάζεται αυτός ο αγώνας. Δύο χρόνια πριν ήμουνα στην Ουκρανία και πραγματικά με συγκινεί ακόμα αυτό το γεγονός. Αν δείτε πόσες εκατοντάδες ευρωπαϊκές σημαίες είχαν οι πολίτες στα χέρια τους στις διαδηλώσεις εκείνες. Ένας φιλόσοφος από την ε, Ουκρανία έλεγε ότι κάποια κράτη, σε κάποια κράτη-μέλη καίνε τις ευρωπαϊκές σημαίες. Ε, η γεωργία, ας πούμε, γιατί η Ρωσία μποϊκοτάρει τα γεωργικά προϊόντα, οπότε καίνε τις ευρωπαϊκές ε, σημαίες γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν στη Ρωσία ντομάτες. Ενώ στο Κίεβο πέθανε κόσμος για να ζήσει ακριβώς με δημοκρατία και ελευθερία και με όλα τα δικαιώματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποιοι πεθαίνουν για την Ευρώπη και κάποιοι καίνε την Ευρωπαϊκή σημαία γιατί δεν, ξε, δεν τους αρέσει το τάδε ή το δίνα που γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες και μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπω ότι οι πολίτες ξυπνούν. Ακούσαμε αυτά που λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, ακούμε και τα όσα λέει ο Πούτιν, την προπαγάνδα που υπονομεύει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και είναι ώρα πλέον να αντισταθούμε, να αντιδράσουμε. Και είναι χαρά μου που βλέπω ότι Μία ε, οικογένεια στην Γερμανία ξεκίνησε να διαδηλώνει α, στην, α, στους δρόμους της πόλης. Κάθε Κυριακή υπάρχουν 10 ακόμη πόλεις ε, στις οποίες οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους με τις σημαίες τους, διαδηλώνουν και περιμένουν βεβαίως να δούνε και τι θα γίνει με τις εκλογές που θα έχουμε αυτή τη χρονιά και βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Ο Έλμαρ και ο Γκί ξεκινήσανε μαζί με άλλους μια νέα ε, κυβερνητική οργάνωση στην Civico Europa και παρουσιάσαμε πραγματικά ένα ε, αφήγημα 7 πυλώνων για να δούμε το μέλλον της Ευρώπης. Θα σας αναφέρω εγώ δύο ή τρία στοιχεία του. Καταρχάς δημοκρατία, συμμετοχή και βεβαίως θα πρέπει και οι πόλεις και οι περιφέρειες να έχουν πολύ πιο ισχυρό ρόλο να παίξουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί αυτό καταλαβαίνουν οι πολίτες. Εκεί, ε, εκεί νιώθουν την πολιτική και τη χάραξη πολιτικής πιο κοντά τους. Και γι' αυτό βεβαίως πρέπει να πολεμήσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε προς αυτό να κάνουμε πολλά. Επίσης, για τους πολίτες, εγώ είμαι η εισηγητή ε, τη ε, γνωμοδότηση για την ε, μεταρρύθμιση των ευρωεκλογών. Έχουμε 28 εθνικούς εκλογικούς νόμους με καταλόγους, δεν έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές και οι πολίτες θεωρούν ότι δεν είναι πραγματικό, είναι πλασματικό αυτό που γίνεται. Επίσης, πέραν της δημοκρατίας έχουμε την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. αν δεν γνωρίζουμε η μεν με τους δε, ε, πώς θα ζήσουμε μαζί. Το Εράσμους για όλους ας πούμε. Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλους. Δεν κοστίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Τι είναι ένα δισεκατομμύριο σήμερα για να μπορέσουν ε, και οι μαθητές αλλά και οι εργαζόμενοι να έχουν την ευκαιρία να πάνε κάποιους μήνες το χρόνο σε μια άλλη χώρα και να έχουν μια διαφορετική εμπειρία. Ακόμα και η ιδέα για τους ελέγχους ότι αφορά τον πολιτισμό για τους νέους, ας πούμε έναν, τις επιταγές για τον πολιτισμό όπου μπορεί να πάρει κάποιος χρήματα μέσω των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών. Και βεβαίως δεν μιλώ για την οικονομία ή για τον κοινωνικό πυλώνα, για να αποφύγουμε τους φορολογικούς παραδείσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσφέρουμε ασφάλεια ε, θα κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι ο Γιούνκερ μιλώντας ε, στην Ολομέλεια για την, ε, με, σχετικά με τη Λευκή Βίβλο άνοιξε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και η συζήτηση αυτή θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του έτους. Το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα και εγώ θα ήθελα και οι πόλεις αλλά και οι περιφέρειες, κυρίως όμως οι πόλεις, να κάνουν διαλόγους, town halls όπως λέγονται, για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώστε τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και συζητήσουμε όλοι μαζί ποια είναι η κατεύθυνση που, θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή, που θέλουμε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που ξεκινήσαμε σήμερα αυτή τη ε, συζήτηση μέσω της δικής σας ολομέλειας. Σας ευχαριστώ. Thank you, thank you, thank you. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά ήδη σε διάφορες πόλεις, σε δήμους και σε κοινότητες προσπαθούμε να διεξάγουμε τους διαλόγους αυτούς πολιτικούς στους οποίους αναφερθήκατε. Ορισμένοι έπρεπε να αποχωρήσουν από τους ομιλητές μας. Ο Γιώ Λάνιν επίσης πρέπει να αποχωρήσει, αλλά σίγουρα εμείς θα διεξάγουμε μια συζήτηση και μπορούμε έπειτα να υποβάλουμε και μια έκθεση για τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θέλουμε να καλύψουμε. Μπορούμε να αφιερώσουμε ακόμα περίπου μισή ώρα στο ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, στις 6 ώρα με την αντιπροσωπεία που έρχεται από το Ζάλαν. Θέλουμε, θέλω ακριβώς να θίξω το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περίμενα ότι θα συζητούσαμε από τις 5 μέχρι τις 6 μόνο. Έχω κάποιες ενηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να αποχωρήσω. Πρόεδρος, μπορούμε να ακούσουμε τώρα σύντομες παρεμβάσεις. Ο κύριος Σνάιντερ πρώτος για τρία λεπτά. Πρόεδρε, αυτό είναι, αυτή είναι η πιο παράδοξη και εντυπωσιακή συζήτηση που έχω ζήσει. Δεν ξέρω αν θα μιλάει ο καθένας μόνος του ή αν θα σταματήσουμε την ε, συζήτηση. Εσείς τι λέτε. Θα πρέπει να αποφασίσουν τα μέλη, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει ο προγραμματισμός μας μέχρι τις 6.30. Αλλά ούτως ή άλλως για το θέμα αυτό θα έχουμε μια συζήτηση και στην Ολομέλεια του Μαΐου με τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο Κατάινεν και άλλους προσκεκλημένους. Επομένως, θα καταγράψουμε τις, τις συμβολές σας στη συζήτηση. Ίσως θα ήταν καλό και οι πολιτικές ομάδες να καταγράψουν τα πολιτικά μηνύματα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Δεν χρειάζεται να συζητούμε μεταξύ μας εδώ. Ο κύριος Σνάιντερ, προτείνω να μην κάνουμε τώρα συζήτηση, αλλά το Μάιο τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο χθε στο Προεδρείο αυτό το πράγμα είπαμε και να συζητήσουμε και για τη δική μας τη γνωμοδότηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Γιατί είναι μια ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να δεξαχθεί για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τοποθέτηση Επιτροπής των Περιφερειών. Πρόεδρος, ας ακούσουμε και άλλους επικεφαλείς πολιτικών ομάδων γιατί τους άλλους προβλεπόντουσαν κάποιες σύντομες παρεμβάσεις από εσά. Πείτε μου απλώς αν θέλετε να κάνουμε τώρα τη συζήτηση ή αν προτιμάτε να μετατεθεί τον ε, Μάιο. Συμφωνείτε, Σόμερς, συμφωνώ με τα σοφά λόγια του κυρίου Σνάιντερ. Για μία φορά μίλησε πάρα πολύ σοφά, αυτή τη φορά τουλάχιστον. Κατίους Καμαρίνη, παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι ε, για όλους μας είναι κάπως δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον να γίνει αυτό σε αντιπαράθεση μετά όσα είπαν οι ευρωβουλευτές. Θα μπορούσαμε όντως να, να μεταθέσουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά έστω σήμερα να καταλήξουμε σε μια πολιτική τοποθέτηση και όντως το Μάιο να κάνουμε μια πιο διεξοδική συζήτηση βάσει της Λευκής Βίβλου θα μπορούσαμε τουλάχιστον σήμερα, αν μη τι άλλο, να τοποθετηθούμε, μη τι άλλο, πολιτικά. Να υπάρχει, αν θέλετε, ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θα βγει έστω και από τη σημερινή συζήτηση. Άλλη παρακαλώ. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Σνάιντερ. Ίσως όντως είναι καλύτερα να μεταθέσουμε τη συζήτηση αυτή για κάποια άλλη συνεδρίαση. Ας ακούσουμε μία ακόμα παρέμβαση. Έχουμε έναν φοιτητή από τον Μάστριχτ Ας ακούσουμε και τη δική του την άποψη. Τι έχετε να μας πείτε, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να ταινίσουμε μέσω των φοιτητών αυτών και εμείς το μέλλον. Ναι, ευχαριστώ. Ονομάζομαι τα Βέβη. Είμαι φοιτήτρια της πολιτικής ιστορίας και φιλοσοφίας από το Μάστριχτ μαζί με άλλους συμφοιτητές Χαρακτηρίσαμε πέρσι την απόφαση για το Brexit ως το σημείο στο οποίο δεν μπορεί πια να μένει μέτοχη στις εξελίξεις η δική μας γενιά. Μια θετική πρωτοβουλία λοιπόν ως αντιπρόταση για όλους τους ευρωσκεπτικιστές, όλους τους ευρωαπεσιόδοξους. Ένα πρόγραμμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο συμμετέχουν πια πάρα πολλές χώρες, φοιτητές από πολλές χώρες, με μηδενική χρηματοδότηση. Τι θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να συζητήσουμε και συγκινησιακά και με πλαισίωση τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να, να δημιουργήσουμε αυτή την συζήτηση. Πάντα υπέρ, ποτέ κατά. Προσπαθούμε να συζητούμε το γιατί η Ευρώπη, why Europe. Σε αυτή την ερώτηση θέλουμε να δίνουμε τις απαντήσεις μας. Έχουμε 150.000 εντωμεταξύ ε, ανθρώπους που μας ακολουθούν κάθε εβδομάδα και 350.000 στο Twitter. Η πρώτα στο Facebook, δεύτερη στο Twitter. Έτσι λοιπόν έχουμε μια βάση διαλόγου. Ακούμε κάθε άποψη. Με βάση το δεδομένο ότι δεν μπορεί να είναι λύση η επιστροφή στα εθνικά κράτη. Δεν θέλουμε που δεν είναι να προαγάγουμε την τωρινή εκδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τη μεταρρυθμίσουμε. Αλλά μόνο μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι οι επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων λοιπόν συμφωνούν να μεταθέσουμε τη συζήτηση αυτή για το ζήτημα μάλλον αυτό στην Ολομέλεια του Μαΐου. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε τώρα με την γνωμοδότηση που δεν μπορέσαμε να καλύψουμε πριν από δύο ώρες και να περάσουμε και στις υπόλοιπες γνωμοδοτήσεις στη συνέχεια. Ο κύριος Βαλκάρας Σίσο θα έρθει επίσης στις 6.30 για να μιλήσουμε για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Κύριε Ρουγιών, εσείς πάρα πολύ σύντομα. Δύο ακόμα παρεμβάσεις μετά και ολοκληρώνουμε πάντως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω μια συζήτηση. Θα ήθελα απλώς ήδη από τώρα να αρχίσουμε να προωθούμε την ιδέα του Effective Europe, της αποτελεσματικής Ευρώπης και να αρχίσουμε τελικά να διορτόμαστε λίγο περισσότερο για το ποια είναι η άποψη των δικών μας των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Ξέρετε ότι ε, και στη Γαλλία και στην Ιταλία έχει γίνει μια συζήτηση γύρω από το Reflecting Europe. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να συλλέξουμε τις ε, απόψεις των πολιτών, να μπορέσουν οι πολίτες να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια αυτά. Θέλουμε να έχουμε 12.000 τέτοιες συμβολές από τους πολίτες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη συνεδρία Σολομέλης να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούμε σαν ήμασταν μια ομάδα πίεση. Θέλουμε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλε αυτέ τι απόψει στα πλαίσια μια πραγματική δημοκρατική συνέλευση, προκειμένου να μπορέσουν οι απόψει των πολιτών να φτάσουν και σε εμά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σύντομο αυτό μελλοντικό χρονικό διάστημα. Θα ήθελα λοιπόν ήδη από τώρα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του Reflecting Europa. Σα ευχαριστούμε, κύριο Μανλόβ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορούμε να διεξάγουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή για το μέλλον της Ευρώπης. Ακριβώς επειδή το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, παρουσίασε πρόσφατα τη Λευκή Βίβλο και είχαμε και τρεις ομιλητές σήμερα και δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό μαζί τους σήμερα, στη σημερινή Ελομέλεια. Χάσαμε μια ευκαιρία και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και στο παρελθόν τις προηγούμενες δύο ε, συνόδους ολομελίες είχαμε αν θέλετε, ανάλογες εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα χάσμα που διευρύνει τώρα και περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συζήτηση αυτή να λαμβάνει χώρα όταν είναι επίκαιρη. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, επαόριστον να αναβάλουμε τη συζήτηση αυτή, ούτε καν και αν πρόκειται ουσιαστικά για δύο μήνες. Μακάρθη παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ακούω ότι λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε. Ωστόσο, η πολιτική της συνοχής είναι μια ξεχωριστή ιδέα, ένα ξεχωριστό στοιχείο. Όλοι μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε τα ερωτικά ταμεία, αλλά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά, δημόσια, σαν να το ξεχνάμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διάσταση στο Reflecting Europe θα έχουμε τόσε χιλιάδες σχέδια, τόσους χιλιάδες αποδέκτες και συμφωνώ με όσο είπε ο κύριο Ρόλινγκ ότι θα πρέπει να προβλέψουμε ακόμη ένα στάδιο για την επικοινωνιακή μας πολιτική, να μην περιμένουμε μέχρι τον Μάιο δεν εννοώ ότι παραγωνίζουμε την ε, διαρθρωτική πολιτική, την πολιτική της συνοχής ε, στην επικοινωνιακή μας, ε, επικοινωνιακές μας πολιτικές, αλλά τουλάχιστον αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να σας θυμίσω ότι ούτως ή άλλως τώρα πρέπει να δούμε το σημείο 6 για, τα συστήματα υγείας, γιατί στις 6.30 θα δούμε το σημείο 9, όπου έχουμε την ε, γνωμοδότηση για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης με καλεσμένο τον κύριο Βαλκάρσελ Σίσο. Οπότε ας είμαστε λίγο ευέλικτοι και μια που και οι πέντε πρόεδροι συμφωνούν, θα επικεντρωθούμε στην ε, γενική συζήτηση ε, και θα έχουμε τον απαραίτητο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ενδελεχή κουβέντα. Μόνο έτσι μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προβλέψει για σήμερα και για αύριο βέβαια. Οπότε συμφωνούμε, Συζητούμε, ε, ε, κλείνουμε τη συζήτηση αυτή τώρα και θα δούμε την, το θέμα αυτό και του Reflecting Europe και την Λευκή Βίβλο στην ε, ολομέλειά μας. Έχουμε ένα σύντομο βιντεάκι και μετά θα δώσουμε το λόγο στη Μπιργκίτα Σακρεντέους. Να δούμε το βίντεο όμως πρώτα. Ωραία. Οπότε πάμε πίσω στο σημείο 6 για την ολοκλήρωση συνεργασία και επιδόσεις των συστημάτων υγείας. Έχουμε την κυρία Μπιγκίτα Σακρεντέους μαζί μας. Θα της δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της. και βεβαίως έχουμε πολλές τροπολογίες. Θα τις συζητήσουμε και μετά θα δούμε και την ψηφοφορία. Βιργίτα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να κάνει μια γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας, ε, αλλά ο ε, Επίτροπος Αντριουκάητης και οι Υπουργοί Υγείας θεωρούν επίσης καλή ιδέα να γίνει μια τέτοια ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλία. Η Κομισιόν, από ό,τι φαίνεται, θα μελετήσει το θέμα τη υγεία μέσα στην επόμενη διετία για, τα, για το πώ λειτουργεί αυτή στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουν ήδη κάνει κάποια βήματα, έχει υπάρξει έκθεση για, το, για τα συστήματα υγεία, η οποία υιοθετήθηκε στο τέλο τη προηγούμενη χρονιά. Και βεβαίω υπάρχουν διάφορε προκλήσει, τι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η πρόνοια και, τα συστήματα υγείας, όπως είπε ο Επίτροπος, εμπίπτει απολύτως στις ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών. Οπότε η πρόνοια, ε, η παροχή ε, περίθαλψης δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά η υγεία παρόλα αυτά είναι ένας κλάδος που πρέπει να μελετήσουμε και εμείς και κυρίως επειδή αντιμετωπίζει τόσες πολλές προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να τις αντιμετωπίσουμε και σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο ε, κυρίως εκεί προκύπτουν οι προκλήσει αυτέ και εκεί πρέπει να παρέμβουμε για να τι αντιμετωπίσουμε. Είναι ουσιώδες να υπάρχει παροχή υγεία ανάλογα με τι ανάγκε του πληθυσμού. Βεβαίως πολλές φορές υπάρχει υπερκατανάλωση υπηρεσιών. Αλλά βεβαίως πάντα πρέπει να υπάρχει παροχή ε, ε, υπηρεσιών υγεία. Αν δούμε ωστόσο την οικονομία, οι χρόνιες παθήσεις είναι αυτές που οδήγησαν σε, οικονομικούς, σε λυπείς οικονομικούς πόρους για την τομέα της υγείας. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις χρόνιες παθήσεις. Επίσης πρέπει να φτάσουμε στην πρόνοια μέχρι το πρωτογενές επίπεδο. Αλλά ε, ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε και προληπτικά μέτρα. Σήμερα μιλούμε για την σημασία των τροφίμων για την υγεία μας και πολύ προληπτική εργασία έχει γίνει ως προς αυτό, αλλά πρέπει σε αυτό να βελτιωθούμε στις χώρες μας. Κυρίω όταν μιλούμε για την παροχή υπηρεσιών υγεία ε, προ του ηλικιωμένου. Πρέπει να δούμε πώ θα φροντίσουμε του ηλικιωμένου μα. Πρέπει σαφώ να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων που έχουν να κάνουν με τον τομέα τη υγεία. Και επίση πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς να έχουν έλεγχο όλων αυτών των υπηρεσιών. Βεβαίως ε, πρέπει και εμείς να έχουμε μια εντύπωση ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και βεβαίως η παροχή και η πρόνοια για τους ασθενείς είναι πολύ σημαντική. Μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε επαρκές προσωπικό στον τομέα της υγείας όποιος δουλεύει στον κλάδο της υγείας ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να αρχίσουν να εξειδικεύονται σε επαγγέλματα του κλάδου της υγείας. Στην γνωμοδότηση αυτή, επίσης, τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα Εράσμους, όπου τα επαγγέλματα υγείας και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν ανταλλαγές και να μάθουν οι μεν από τους δε. Υπάρχει βεβαίως ε, ελπίδα μέσω και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν και εκεί σημαντικές εξελίξεις για τον τομέα της υγείας. Μπορεί ας πούμε, να υπάρχει μια ε, εφαρμογή. Πολλοί μπορούν να λάβουν υπηρεσίες υγείας μέσω μιας ε, εφαρμογής κυρίως ε, εμείς που ζούμε σε αεροκατοικημένες περιοχές, ε, μπορούμε, να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, η αντιμικροβιακή αντίσταση είναι πολύ σημαντικό και η Κομισιόν δουλεύει πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Φυσικά, καλωσορίζουμε στη γνωμοδότηση αυτή το ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός δικτύου για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία κυρίως σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Πρέπει να δούμε την παροχή ε, θεραπείων, πρέπει να δούμε τι δουλεύει και τι όχι και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο από κοινού. Πάμε τώρα στις τροπολογίες. Τρεις τροπολογίες είναι αυτές που θα ήθελα εγώ να αναφέρω. Μία η τροπολογία 3. Μιλούμε για την ε, μετανάστευση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα πνευματικής υγείας. Ε, έχω μιλήσει γενικόλογα εδώ για, τις, ε, για την πνευματική υγεία, την ψυχική υγεία, ψυχικές παθήσεις, για να μην κατονομάσω πολύ συγκεκριμένες ομάδες. θέλω να παραμείνει γενικόλογη η ε, αναφορά στο σημείο αυτό. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία. Στο, στην τροπολογία 6, αν η περίθαλψη θέλουμε να λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ του ιατρού ή του ιατρικού προσωπικού και του ασθενή. Ο ασθενής πολύ συχνά θέλει να επιλέξει ποιο θα του παράσχει την ε, περίθαλψη. Υπάρχουν ε, γιατροί ή ε, νοσηλευτικό προσωπικό που εμπιστεύονται καλύτερα. Δεν μπορώ όμω να δεχτώ την προσθήκη που θέλετε να γίνει μέσω τη τροπολογίας 6 στο σημείο 21. Και επίση για την τροπολογία 7, και εδώ δεν μπορώ να τη δεχτώ, γιατί δεν ισχύει ότι είναι τα δημόσια συστήματα υγείας αυτά που χρηματοδοτούν τον τομέα της υγείας. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν ε, κάποιες ε, επιλογές μέσω ασφαλιστικών εταιριών και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πλήρως τον τομέα της υγείας από το δημόσιο κορβανά, κάποια, άλλα, κάποια κρατημέλη έχουν διαφορετικές επιλογές. Γι' αυτό ε, δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία 7. Οπότε θα κλείσω εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον εμπειρογνώμονά μου, τον Έρικ, ο οποίος ήταν πραγματικά ιδιαιτέρως χρήσιμος στην σύνταξη της νομοδότησης και όλο το προσωπικό είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Θέλει να πάρει κάποιος το λόγο ή μπορούμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Λοιπόν, πάμε στις τροπολογίες τότε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ψηφίστε. Ευχαριστώ κατά. Ουδή. εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία υπαριθμών 2. Αν εγκριθεί μάλλον πρόκειται για τροπολογία της εισηγήτριας, αν εγκριθεί, τότε οι δύο καταπίπτει. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει δύο λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 3. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οι περισσότεροι είστε υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 4. Αν εγκριθεί εδώ πέρα η τροπολογία της ηγήτριας, τότε καταπίπτει η αρχική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ για την τροπολογία της ηγήτριας. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται λοιπόν, καταπίπτει 4. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 5 της ηγήτριας. Αν εγκριθεί, καταπίπτει η αρχική τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία παριθμών 6. Κύριε Πέτισεν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στη Δανία κάνουμε δεκάδες έρευνες ικανοποίησης είναι συντριπτικά τα ποσότητα των ικανοποιημένων πολιτών. Εκείνοι που δηλώνουν μη ικανοποιημένοι επισημαίνουν την απουσία ενημέρωσης ως λόγο των δυσχεριών. Και αυτό ακριβώς προσπαθώ να ε, επισημάνω με την τροπολογία ότι ο ασθενής ζητά περισσότερες πληροφορίες, όσο το δυνατόν περισσότερες πριν μπει ε, στο νοσοκομείο, πριν νοσηλευτεί. Απάντηση η Θα ήθελα να σας επισημάνω, κύριε συνάδελφε, ότι εδώ μιλάτε είτε για εξωτερική είτε για εσωτερική νοσηλεία ή αγωγή. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε πριν από την εισαγωγή του ασθενούς, γιατί δεν εισάγονται όλοι οι ασθενείς στο νοσοκομείο. Επομένως, η πρόταση σας δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές συνθήκες. Κύριο Γκόρ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ιδίω πρόβλημα με την διατύπωση εδώ, γιατί η κατάσταση του Ηνωμένου Βασίλειου είναι αντίστοιχη με αυτή της Δανίας. Μπορεί κανείς να καταφύγει σε ένα ιστότοπο και να επιλέξει όχι μόνο το νοσοκομείο του, αλλά και τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό. Αυτό προβλέπεται ήδη στο σύστημά μας. Επομένως είναι ελλειπής η διατύπωση εδώ γιατί δεν καταγράφει την κατάσταση όπως αυτή ισχύει σε ορισμένα τουλάχιστον κρατημέλη. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τροπολογία 6. Ναι ή όχι, η συγκέντρια επενθυμίζω είναι κατά. So that I can see what is. Oh, yes, for sure. Yeah. Okay. Okay, we can uh, close the vote. Καλώς, κύριε το της, της ε, ψηφοφορίας. Απορρίπτεται από την πλειοψηφία. Τροπολογία 7. Η συγγετρία είναι κατά υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Η συγγετρία κατά. Κύριε Πέτερσεν. εδώ. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε μια πρόταση τύπου Florence Nightingale. δηλαδή μπορούμε να θεραπευτούμε αν πιστεύουμε σε αυτό. Ναι, μπορούμε να διοχετεύσουμε προς νέους, αλλά δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Και γι' αυτό ζητούμε τη διαγραφή του σχετικού εδαφείου. Το να, ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερους εργαζόμενους νέους, να προσλάβουμε περισσότερους νέους. Αυτό δεν ε, γίνεται με ευχολόγια, δεν αρκούν τα ευχολόγια, η Συνομίλησα με το δίκτυο και ρώτησα τι πρέπει να κάνουμε Σε σχέση με αυτήν την ε, μαζική μετατόπιση νοσηλευτικού προσωπικού από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης προς τις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Δεν είναι ένδειξη αλληλεγγύης η κατάσταση που έχουμε. Πρέπει να μπορεί να παραμείνει κανείς στο δομέα του και στη χώρα του και γι' αυτό έχω κάνει τη σχετική έρευνα σε συνεργασία με το δίκτυο και από την Επιτροπή ενημερώνομαι ότι αυτή η προσήλωση, για αυτή η δέσμευση για ένα ευρωπαϊκό σώμα ε, αλληλεγγύης μπορεί να επιτρέψει την εκδήλωση αλληλεγγύης και αυτό ξέρουμε ότι δεν έχει ε, αναπτυχθεί επαρκώς στο χώρο της ε, υγείας γιατί υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε χώρες Αφρικής αλλά ε, δεν έχουμε αντίστοιχη δράση σε χώρε τη Ευρώπη. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ελληνική. Και πιστεύουμε ότι και στο χώρο τη υγεία πολλοί είναι οι νέοι οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι της, ε, των υπηρεσιών υγείας που θα μπορούσαν να αποτελούν ε, και, αποτελεί και πηγή έμπνευση για τους νέους, όπως άλλωστε και άλλοι τομείς. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για πρόταση τη Επιτροπής. Καλώς, λέει ο Πρόεδρο. ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν, η συγκεντρία είναι κατά υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, η συγκεκριά είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Η παριθμόν 10 της εισηγητρίας και αν εγκριθεί καταπίπτει η αρχική 10. Υπέρ της τροπολογίας εισηγητρίας λοιπόν. Κατά. Εγκρίνεται και καταπίπτει η αρχική 10. Τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε κατόπιν της ψηφοφορίας. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. μία, μία ψήφος κατά αποχές. Όχι και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην συγκεντρία. Okay, we are ready to... Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Θα γίνει μια συζήτηση γι' αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρώην Προεδρό μας και νυν Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ραμόν Λουίς Βαλκαρθέλ Σίζο. Uh, και βέβαια να καλέσω και τον εισηγητή μας, τον Μικέλ Ιρουχό, να έρθει και αυτός εδώ στο Προεδρείο. Okay, uh, Πολύ ωραία. Περιμένοντας να έρθει και ο συγητής μας, σας πω κάποια εισαγωγικά λόγια Κάτι το οποίο συνδέεται ουσιαστικά με αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Ξέρετε ότι έχουμε ένα βραβείο κάθε δύο χρόνια όσον αφορά τις πρωτεύουσε της καινοτομία. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει αύριο. Ο Επίτροπος Μένας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει όθηση στην πρωτοβουλία αυτή αλλά βέβαια καθότι συμβάλλουν οι πόλεις μας, οι περιφέρειές μας και οι δήμοι μας, μας ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας ενημερώνω σήμερα και επίσημη διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αύριο. Θα μπορώ να σας πω και ποια είναι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται, αλλά προτιμώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας ενημερώσει επισήμως αύριο και στην επιστολή προς τα μέλη την οποία θα σας αποστείλω θα σας μιλήσω περισσότερο για το διαγωνισμό αυτό όσον αφορά τις πρωτεύουσες καινοτομίας. Στο παρελθόν η διαδικασία αυτή ε, είχε αναδείξει το Άμστερνταμ πριν τη Βαρκελόνη παλαιότερα και θέλουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η τρίτη κατά σειρά πρωτεύουσα καινοτομία. Σας το λέω λοιπόν ήδη από σήμερα. Η επίσημη δικασία θα ξεκινήσει αύριο και είχαμε ξεκινήσει βέβαια άλλο διαδικασία όπως ξέρετε και πέρυσι. Είχαμε καταλήξει τότε σε τρεις νικητές που είχαν λάβει και αυτοί ένα βραβείο. Ουσιαστικά ήταν ένα χρηματικό έπαθλο για τα καινοτόμα αυτά αποτελέσματα τα οποία είχαν πετύχει και για το ότι είχαν δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας για τις νέες αυτές καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες λειτουργούν θετικά για τους Δήμους και τις πόλεις. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να ενημερώσετε και εσείς για το διαγωνισμό αυτό, για τη δικασία αυτή τους Δήμους και τις κοινότητές σας και τις πόλεις σας. Ας αφήσουμε όμως πρώτα τον εισηγητή μας να μας μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα, να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του και χαίρομαι πάρα πολύ, όπως σας είπα, που έχουμε τον Ραμόν Λουίς Βαλκαρέθα Σίζο μαζί μας, ο οποίος ήταν συντάκτης γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε να περάσουμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό και μέσω της δικής μας γνωμοδότησης να φωτίσουμε, θέλετε, τη διάσταση ή την πτυχή της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να προκύψουν και να ωφελήσουν το σύνολο της Ευρώπης. Από κοινού, λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες βάσει των νέων αυτών πλατφορμών στρατηγικών έξυπνη εξειδίκευση. Να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μα. Μικέλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω βασικά. Χαίρομαι που είμαι εδώ ως εκπρόσωπο τη Ναβάρα και μπορώ να μιλήσω την ε, γλώσσα μου, τη βασική. Θα μιλήσω λοιπόν για τις στρατηγικές ευφύους εξειδίκευσης που έχουμε αναπτύξει στο θέμα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια στρατηγική που πρέπει να είναι πάντοτε αηφόρος. Στόχοι είναι η επασχόληση, οι γλώσσες, οι κοινωνικές πτυχές, η ενέργεια κτλ. αυτές οι στρατηγικές εφίους εξιδικεύσεις πρέπει να ορίσουν και ένα μοντέλο, ένα πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις οικονομικές ε, και άλλες σχέσεις. Και βέβαια μιλούμε για πολύ σημαντικά εκτίματα για τις ε, περιφέρειες από την εξειδίκευση αυτή. Ένα θετικό αντίκτυπο δηλαδή στην ανάπτυξη των περιφερειών αυτών. και βέβαια και σε σχέση με την διεύρυνση των ε, οικονομικών πόρων που είναι περιορισμένοι προς το παρόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στάδιο και ο στόχος είναι ο στόχος της ε, κινητοποίησης και εξασφάλισης πόρων αλλά και ενίσχυσης της συνεργασίας σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο. Βεβαίως πρέπει να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε όθηση και στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία μέσω προγραμμάτων συνεργασίας. Με το τρίπτυχο αυτό. Έχουμε μία προϋπόθεση, έναν όρο εξάντε, γιατί πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, και όπως είπα, αυτός είναι να ενισχυθούν, να ενθαρρυνθούν οι αλλαγές προς την έξυπνη εξειδίκευση, πάντα με σεβασμό στην διαφορά και στην ποικιλία. Υπήρχαν, υπάρχουν δύο είδη κρατών στην Ευρώπη, όπως υπόθηκε νωρίτερα, τα μικρά κράτη και αυτά που δεν καταλαβαίνουν ακόμη ότι είναι μικρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και από την ε, έποψη της ε, μετά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είχε υποθεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η ενέργεια, η ε, καινοτομία και εμείς στην Αβάρα προχωρήσαμε ως πρωτοπόροι για την περιοχή μας και μπορέσαμε να αναπτύξουμε δοκιμές και εργαστήρια του τύπου αυτού. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία ε, επένδυση σε εργαστήρια του τύπου αυτού που δεν έχουν ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε και η Κίνα. Βεβαίως κάθε κράτος πρέπει να μπορεί να διαφυλάσει την ελευθερία επιλογών. Ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με επιλογές που γίνονται χωρίς ε, διάλογο ή χωρίς μια προηγούμενη στρατηγική. Άρα χρειάζεται μια συνεργασία για ε, να βελτιωθεί το αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών επιλογών και μετά πρέπει να περάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο που είναι η συνεργασία με τις περιφέρειες για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων, αλυσίδων πραγματικών σε περιφερειακό επίπεδο για την ανταλλαγή και ερευνητών, αλλά και γνώσεων ως προς τις υποδομές, ε, επιχειρήσεις κτλ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα βελτίωνε την αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ένας από τους ιδρυτές της Ευρώπης είχε πει ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα κατασκευαστεί σταδιακά. Και εμείς πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε με την έκθεση αυτή, με την ομοδότηση αυτή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί δεν υπάρχουν ούτε περιφέρειες, ούτε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνα τους μπορούν να επιτύχουν αυτή την αριστεία αν δεν συνεργάζονται με τα άλλα. Η έννοια λοιπόν της συνεργατικής σχέσης στην καινοτομία και ε, αποτρέπει την ε, ε, χρήση διπλών πόρων και προσπαθειών, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και ε, κοινή προσπάθεια όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια των κρατών και των περιφερειών. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βαλκάρθελ Σίσο στα Ισπανικά. Διαφορετική εκδοχή των Ισπανικών αυτή τη φορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, αξιότιμη κύριε Μαρκούλα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Λάμπερτς, κυρίες και κύριοι, κύριε Ρούχο, κύριε Σίγητα για την γνωμοδότηση αυτή. Αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε, είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι και πάλι εδώ μαζί σας στην Επιτροπή των Περιφερειών Ήμουνα περίπου για δύο δεκαετίες μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, ήμουνα πρόεδρος πριν γίνω ευρωβουλευτή. Νιώθω λοιπόν σαν στο σπίτι μου όταν είμαι εδώ μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, όντως ε, η Ευρώπη περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση Το 2017 ορτάζουμε την επέτειο των 60 ετών υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αγώνας για την δημοκρατία συνεχίζεται, η αύξηση των λαϊκιστικών κινημάτων. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας. Πρέπει να τους φέρουμε πιο κοντά στα θεσμικά μας όργανα. Γι' αυτό εσείς και το, τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο είσαστε παίχτες κλειδιά σε αυτή τη διαδικασία. Με τη βοήθεια βεβαίως των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχουν ε, ξεκινήσει και εκτελέσει πολλά ευρωπαϊκά project, δείχνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τους πολίτες της να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και βεβαίως θέλω να επαναλάβω και εγώ τη δική μου στήριξη και τη δέσμευσή μου στην Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ είμαι εδώ όχι μόνο ως μέλος της ε, Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπεύθυνο για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπής των Περιφερειών. Συζητούμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα το απόγευμα. Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό. Τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει μια νέα πρωτοβουλία για τις στρατηγική αυτή. Θα μα ανακοινώσουν τι πρόκειται να κάνουν. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τι απόψει του τοπικού και του περιφερειακού επίπεδου υπόψη τη. Οι στρατηγικέ έξυπνη ε, εξειδίκευση αποτελούν ένα κοινό εγχείρημα όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει θέσει εργασία που, δίνουν ευκαιρίες στις ε, περιφέρειες να εξυγχρονιστούν, να μετατραπούν σε πιο καινοτόμους κόμβους σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο. Η ε, γνωμοδότηση αυτή που προετοίμασε ο κύριος Ιρούχο παραθέτει τα βασικά ζητήματα που βεβαίως μας απασχολούν όλους. Υπάρχουν στρατηγικέ ε, που πρέπει να παραμείνουν σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν πρέπει κατά κανέναν τρόπο να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό. Επίση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει διακυβέρνηση πολυεπίπεδη και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλη αυτή τη διαδικασία χάραξη αυτών των στρατηγικών. Επίση, πρέπει συνεχώ να αναθεωρούμε αυτέ τι στρατηγικέ και να ενισχύσουμε την συμμετοχική διαδικασία να την επιταχύνουμε και πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη και την, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι σημαντικό πρέπει να προχωρήσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα υπάρξουν καλώς λειτουργούσες και αποτελεσματικές στρατηγικές. Έχουμε κάποια αποτελέσματα ήδη, μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο εφαρμογή των στρατηγικών που οδήγησαν στα καλά αποτελέσματα αυτά και επίση η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ενίσχυση των συνεργειών, την συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και τη διεύρυνση των διαφόρων κλάστερ, των διαφόρων κόμβων που υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορούν οι περιφέρειες να ανταλλάσσουν ευέλικτε πρακτικές και να ενισχύουν τα project που έχουν ξεκινήσει και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προσπάθειες που κάνουν έτσι ώστε και η οικονομία να είναι πιο ανταγωνιστική και να έχουμε και πιο ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας. Τέλος, θέλω να πω ότι να τονίσω την σύσταση του εισηγητού για την ενδιάμεση αναθεώρηση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Κυρίως σε ό,τι αφορά τον, την όλη διαδικασία ελέγχου και αναθεώρησης. Γίνονται διάφορες παραπομπές, διάφορες αναφορές στην ε, χρηματοδότηση, το ορίζοντος 2020 και το σχέδιο Juncker που ούτως ή άλλω είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και τα οποία θα μελετήσουμε την επόμενη περίοδο. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, το σχέδιο αυτογνωμοδότησης έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου βελτιώνουμε τι στρατηγικέ μα, Έχουμε το πολιετές ε, πρόγραμμα ε, μέχρι το 2020, από το 2014 στο 2020. Έχουμε τις πολιτικές συνοχής. Έχουμε το ε, RIS3 και έχουμε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, την οποία εγώ συνέταξα ως συγητής, έτσι μας βοηθούν όλα τα στοιχεία αυτά για τις στρατηγικές ε, ε, εξειδικεύσεις, πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να τις καταστήσουμε αποτελεσματικές και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν αντίκτυπο. Η γνωμοδότηση αυτή προωθεί την βελτίωση των πραγμάτων έτσι ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία. Και βεβαίως αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες. Όταν το Κοινοβούλιο συνέταξε την έκθεσή του, είχα την ε, ευκαιρία να έχω μια πολύ καλή διαβούλευση με τις περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ήταν καθήλυνα αρμόδιε για τι στρατηγικές αυτέ, και βεβαίω θέλω να ευχαριστήσω όλου για τη συμμετοχή του, και οι ιδέες τους πρέπει να πω ότι ελήφθησαν υπόψη, συμπεριλήφθησαν στην έκθεση και εγκρίθηκε η έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, επαναλαμβάνω την δέσμευσή μου για την αποτελεσματική ε, εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή και για την εφαρμογή βεβαίω του RIS 3. Και επίσης πολύ σύντομα να πω ότι η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και τα σωστά πραγματικά αυτά αποτελέσματα θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συζήτησης για την μελλοντική περιφερειακή πολιτική. Πάντα δουλεύουμε με βάση την αλληλεγγύη. Την πίστη μας στην ελληνική, η οποία βρίσκεται πραγματικά στον πυρήνα των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση του τουλεχθέντος γνωρίζω πολύ καλά τις διάφορες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει να να γίνονται σε απάντηση της ε, συζήτησης που κάνει η Κομισιόν για το RIS 3 και βεβαίως εγώ θα συνεχίσω να παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Θα δω τι θα προκύψει από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της διάσκεψης στο Ελσίνκι που θα γίνει τον Ιούνιο. Με βάση λοιπόν όλες αυτές τις δραστηριότητες θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τη δουλειά που γίνεται και τα στοιχεία που υπάρχουν και βεβαίως αυτό θα ενισχυθεί και από την συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την ενίσχυση των πολιτικών συνοχής και την ε, αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης είναι πολύ σημαντικές για όλες τις περιφέρειες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παρεμβάσεις από τα μέλη. Ο κύριο Μακάρθη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι πολύ σημαντική και συνδέει πάρα πολλά από τα στοιχεία της ατζέντα για την κοινοτομία, τα οποία μελετάμε τα δύο τελευταία χρόνια. Έρθε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή η γνωμοδότηση αυτή και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες νομοθετικές γύρω από τα δίκτυα έξυπνης εξειδίκευσης. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των ε, συστημάτων αυτών προκειμένου να καταφέρουν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Ακριβώ όπω έχουμε και τι πρωτο... πρωτεύουσε καινοτομίε, θα πρέπει να καταφέρουμε να δούμε ποιε είναι οι νέε αυτέ πλατφόρμε, οι οποίε υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κλάστερ και κόμβι στου οποίου αναφερθήκατε, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερα, περισσότερο τι στρατηγικέ έξυπνη εξειδίκευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω της, των δικτύων αυτών να ε, έχουμε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους άρχισε να, δει, να βλέπει λίγο τις ανάγκες χρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καλύτερη ευφύης ανάλυση, αν θέλετε, των πραγματικών αναγκών των δικτύων αυτών. Και να συγχαρώ και τον συντάκτη της γνωμοδότησης, γιατί πραγματικά η γνωμοδότηση αυτή είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε να κάνω μία πρόταση αυτή τη στιγμή προς τον Ευρωβουλευτή που μαζί μας, τον Ραμόν Λουίσα. Ένα από τα σημαντικά πράγματα που κάνετε στα πλαίσια του ε, Κοινοβουλίου και στα πλαίσια των υπηρεσιών έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με το ζήτημα αυτό της εφιούς εξειδίκευσης, όπου προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες εκείνες οι οποίες έχουν τα ίδια θεματικά ενδιαφέροντα να συνεργαστούν και να συμβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο στην οικονομική μεταρρύθμιση και στην οικονομική ανάπτυξή του, στον οικονομικό μετασχηματισμό του, αν θέλετε. Νομίζω λοιπόν ότι η εργασία που επιτελείται από τις, ε, ευρωπαϊκ... από τις υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική και συμβάλλει πραγματικά στην καλύτερη λειτουργία των δικτύων αυτών έξυπνη εξειδίκευση. Θα ήθελα λοιπόν να το θίξω αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσετε περισσότερο και την εργασία λοιπόν αυτή που κάνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που συνάδει πάρα πολύ με τις προτάσεις που κάνει και ο δικός μας ο συντάκτης γνωμοδότησης στη δική του την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πάρουμε τις βασικές ιδέες τις οποίες ε, εκπονείτε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταφέρουμε να τις υλοποιήσουμε στην πράξη. Η εργασία μας δεν πρέπει να σταματά όταν εγκρίνεται μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια γνωμοδότηση στη δική μας την Επιτροπή, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι ιδέες αυτές να εφαρμόζονται, να ελομπιούνται στην πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα επικοδομητική συνεργασία και προστιθέμενη ευρωπαϊκή ε, αξία μέσω τη συνεργασία αυτή που έχουμε ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών. Δεν ξέρω αν ο εισηγητή θέλει αυτή τη στιγμή να ξαναπάρει το λόγο μετά τι παρατηρήσει αυτέ ή μάλλον πρώτα α ακούσουμε μια παρατήρηση ακόμα. Εσύ έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρέμβασή του, με την οποία συμφωνώ γενικώ. Έχω μια σειρά τροπολογιών, τις οποίες έχω αποστείλει, οι οποίες σχετίζονται ε, με ένα σημείο όπου έχω διαφορετική άποψη από τον εισηγητή, ότι οι στρατηγικές έξυπνες εξειδίκευσης μας έχουν βοηθήσει να προωθήσουμε πολλά project, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά ακριβώς τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα στον κανονισμό τα οποία αρκούν. Οι επιπλέον υποχρεώσεις των περιφερειών για την, ε, για την περισσότερη ευελιξία στις στρατηγικές τους νομίζω ότι θα περιορίσουν τις δυνατότητες παρέμβασης των περιφερειών. Ούτω ή άλλω η στρατηγική αυτή είναι στρατηγική που βρίσκεται στην ε, ευχέρεια των εθνικών αλλά και των περιφερειακών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τι ε, ε, καταστάσει που υπάρχουν, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι μα και θα πρέπει να εκπονήσουμε τους, τον τρόπο για να του επιτύχουμε. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο περαιτέρω λοιπόν υποχρεώσει και ρυθμίσει για τι περιφέρειε νομίζω ότι θα είναι αντιπαραγωγικέ. Γιατί οι περιφέρειε θα πρέπει να έχουν την ελευθερία και την ευελιξία να εκπονήσουν τι δικέ του στρατηγικέ και αυτό, αν περάσει, θα τι περιορίσει. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι με το να πιέσουμε την Κομισιόν να περιορίσει ακόμη περισσότερο τι δραστηριότητε των περιφερειών. Κάποιες από τις τροπολογίες έχουν γίνει δεκτές από τον ε, εισηγητή, αλλά κάποιες ε, αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης ε, σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων αυτή και από, τον, από την οποία προέρχομαι εγώ. Οι στρατηγικέ τη έξυπνη εξειδίκευση ναι είναι σημαντικέ, αλλά θέλουμε να έχουμε και την ελευθερία ώστε οι περιφέρειες να μπορούν να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν πώ θα δομηθούν αυτέ οι στρατηγικέ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Σιγητά, μια σύντομη απάντηση για όσα ακούσατε και μετά να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι η γνωμοδότηση αυτή, όπως το είπε και ο συνάδελφος Βαρκάθελ Σίσο, έρχεται μια επίκαιρη στιγμή δύο μέρες προτού ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο μήνες προτού υποβληθεί η πρώτη ανακοίνωση σχετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως Επιτροπή λοιπόν των Περιφερειών ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε, θα καταφέρουμε να είμαστε παρόντες στη συνδιάσκεψη του Ελσίνκη τον Ιούνιο. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της γνωμοδότησης αυτής, ήρθα σε επαφή και διαβούλευση με πάρα πολλές περιφέρειες και εδώ στις Βρυξέλλες και με τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας εδώ. Και ήρθα σε επαφή βέβαια και με πάρα πολλούς ανθρώπους που εκπροσωπούν πολλές διαφορετικές περιφέρειες και είδα ότι η κατάσταση διαφέρει πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να αποκρισταλώσω στη γνωμοδότηση αυτή και ουδέποτε αναφέρομαι σε ρύθμιση ή σε κανονισμό ενδεχομένως να εμφανίζεται σε κάποιες τροπολογίες. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν προσπαθώ να περιορίσω την ευελιξία των περιφερειών. Αντιθέτως, διατηρείται αυτή η ευελιξία μέσω της γνωμοδότησής μου. Αυτό το οποίο ζητώ είναι στα πλαίσια των στρατηγικών έξυπνης εξειδικευσής RIS3 να μπορεί να συμβάλλει περισσότερο το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες και ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές περιφέρειες οι οποίες έχουν ζητήσει υποστήριξη, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το κεντρικό δηλαδή επίπεδο, προκειμένου να καταφέρουν να εφαρμόσουν τις στρατηγικές αυτές έξυπνης εξειδίκευση. Αυτό ζητάμε στη γνωμοδότηση αυτή, αυτή την έκκληση κάνουμε. Θέλουμε μία αποσαφήνιση των κανόνων, διότι το 2013 Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η εξάντε προϋπόθεση ρεσιμότητα πλέον όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία. Ουσιαστικά πολλές περιφέρειες οι οποίες προσπαθούν να ανταχθούν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης δεν έχουν τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες ή τους απαραίτητους πόρου και γι' αυτό το λόγο ζητούν υποστήριξη αλλά και διευκρινήσεις από το κεντρικό επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Θέλουν να γνωρίζουν ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να εφαρμόσουν σωστά τις στρατηγικές αυτές έξυπνες ε, εξειδίκευσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις στρατηγικές έξυπνες εξειδίκευσης, τα RIS3, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις ε, περιφερειακές ε, αξιακές αλυσίδες ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε την ευελιξία ή το περιθώριο ελιγμού, αν θέλετε, κάθε περιφέρειας. Αντίθετα, προσπαθούμε μέσω περισσότερων διευκρινήσεων να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε περιφέρεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορεί να εφαρμόσει στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον ε, Ραμόν Λουίς Βαλκαρέφ για την παρουσία του εδώ. Και μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Και μετά θα ζητήσω από τον Καλχάινς να προεδρεύσει. Περνάμε στην τροπολογία παριθμών 1. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 2, γλωσσική τροποποίηση εδώ, μόνο για την ελληνική εκδοχή. Καλύπτεται λοιπόν από τεχνικής πλευράς υπεριθμών 4 τροπολογία υπέρ ο υπέρ παρακαλώ. Συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος. Τροπολογία υπεριθμών 3. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οι περισσότεροι είναι υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία υπεριθμών 4. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ουδή εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία περιθμών 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οι περισσότεροι είστε υπέρ, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία παριθμών 6, τροπολογία του εισηγητή. Αν εγκριθεί τότε αρχική 6 καταπίπτει υπέρ για την τροπολογία του εισηγητή παρακαλώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται λοιπόν Καταπίπτει η αρχική τροπολογία 6, τροπολογία παριθμών 7 του εισηγητή. Αν εγκριθεί οι αρχικέ 7 και 8 καταπίπτουν, ε, υπέρ παρακαλώ για τι τροπολογίε του εισηγητή κατά. Οι περισσότερε υπέρ εγκρίνονται. Περνάμε στην... Ε, οι 7 και 8 καταπίπτουν οι αρχικέ, δηλαδή τροπολογία 9. Ο εισηγητή είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία αριθμών 10 του εισηγητή που καλύπτει τις 10, 11, 12, 13, 14 υπέρ παρακαλώ για τις τροπολογίες του εισηγητή κατά ουδείς εγκρίνονται οι 10, 11, 12, 13 και 14 αρχικές καταπίπτουν τροπολογία υπαριθμών 15 ο εισηγητής είναι κατά υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 16. Ο συγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 και 18 ταυτόσιμες. Τις ψηφίσουμε από κοινού. Είναι κατά ο συγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οι περισσότεροι είστε κατά. Απορρίπτονται λοιπόν τροπολογία υπαριθμών 19, ο συγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπάρχει μια προφορική συμβαστική τροπολογία για τις 20, 21 και 23. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ναι. Επιτρέψτε να παρέμβω γιατί υπάρχει μια προφορική συμβαστική της τελευταίας στιγμής. Τη βλέπετε στην οθόνη. Είναι εντάξει μεν, αλλά θα εξαφανιστεί η λέξη regulatory, ρυθμιστικός. Και το ensure γίνεται encourage. Αντί για εξασφαλίζει, ενθαρρύνει. Εξαφανίζεται, διαγράφεται το regulatory. Ο πρόεδρος υπέρ παρακαλώ με τη συμβαστική κατά ουδής εγκρίνεται οι 20-21-23 καταπίπτουν άλλη προφορική για την 23 και 4 και ο συγκητής την έχετε στην οθόνη αν δέχεστε να την ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ Ευχαριστώ κατά. Εγκρίνεται η προφορική, συμβαστική τροπολογία και καταπίπτουν οι αντίστοιχε. 25. Πάλι προφορική συμβαστική, καταπίπτουν τότε 25, 26 και 27 αν την εγκρίνεται. Την έχετε στην οθόνη σας, παρακαλώ, υπέρ, κατά, κανείς, εγκρίνεται, πίπτων 25, 26, 27, η 30 του εισηγητή, η 28R, η 30 για την 28R, καταπίπτει επομένως 28R, υπέρ παρακαλώ, κατά. Κανείς εγκρίνεται, 29 συγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Ουδής εγκρίνεται, Συνεχίζουμε πέρα κατά εγκρίνεται 31 και πάλι είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά. Ο Λίγη, αλλά η πλειοψηφία είναι υπέρ, 32. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ψηφίστε παρακαλώ, ευχαριστώ, κατά. Εγκρίνεται 33 τότε θα καταπέσει 34 υπέρ της 33 κατά απερίφθη 34 υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνεται η 35R Εάν εγκριθεί καταπίπτουν 35 και 36. Ε, παρακαλώ ψηφίστε. Ευχαριστώ κατά. Ουδής εγκρίνεται. 37 ο εισηγητής είναι υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 38 ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 39 και 40 προφορική τροπολογία την έχετε στην οθόνη σας του εισηγητή. Υπέρ της προφορικής συμβαστικής κατά ουδής εγκρίνεται 41 ο εισηγητής είναι κατά υπέρ παρακαλώ κατά απερίφθη 42. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Εγκρίνεται. 43. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 άρτου εισηγητή Εάν εγκριθεί 44, 45, 46, 48 καταπίπτουν, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και, κατα... και καταπίπτουν οι τροπολογίες και τη 48. Ο εισηγητής. 49. Θέλετε το λόγο. Πολύ σύντομα και πάλι στη βασική γλώσσα. Θέλω μόνο να επισημάνω μια πτυχή. Εδώ μιλούμε για μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σύσταση και αναφερόμαστε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το αίτημα. Συμμετοχή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περαιτέρω παρακολούθηση της υπόθεσης με μια ομάδα εργασίας που θα συγκροτηθεί, στην οποία θα συμμετέχουν τα μέλη. Καλώς, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, παρακαλώ. κατά ουδής αποχές ουδεμία και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Uh, uh, Δύο ανακοινώσεις έχω. Υπάρχει καταρχάς φωτογράφος έξω από την αίθουσα για να μπορέσετε να βγάλετε νέες φωτογραφίες εφόσον το επιθυμείτε. Θα είναι εδώ μέχρι τις 9 ή τέλος πάντων μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας και στο τέλος της Ολομέλειας θα έχουμε την ε, δεξίωση της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας στο, κτίριο της Επιτροπής των ε, Περιφερειών. Οπότε μόλις τελειώσουμε από εδώ μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην α, δεξίωση. Θα δώσω την προεδρία τώρα στο Καρλ Χάινς. Υπάρχουν διάφορες α, ε, ε, δραστηριότητες, συναντήσεις για την ψηφιοποίηση, στις οποίες θα πρέπει να παρευρεθώ και διάφορες εκδηλώσεις και την Παρασκευή, όπως είπα, και βεβαίως θα συμμετάσχω εξ ονόματος όλων μας στην μεγάλη σύνοδο που θα γίνει και στις ε, δραστηριότητες του Σαββάτου. Οπότε ο Καρχάινς θα αναλάβει από εδώ και μπρος την Προεδρία. Να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να πάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερησία διάταξη για σήμερα. Ψήφισμα για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εν ώψη του προγράμματο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2018. Ποιος θέλει το λόγο. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Καλά ξεκινάμε. Οπότε πάμε κατευθείαν στις τροπολογίες. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άλμπερτ, έχεις το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Ο ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αυτή η τροπολογία εκ πρώτη όψη φαίνεται ότι θα μπορούσε να τύχει υποστήριξη, αλλά οι πυλώνε που αναφέρονται στο αρχικό σημείο ε, έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη βρίσκονται στην Ευρώπη 2020. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι κάποιες, ε, επιπλέον, κάποιοι επιπλέον όροι ε, ανθεκτικοί και ανταγωνιστικοί ως αποτέλεσμα του ότι αυτοί οι όροι υπάρχουν και στην Λευκή Βίβλο. Η Λευκή Βίβλος όμως είναι Λευκή Βίβλος προς το παρόν, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, οπότε θα ήθελα να παραμείνουμε στην φρασιολογία που υπάρχει στα έγγραφα που είναι ήδη εγκεκριμένα και τα οποία ήδη έχουμε υποστηρίξει. Άλλος κανείς που να θέλει το λόγο? Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι κατά? Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Α, συγγνώμη. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θέλω να ενθαρρύνω τους συναδέλφους, Πρόεδρε, να υποστηρίξουν την τροπολογία αυτή. Θέλουμε να επανεπιβεβαιώσουμε αρχές τις οποίες έχουμε εγκρίνει στο παρελθόν ως Επιτροπή των Περιφερειών. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιστάσεις όπου όντως έχουν υπάρξει ασύμετρα σοκ και στα οποία δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Οπότε δεν βλέπω τι ακριβώς είναι το απαράδεκτο στο να προσθέσουμε τις σχετικές, τους σχετικούς όρους στο τέλος του σημείου 4. Ε, ελπίζω να μπορούν οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν την τροπολογία. Άλλος κανείς που να θέλει το λόγο. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. να δούμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is clo closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 6. Υπέρ. Συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που συνέχεια παρεμβαίνω. Αλλά... Συνάδελφοι, έχουμε μία δήλωση σχετική ήδη στην γνωμοδότηση για το πολυετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και στην συνεδρίαση που κάναμε έχουμε υιοθετήσει μια διατύπωση η οποία βρίσκεται ακριβώς στην διατύπωση που θέλουμε να προσθεθεί στο σημείο 4. Οπότε ελπίζω να μπορείτε να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Άλμπερτ. Πρόεδρε. Έχουμε την Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν ε, εντός αυτής διάφορα σενάρια τα οποία μάλλον θα επηρεάσουν και την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή είναι και σημαντικός πυλώνας για την Επιτροπή των Περιφερειών και έχει υπάρξει σημαντικός πυλώνας για πολλά χρόνια. Ελπίζω λοιπόν να μπορούμε να δεχτούμε την προσθήκη αυτών των όρων που ε, δείχνουν ότι η ε, ε, Λευκή Βίβλος δεν περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν την πολιτική συνοχή. Δεν συμφωνούμε με την τροπολογία αυτή. Ήδη αποφασίσαμε το πρωί να συζητήσουμε το θέμα αυτό και τον Μάιο. Νομίζω ότι εκεί είναι το κατάλληλο βήμα. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Άλλος κανείς που να θέλει το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Περνάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 15 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 η οποία αν εγκριθεί οι 21 και 22 καταπίπτουν. Υπέρ της 20 παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 η οποία να εγκριθεί οδηγεί, μάλλον 25 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Η τροπολογία απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 26 όπου έχουμε προφορική συμβαστική τροπολογία, τη βλέπετε στις οθόνες σας. Αν γίνει αποδεκτή η συμβαστική αυτή τροπολογία, η τροπολογία 26 αρχική καταπίπτει. Προφανώς. Υπέρ λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Ψηφίσουμε πάλι ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρα. Η τροπολογία 30 απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Αν εγκριθεί η 34 καταπίπτει. Υπέρ παρακαλώ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 42 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 43 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση άρτη ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Α, συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρο. Έχετε το λόγο, Άλμπερτ. Τελευταία φορά παίρνω το λόγο, κύριε πρόεδρε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ad hoc ε, ορισμένες ε, καταστάσεις όπως για παράδειγμα εδώ πέρα ανθρωπιστική βοήθεια, παράνομη διακίνηση των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει προφανώς όλους αντίθετους. Το μόνο το οποίο λέμε εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο συνάδει με πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νομοθετικά μέτρα για τα ζητήματα αυτά. Ελπίζω λοιπόν ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να στηρίξουν αυτή την τροπολογία. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Υπέρ, λοιπόν, παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας και να πάμε στη δεξίωση. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9.